Να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Μίρεκ Τοπολάνεκ, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Σας καλωσορίζουμε θερμά, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τοπολάνεκ. Επίσης, θα ήθελα να ε, καλωσορίσω θερμά και τον κύριο Μπαρόζο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, Όλοι μας ε, γνωρίζουμε ότι η Προεδρία είναι μια ιδιαίτερη πρόκληση και γνωρίζω ότι ο Πρωθυπουργό κύριος ε, Τοπολάνεκ ε, και πνευματικά αλλά και συναισθηματικά το εκλαμβάνει την Προεδρία ως πρόκληση ε, διότι έχει ζήσει τα χρόνια του κομμουνισμού και τώρα ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα λειτουργεί πλέον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά τη Σλοβενία αυτή είναι η δεύτερη Προεδρία μιας χώρας η οποία προσεχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Και φαντάζομαι εξ όλων μπορώ να πω ότι η τσεχική Προεδρία ε, χέρι της αμέριστης υποστήριξής μας και επιθυμούμε όλοι διακαώς σε τόσο δύσκολες εποχές η Τσεχική Προεδρία να στεφθεί από επιτυχία. Μετά από αυτά θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Προεδρεύοντα, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Τοπολάνεκ να απευθύνετε το λόγο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για άλλη μια φορά σας καλωσορίζουμε θερμά στο χώρο αυτό. Vážené Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έρχομαι εδώ σήμερα μπροστά σας για πρώτη φορά υπό την ιδιότητά μου ως Προεδρεύων του, του Συμβουλίου. Η τσεχική δημοκρατία πήρε τη σκητάλη τη ηγεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Γαλλία. Πολύ συμβολικό αυτό. Η Γαλλία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο για τη γέννηση της, αναγέννηση της Τσεχοσλοβακίας. Από τα παλιά χρόνια. Και ο βασιλιάς Κάρλος της Γαλλίας ε, ίδρυσε και το Πανεπιστήμιο στην ε, Τσεχία, στην Πράγα και τη Σορβόνη στη Γαλλία. Ε, συνδεόμαστε με τη Γαλλία όσον αφορά τη φιλοσοφία που ακολουθούμε για τις παγκόσμιες καθολικές αξίες. Δύσκολο να ιδρύσουμε πανεπιστήμιο στην Πράγα που να συναγωνιστεί την Σορβόνη. Εξίσου δύσκολο είναι να ανταγωνιστούμε τη Γαλλική Προεδρία. Δεν ήταν τυχαίο το ότι επέλεξα το παράδειγμα αυτό του μεσαιωνικού μονάρχη που σας προανέφερα για να δείξω τι σχέσεις είχαμε με τη Γαλλία και με τις ευρωπαϊκές αξίες. Ο Κάρλος IV, τον οποίο προανέφερα, στην πολιτική του δεν μπορούσε να ακολουθεί μόνο εθνικές κατευθύνσεις, έπρεπε να αντικατοπτρίζει και την ποικιλομορφία του, της αυτοκατορίας του. Και ακολουθεί κάπως την ιστορία του Μεσαίων αυτή την ιστορία η Γαλλία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολουθούμε γενικά μια κοινή προσέγγιση το γενικό συμφέρον έναντι του συμφέροντος κάθε χώρας. Δεν θέλουμε να ανάψυχει τη γραφειοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ πιστεύω στην προαναφερθήσα Ευρώπη, στην Ευρώπη της ελευθερίας, του νόμου, των ιδεών, των κανόνων, των νόμων. Εκεί που ο νόμος είναι πάνω από το άτομο, δεν μετράει το μέγεθος μιας χώρας. Αυτό που μετράει είναι η εξυπηρέτηση ενός κοινού σκοπού, μιας κοινή ιδέας. Ο ρόλος της χώρας που κατέχει την Προεδρία δεν είναι να προωθεί στα δικά της συμφέροντα ούτε να παίρνει αποφάσεις για άλλους. Ο ρόλος της χώρας είναι να είναι η διαμεσολαβήτρια και να τροφοδοτεί τη συζήτηση. Σήμερα δεν στέχομαι εδώ σαν Πρωθυπουργό της Τσεχικής Δημοκρατίας αλλά ως Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και οι απόψεις που θα σας ε, παρουσιάσω το επόμενο εξάμεινο δεν θα είναι προσωπικές απόψεις ούτε τσεχικές θέσεις αλλά θα είναι οι θέσεις των 27 κρατών μελών όπως συμπεριλαμβάνονται σε συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και δεν θα μπορούσα να φανταστώ την παρουσία μου μπροστά σας διαφορετική. Ως ερετά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε ερωτήσεις επί παντό επιστητού και με τα να εξηγήσω τη τσεχική θέση. Αυτό δεν είναι το ουσιαστικό όμως. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ο χώρος ε, που εκπροσωπούνται τα εθνικά συμφέροντα. Υπάρχει περίπλοκος ε, τρόπος ελέγχων εκεί για τη διασφάλιση και την προστασία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Θέλουμε να, βρούμε, ε, να βρίσκουμε συμβιβασμούς, κοινό τόπο και αυτό είναι πάντα κάτι το οποίο θα υπερασπίζομαι εδώ. Οι Τσέχοι πάντα εξέφραζαν κάποια προβλήματα, μάλλον δημιουργούσαν την εικόνα ότι είμαστε οι γκρινιάριδες, ότι πρέπει να μας φοβούνται ότι διαμαρτυρόμαστε συνέχεια και βάζουμε πρώτα τη χώρα μας και μετά όλα τα άλλα. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή την ιδέα και αυτές τι επικρίσεις που ακούγονται. Όπως και με τον πρώτο μας πρόεδρο, τον κύριο Μάζαρεκ, εγώ πιστεύω ότι τα τσεχικά θέματα είναι ευρωπαϊκά θέματα. Πάντα κινούμεθα εντός του πανευρωπαϊκού πλαισίου πάνω σε κοινέ ευρωπαϊκέ αξίε και παρακολουθώ τι εξελίξει σε άλλε χώρε. Όπω έγραψε πριν από 100 χρόνια ο πρόεδρο Μάζαρεκ το τσεχικό, για το τσεχικό ζήτημα, η εθνική μα και η λογοτεχνική αναγεννησία, αναζωογόνηση έλαβε χώρα όπως και αναζωογονήσεις και ε, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός ε, αυτό, ε, αντιστοιχούσε στις γενικότερες ευρωπαϊκές εξελίξεις η αναζωογόνηση και η ανάσταση αν θέλετε της Τσεχίας. Και αυτό συμβαίνει και σήμερα. Η Ευρώπη ζητά ένα νέο πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο θα την κατοπτίζει παραδοσιακές ευρωπαϊκές αξίες και ε, θα κοιτάζει πάντα και προς τον 21ο αιώνα. Θα ακολουθούμε το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, δηλαδή ε, ένωση στην ε, διαφορά. Και όπως και στο 19ο αιώνα, έτσι και τώρα οι Τσέχοι μπαίνουν σε αυτή τη συζήτηση σαν ένα νέο κράτος μέλος, μικρό κράτος μέλος, αλλά θεωρούμε ότι ανήκουμε από παλιά στην ευρωπαϊκή οικογένεια και νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να το αποδείξουμε αυτό κατά το επόμενο εξάμεινο. Η Τσεχική Προεδρία ε, λαμβάνει χώρα ένα πολύ σημαντικό έτος, πέντε χρόνια πέρασαν φέτος, μετά το μεγαλύτερο κύμα της Ευρωπαϊκής Διευρύνσεως το 2004, που ήταν και το αποτέλεσμα της επιτυχούς διαδικασίας της επανενώσεως στην Ευρώπη και φέτος η Ευρώπη θα γιορτάσει τα 20 χρόνια μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος που επέτρεψε στις χώρες του πρώην, της πρώην Σοβιετικής Ένωσης να μπουν στο χώρο της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Επίσης το 2009 θα έχουν περάσει 30 χρόνια μετά από τις πρώτες άμεσες εκλογές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από το τρίγωνο των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εκείνο που πιστεύουμε ότι είναι η πηγή της ε, άμεσης πολιτικής νομιμότητας. Είναι ο μόνος άμεσα εκλεγμένος φορέας της Ευρωπαϊκής Ενώσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και επειδή ζητείται πάντα η μείωση του δημοκρατικού ελλείμματος, γι' αυτό αυξήθηκαν σταδιακά και εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλος, φέτος πέρασαν 60 χρόνια μετά από την είδηση του ΝΑΤΟ, που είναι και η πιο σημαντική διατλαντική συμμαχία εκδηλώνει τους διατλαντικούς δεσμούς στον τομέα της ασφάλειας και επιβεβαιώνει και την αξία που έχουν οι ευρωπαϊκοί προσανατολισμοί. Το 2009 δεν θα είναι μόνο οι σημαντικές αυτές επέτειοι που λαμβάνουν χώρα, αλλά θα αντιμετωπιστούν και σημαντικές προκλήσεις. Θα πρέπει να εξακολουθήσουμε τις προσπάθειες στην επίλυση θεσμικών θεμάτων. Ο διεθνής ρόλος Ευρωπαϊκής Ενώσεως δοκιμάζεται, διότι υπάρχουν ανεπίλητα προβλήματα, σύγκρουση στη Γεωργία, αλλά και νέα κλιμάκωση των γεγονότων στην Μέση Ανατολή. Και τέλος, το θέμα της ασφαλείας είναι καυτό ζήτημα για μία ακόμη φορά όπω ήταν και κατά τη διάρκεια τη Γαλλική Προεδρία. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα νέα αυτά γεγονότα και προβλήματα και δεν αποκλείονται και νέε εκπλήξει. Το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είναι κάτι που μπορεί να επηρεάσει η χώρα που έχει την Προεδρία. Μπορούμε να επιλέξουμε όμω την επιλογή των ε, προτεραιοτήτων. Και είμαι εδώ σήμερα για να σα παρουσιάσω αυτές τις προτεραιότητε. Πρωταρχικός μα στόχο ήταν να εξασφαλίσουμε το ότι αυτέ οι προτεραιότητε δεν αντικατοπτρίζουν μόνο τι τσεχικέ θέσει, αλλά αντικατοπτρίζουν και τι εξελίξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώ και τι θέσει και οι ιδέε ε, των άλλων κρατών μελών. Προσπαθήσαμε να πετυχαίνουμε πάντα συνένεση και δεν θέλουμε αντιπαραθέσεις. Παρόλο που δεν θα συμφωνούν όλοι βέβαια με όλε αυτέ τι προτεραιότητε που είναι δικέ μα, ελπίζω ότι ο καθένα από εσά θα βρει μεταξύ των προτεραιοτήτων κάτι με το οποίο συμφωνεί. Ταυτόχρονα, όπω για κάθε κράτο μέλο, έτσι και η τσεχική δημοκρατία, η Προεδρία αποτελεί ευκαιρία να επιστήσει την προσοχή σε τομεί όπου μπορούμε να παράσχουμε προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Ποιοι είναι αυτοί οι τομεί, σαν χώρα που εξαρτάται από την εισαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου και σαν χώρα που ανήκε στο Ανατολικό Μπλοκ καταλαβαίνουμε ποια είναι η έννοια του ασφαλούς ενεργειακού εφοδιασμού αλλά είναι προϋπόθεση και μόνο για οικονομική ευμάρεια αλλά και μια ελεύθερη και ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Σαν νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως με εμπειρία του ολοκληρωτισμού Εκτιμούμε το ότι μπορούμε να συμμετέχουμε σε αυτήν την κοινότητα και είναι ηθικό μας καθήκον να ενισχύσουμε την συνεργασία με εκείνους που παρέμειναν εκτός. Και όπως ε, και η Γαλλία χρησιμοποίησε τεχνογνωσία της στη Μεσόγειο, θέλουμε να τονίσουμε και εμείς πόσο σημαντική είναι η συνεργασία μας με τις ανατολικές χώρες. Άλλη συνεισφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εμπειρία που έχουμε με την τραπεζική κρίση που περάσαμε τη δεκαετία των 90. Χάρη στη σταθεροποίηση των, δικών μας τραπεζών είμαστε από τις λίγες χώρες σήμερα που δεν έπρεπε να ε, προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις τράπεζές μας στα πλαίσια της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι προτεραιότητές μας αντικατοπτρίζουν τη γνωσία τη τσεχική, την εμπειρία της Τσεχίας και σεβόμαστε βέβαια και τη συνέχεια των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως γνωρίζετε, σύνθημα της Προεδρίας μας είναι η Ευρώπη άνευ εμποδίων, ανεφραγμών, ανεφορίων. Υπότιτλος θα μπορούσε να είναι η Ευρώπη των κανόνων, υπότιτλος αυτού του συνθήματος. Αυτό το όραμα απαιτεί να δοθεί νέα σημασία ε, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Πιστεύουμε μόνο ότι η Ευρώπη που χρησιμοποιεί πλήρως το δυναμικό το οικονομικό και το ανθρώπινο και το πολιτιστικό μπορεί να σταθεί ε, στον πολιτικό και τον οικονομικό ανταγωνισμό. Κάτι που ισχύει έτσι περαιτέρω τώρα που περνάμε την κρίση και εμποδίζεται η πλήρη χρήση τη δυναμικότητα τη Ευρώπη από εσωτερικού φραγμού. Και εδώ μιλάω για τα τελευταία εμπόδια που υπάρχουν για την ολοκλήρωση των τεσσάρων βασικών ελευθεριών τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Μιλώ για τον διοικητικό φόρτο, για τις επιχειρήσεις και το γεγονός ότι δεν υπάρχει αλληλοσύνδεση των δικτύων ενεργείας. Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε μια Ευρώπη χωρίς κανόνες και σύνορα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τις παράνομες δραστηριότητες οι οποίες απειλούν την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός ο σαφής ορισμός των εμποδίων θα μας βοηθήσει να άρουμε τα εξωτερικά προσκόμματα όπως ισχύουν στο εξωτερικό εμπόριο και να λάβουμε υπόψη και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας. Η δημοκρατία της Τσεχίας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να ανταποκριθεί σε τρεις βασικούς ε, στόχους. οικονομία, ενέργεια και Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο. Πιστεύω ότι αυτά τα τρία ε θα ε, αφορούσαν στην ουσία μάλλον επικεντρώνεται στο φυσικό αέριο και στην Γάζα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες και νομίζω ότι το φυσικό αέριο και η Γάζα αποτελούν έναν ειδικό φόρτο για εμάς. Βεβαίως θα μπορούσα να μιλήσω και για μεμονωμένες προτεραιότητες, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ε, σήμερα βρισκόμαστε στην 14η Ιανουαρίου και καταφέραμε να επιλύσουμε το δυσχερές πρόβλημα με τη Ρωσία για την παροχή φυσικού αερίου για να ξανανοίξουν οι στρόφιγγες και επίσης προσπαθούμε να άρουμε τα προσκόμματα στο Μεσανατολικό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διανοιχθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι προς τη λωρίδα της Γάζας, κάτι το οποίο εν μέρη έχουμε επιτύχει. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Πιστεύω ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να τορπιλήσει τις προσπάθειές μας. Και νομίζω ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό, δηλαδή να μην το μετατρέψουμε σε ένα εσωτερικό πόλεμο που αφορά τα εσωτερικά της ε, Τσεχίας. Θα προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε τις δηλώσεις της διάσκεψης κορυφής των G20 καθώς και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μην έχουμε υπερρύθμιση και να αποφύγουμε τον προστατευτισμό. Δηλαδή θα πρέπει να βασιστούμε σε συγκεκριμένους κανόνες, δεν θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια πολιτική εσωστρέφειας, αλλά να ανοίξουμε τα, τα σύνορά μας προς τον ε, κόσμο. Όπως είπε και ο κύριος ε, Ντόλ, η παρούσα χρηματοπιστωτική κρίση δεν σημαίνει ότι έχει αποτύχει το σύστημα του καπιταλισμού. Απλώς ανασχηματίζεται. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν θέματα κεφαλαιακής επάρκειας και επίσης να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οδηγία για τις ε, πληρωμές ε, στην Ευρώπη, καθώς και να δούμε πώς θα εφαρμόσουμε τον οδικό χάρτη του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων και του Συμβουλίου Οικονομικών Υποθέσεων. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ πλήρως Πιστεύω ότι μία ε, οικονομική ευμάρεια στην Ευρώπη θα μπορέσει να διασφαλίσει και το εμπόριο και την ασφάλεια και το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης. Επίσης, τονίζουμε την εφαρμογή της στρατηγικής της Λισαβόνας μέσα στα πλαίσια μακρόπνων πολιτικών διαρθρώσεων. Ως προς την ΚΑΠ θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε το σύστημα άμεσων πληρωμών. Αυτό αφορά το ποσό, το ίδιο το ποσό ή το αντίτιμο πληρωμών, καθώς και το σύστημα πληρωμών. Θα θέλαμε να λάβουμε υπόψη το όλο ζήτημα για την μελλοντική συζήτηση που θα αφορά την ΚΑΠ μετά το 2013. Πιστεύω ότι οι ολέθριες συνέπειες της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης μας οδηγούν στο να ξανασκεφτούμε ζητήματα ανταγωνισμού και ιδιαίτερα τις ε, τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίας. Επίσης θα ήθελα να προσθέσω μια πέμπτη ελευθερία, την ελεύθερη κυκλοφορία της γνώσης, έτσι ώστε να καταπολεμήσουμε τον ε, σκοταδισμό. Θα πρέπει λοιπόν να μειώσουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και η τσεχική δημοκρατία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή. Ως προς το εξωτερικό εμπόριο θα προσπαθήσουμε να αναζωπυρώσουμε τις συζητήσεις του ΠΟΕ πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ε, τελειώσουμε με το γύρο της Ντόχα ως προς την, ατζέντα, την αναπτυξιακή ατζέντα και πιστεύουμε ότι η Προεδρία μας θα προωθήσει πολυμελείς συζητήσεις και συμφωνίες. Πολυμερείς συμφωνίες, με συγχωρείτε. Επίσης θα πρέπει να ασχοληθούμε με θέματα έρευνας και ανάπτυξης έτσι ώστε να άρουμε τον διοικητικό φόρτο. Ο Μάρτιν Σούλτς πολύ σωστά είχε πει ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να ανταγωνιστεί άλλες περιφέρειες του κόσμου ως προς το χαμηλά ημερομίστια αλλά ως προς την καινοτομία και την γνώση. καθώς και την τεχνογνωσία. Ενέργεια. Αυτή είναι η δεύτερη προτεραιότητά μας, η οποία εντάσσεται πολύ καλά στο παρόν ε, χρηματοοικονομικό πλαίσιο. Η παρούσα ε, κρίση ίσως ε, οδηγεί σε ευθύνουσα πορεία, την πορεία της Ευρώπης, αλλά νομίζω ότι μας οδηγεί σε μια αναδιάρθρωση πολιτικών οικονομίας και ασφάλειας και εμείς θα προσπαθήσουμε να προωθήσουμε την, ε, μια βιώσιμη πολιτική ενέργειας για την Ευρώπη. Επίσης, θα πρέπει να, να προωθήσουμε τη δεύτερη στρατηγική αναθεώρηση του τομέα της ενέργειας που αφορά την ε, προσφορά και τη ζήτηση ενέργειας. Θα προσπαθήσουμε να, να προωθήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα υποδομής και θα προσπαθήσουμε να έχουμε ελάχιστα αποθέματα αργού πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στο ορόσημο των 120 ημερών, δηλαδή να έχουμε επάρκεια για 120 ημέρες. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και τα ευρωπαϊκά ενεργειακά δίκτυα. Επίσης, να υπόψη μας και το νομοθετικό πακέτο το οποίο έκρινε η Κομισιόν για το 2008. Όσον αφορά τα νέα ενεργειακά δίκτυα τα οποία ε, θα συνδέουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι στο θέμα αυτό θα μπορούμε να υπολογίζουμε στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξάλλου, επιθυμούμε να αυξήσουμε τον αριθμό των προμηθευτών και να επεκτείνουμε τις ε, διαδρομές. Εδώ βέβαια εντάσσεται ο αγωγός Ναμπούκ Επιθυμούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος και να δώσουμε σημασία στις, ε, στις επενδύσεις για νέες τεχνολογίες. Όσον αφορά τώρα τις ε, επιτυχίες μας, αυτές που επιδιώκουμε, εδώ θέλω να αναφέρω ότι επιθυμούμε να εγκαταστήσουμε ένα μηχανισμό ελέγχου όσον αφορά τη μεταφορά αερίου από τη Ρωσία στην Ουκρανία. Στόχος είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ρωσική Ομοσπονδία και την Ουκρανία και μεγαλύτερη διαφάνεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών και καλύτερο ενεργειακό μείγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οφείλουμε να σκεφτούμε σοβαρά το πώς ε, θα μπορέσουμε να έχουμε και ασφαλή πυρηνική ενέργεια. Η σχετική υποδομή πρέπει να βελτιωθεί στην Πυρηνική Ένωση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνδέονται αποτελεσματικά μεταξύ τους και να μπορούμε και εμείς να επιδιώξουμε την ε, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει και εξυγχρονισμός των συστημάτων εφοδιασμού. Ε, μας ενδιαφέρει να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν στο δίκτυο. Όσον αφορά το νομοθετικό έργο σε αυτό τον τομέα, θα ήθελα να αναφερθώ στο τρίτο πακέτο για τον ενεργειακό τομέα, το οποίο επιθυμούμε και να ολοκληρώσουμε. Να επανεξεταστούν οι δύο οδηγίε και οι δύο κανονισμοί για, τον, για, τον, για την αγορά ηλεκτρικού ρεύματος. Στόχος είναι η αγορά ε, για ηλεκτρική ενέργεια και αέριο να ε, απελευθερωθεί. Ένας άλλος σημαντικός τομέας είναι η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Αυτός είναι ένας στόχος της δικής μας, της τσεχικής προεδρίας και τούτο σημαίνει ότι η Τσεχία η Σουηδία και η Γαλλία, η Τρόικα αυτή, θα αντιμετωπίσει το όλο θέμα της ενέργειας ε, κάτω από όλα τα πρίσματα. Για μας λοιπόν πρώτη προτεραιότητα είναι η ενέργεια η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική προστασία του κλίματος. Και εδώ θα θέλαμε να έχουμε μια αποδεκτή συμφωνία σχετικά με τις υποχρεώσεις μας μετά το 2012. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα πρέπει να συμμετάσχουν σε αυτό το παιχνίδι έτσι ώστε να ε, προετοιμάσουμε την διεθνή συνένεση που θα επιδιώξουμε το 2010 στην ε, Κοπενχάγη στις αρχές αυτού του έτους θυμηθήκαμε ότι πάντα μπορούν να ε, προκύψουν απρόβλεπτα γεγονότα. Αναφέρομαι στην κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στο Ισραήλ και, το, τη Χαμάς και αυτό απαιτεί τον ε, συντονισμό και με διεθνείς και με τοπικούς παράγοντες. Είναι αδύνατον να επιτευχθεί η ειρήνη εάν η Παλαιστίνη δεν αντιμετωπίζεται ως ένα κράτος το οποίο βέβαια εγγυάται την ασφάλεια των γειτόνων του. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οφείλει να συνεχίσει τις ε, προσπάθειές της, τη βοήθειά της για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους. Η Τσεχική Προεδρία τις καλές ε, στις σχέσεις με τους Παλαιστίνιους αλλά και με τους Ισραηλινούς θα τις εκμεταλλευτεί για να επιδιώξει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Αλλά αν δεν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι αδύνατο να υπάρξει και ε, ειρήνη διαρκείας. Εδώ θα ήθελα να σας επισημάνω πόσο ε, σημαντική είναι και η γεωργία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την περιοχή αυτή οφείλουμε να αναπτύξουμε μια στρατηγική και να επιδιώξουμε καλύτερη συνεργασία με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής, δηλαδή και με την Ουκρανία και με άλλες χώρες του Καυκάσου και της Κασπίας. Αυτό είναι σημαντικό και για καθαρά πρακτικούς λόγους. Όσον αφορά τώρα τις διατλαντικές σχέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρέπει να ε, επιδιώξει εξβελτίωση των σχέσεων με τι ΗΠΑ, γιατί αλλιώ δεν μπορεί να αναδειχθεί σε παγκόσμιο παίκτη. Τώρα όλο αυτό δεν μπορεί να τον αναλαμβάνουν μόνο οι ΗΠΑ, ε, ανήκει και σε εμά. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει σημασία σε ουσιαστικό διάλογο με του εκπροσώπου τη νέα Αμερικανική κυβέρνηση, κυρίω στου τομεί ε, ενέργεια, ε, κλίμα, σχέσει με Αφγανιστάν, Πακιστάν, Ρωσία και Μέση Ανατολή. Βεβαίως η θέση των κρατών ε, μελών ε, στην διαπραγμάτευση νέων συμφώνων με τη Ρωσία θα παίξει σημαντικό ρόλο. Τα τους τελευταίους μήνες ε, διαφάνηκε πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε κοινή ανάλυση, κοινή κατανόηση των θεμάτων της Ρωσίας. Άρα δηλαδή ε, χρειαζόμαστε τη συνεργασία με εμπειρογνώμονες από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Τσεχική Προεδρία επιθυμεί επίσης ε, να επιδιώξει τη διεύρυνση ε, στα Δυτικά Βαλκάνια που καλύπτει και την Τουρκία. εν ώψη της ε, χρηματοεπιστωτικής κρίσης και λόγω αυτής δεν πρέπει να ξεχνάμε τα προβλήματα στα Βαλκάνια. Η Κροατία απέδειξε ότι ε, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί οφείλουμε να τη στηρίξουμε σε αυτή την προσπάθεια. Η Τσεχική Προεδρία επιθυμεί να επιδιώξει ε, την βελτίωση της ε, πολιτικής γειτονίας και να βελτιώσουμε και τις σχέσεις ανάμεσα εταίρους. Εδώ αναφέρομαι στο Ισραήλ αλλά γενικότερα και στην διαδικασία ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Οι δραματικές εξελίξεις στην περιοχή αυτή δεν πρέπει να μας αποσπάσουν από τις προσπάθειές μας να ε, ενισχύσουμε περισσότερες περιοχές αυτές και να επιδιώξουμε την ειρήνη. Όλο και περισσότερο λοιπόν βλέπουμε να διαφαίνονται προβλήματα στον τομέα της ασφάλειας. Τα προβλήματα αυτά αφορούν όλους μας. Γι' αυτό λοιπόν οφείλουμε να επιδιώξουμε καλύτερη συνεργασία σε θέματα ποινικού, αστικού δικαίου. Γνωρίζουμε βέβαια πολύ καλά ότι οι ε, μεσούσεις της Προεδρίας μας ε, θα έχουμε τις ευρωεκλογέ. Ήδη πριν από το τέλος της ε, θητείας του Κοινοβουλίου πρέπει να ολοκληρωθούν αρκετές ε, νομοθετικές πράξεις. Αυτό που ενδιαφέρει επίση ε, είναι και το θέμα της ε, Ιρλανδίας, το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία, το ε, Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Θέλω λοιπόν να πω ότι αν γίνεται το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία η απάντηση ήταν αρνητική. Εμείς ε, χρειαζόμαστε μια λύση που να γίνει αποδεκτή από τους περισσότερους Ιρλανδούς. Αυτό θα βοηθήσει και στη δική μας την εσωτερική συζήτηση. Αλλά το θέμα της ε, Ιρλανδίας είναι και ευρωπαϊκό θέμα. Θεωρώ ότι Καμία άλλη χώρα δεν έχει αποδώσει σε θέματα ταυτότητας μεγαλύτερη σημασία από εμάς. Και αυτό μας ε, συνδέει με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, με την κατάσταση που βιώνει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αναζητά ένα νέο πρόσωπο, νέους στόχους και οράματα. Αυτό το γνωρίζουμε και εμείς από τη δική μας την ιστορία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε να σας προσφέρουμε εμπειρία 200 ετών αναζήτησης του ιστορικού μας ρόλου. Σκεπτόμενος λοιπόν τις σχέσεις ανάμεσα στην Ευρώπη και την Τσεχία, φτάνω στο να θυμάμαι αυτό το οποίο είπε πριν από 70 χρόνια ένας Τσέχος φιλόσοφος αν ισχυριζόμενος ότι η Τσέχη είναι η καρδιά της Ευρώπης, αυτό δεν το, δεν το εννοώ ε, γεωγραφικά, αλλά πνευματικά. Ε, εμείς είμαστε στο σταυροδρόμι της Ευρώπης όπου συγκεντρώνονται όλες οι κινήσεις και ε, οι πνευματικές εξελίξεις. Και το λέω αυτό Ακριβώς διότι έχουμε αυτή τη μοναδική θέση, άρα δηλαδή ο δικός μας ο στόχος είναι να παίξουμε το ρόλο του ε, διαπραγματευτή ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Πρόεδρος, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σας ευχαριστούμε θερμά για την ε, επικοδομητική και ε, περιεκτική εισήγησή σας και σας ευχόμεθα κάθε καλό. Τώρα δίνουμε το λόγο στον Πρόεδρο της Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κυρίε και κύριοι, οι πρώτε μέρε του 2009 δεν αφήνουν καμία αμφιβολία. Το επόμενο εξάμεινο θα θέσει σε δοκιμασία την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρώπη θα πρέπει να αποδείξει την αποφασιστικότητά τη, να βοηθήσει του ε, πολίτε, του εργαζομένου, τι επιχειρήσει, να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση. Θα πρέπει να αποδείξει την αλληλεγγύη της της περιπτώσεις ανάγκης όπως το απότομα σταμάτημα του φωδιασμού σε διακοπή σε φωδιασμό φυσικού αερίου που ζούμε θα πρέπει να δείξει τη δυνατότητα που έχει η Ευρώπη να επηρεάσει να ε, χρησιμοποιήσει την επιρροή της διευθέτηση των προβλημάτων που ε, εκπροσωπούν μια απειλή την στον κόσμο όπως το πρόβλημα στη Γάζα. Σε στενή συνεργασία με την Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου και θέλω να χαιρετήσω τον Πρωθυπουργό τον κ. Πολάνε και την ομάδα του και τους εύχομαι κάθε επιτυχία στην ηγεσία του Συμβουλίου και έχω πλήρη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της ε, τσεχικής δημοκρατίας να εκπληρώσει το σημαντικό της αυτό καθήκον. Σε στενή συνεργασία με τη τσεχική Προεδρία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θελήσει να αποδείξει ότι ανταποκρίνεται στο ύψο των περιστάσεων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μαζί μπορούμε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου να αποδείξουμε στου πολίτε γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τόσο απαραίτητη σήμερα να δείξουμε στους Ευρωπαίους γιατί έχουν άμεσο συμφέρον να εκφράζουν την άποψή τους εκλέγοντας τους βουλευτές ε, στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου. Να δείξουμε στους συμπολίτες μας γιατί η Ευρώπη χρειάζεται ε, βελτίωση στη δημοκρατία και στην αποτελεσματικότητα, κάτι που επιφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας και γιατί χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ τώρα. Που θέλουμε να κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Ξεκινάμε από στέρευα. Το 2008 η Ευρωπαϊκή Ένωση επέδειξε ότι μπορεί να πάρει δύσκολε αποφάσει που δεσμεύουν τι κοινωνίε μα για σειρά ετών. Το πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα αποδεικνύει πολύ καλά την πολιτική βούληση που επικρατεί στην Ευρώπη, που έχει οράματα και είναι αποφασισμένη. Αυτό το πακέτο μα επιτρέπει να προχωρήσουμε προ μια συμφωνία διεθνή φιλόδοξη το Δεκέμβριο του έτου. έτους. Το 2008 απέδειξε η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα που έχει να προσαρμόζεται στι αλλαγέ πολύ γρήγορα βρήκε τα μέσα να αντιδράσει στην κρίση του χρηματοδοτικού τομέα και πολύ γρήγορα συνεφώνησε επισχεδίου ανακάμψεως για να τονώσει την οικονομία χωρίς να περιμένει. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα. Το 2009 ε, προωθεί τη φήμη της στο προσκήνιο το διεθνές. Ήταν στην πρώτη γραμμή για να επιληθεί η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας και δεν φίδεται προσπαθειών για να πλησιάσουν οι δύο πλευρές στη Γάζα. Και χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον έχει ανοίξει, έχουν ανοίξει ανθρωπιστικοί διάδρομοι ούτω ώστε να βοηθηθεί ο Παλαιστινιακός λαός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης ενέπνευσε και τα θέματα που συζήτησαν οι G20 για να επιτεθούν κατά της οικονομικής κρίσεως και άνευ επιφυλάξεως υποστήριξε το άνοιγμα των αγορών κυρίως στα συμπεράσματα φαίνεται αυτό της διαδικασίας της Ντόχα για την ανάπτυξη και το εμπόριο και επίσης και ανταποκρίνεται στους στόχους της χιλιετίας. Η κρίση δεν θα πρέπει να υπονομεύσει στους στόχους της χιλιετίας. Η Ευρώπη θα πρέπει επίσης να συνεχίσει να κάνει τα πάντα για να ανταποκριθεί στις σημερινέ προκλήσεις και νομίζω ότι έχουμε κάθε λόγο να έχουμε εμπιστοσύνη στι ικανότητε Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει αυτό το χρόνο να κάνει τα πάντα, ούτω ώστε να μην χαθεί αυτή η ορμή που ξεκίνησε στην ε, Ουάσιγκτον κατά τη διάρκεια τη συνόδου των G20. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να συνεχίσουμε κάθε προσπάθεια για μια μεταρρύθμιση του χρηματοπιστικού συστήματος του παγκοσμίου και επίσης έχουμε στο Λονδίνο, στους G20, έχουμε ευκαιρία, θα πρέπει με μια φωνή εκεί να μιλήσει η Ευρώπη και να συνεχίσει να ηγείται στο θέμα τη μεταρρυθμίσεω του παγκοσμίου χρηματοστικού Συστήματος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίζει να προτείνει πρωτοβουλίε σημαντικέ φέτο, κυρίω για την καλύτερη ρύθμιση τη λειτουργία των χρηματοστικών αγορών, να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα δράση στον τομέα τη δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια και να προτείνει και μέτρα προσαρμογή στι αλλαγέ του κλίματο. Θα προετοιμάσουμε τι προτάσει μα ούτως ώστε να γίνει επανεξέταση το θέμα των δημοσιονομικών και θα προσέξουμε όλες ιδιαίτερες εξελίξεις τις οικονομικές και κοινωνικές και θα αναλάβουμε κάθε δέουσα πρωτοβουλία. Ε, πολύ σημαντικές προτάσεις εξετάζονται από εσά, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν χάρη στη δέσμευση της ψυχικής προεδρίας να υιοθετηθούν οι προτάσεις αυτές πριν από το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου όπως είναι η προτάση που αφορά την οικονομική χρηματοπιστωτική κρίση, το κοινωνικό πακέτο, η εσωτερική αγορά ενέργειας, που είναι κάτι πολύ επικαιρό και δείχνει πόσο είναι απαραίτητο κάτι τέτοια επικαιρότητα. Και το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και επίσης και για τις οδικές μεταφορές. Κυρίες και κύριοι, θα εστιάσω τα σχόλιά μας στο θέμα της ενέργειας και της οικονομίας. Οι πολίτες της Ευρώπης νιώθουν αυτή την πίεση φέτος. Και εδώ χρειάζεται αποτελεσματική δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται επίγοντα και αποτελεσματικά μέτρα στον τομέα του φυσικού αερίου, όπου έπρεπε να ασχοληθούμε ως προς αυτή την διαφορά μεταξύ Ουκρανίας-Ρωσίας για την διαμετακόμιση του φυσικού αερίου. Αυτό είναι κάτι το απαράδεκτο. Απαράδεκτο διότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές σε ορισμένα κράτη-μέλη βρίσκονται χωρίς φυσικό αέριο μία βδομάδα μετά από την διακοπή παροχής. Και όπως ξέρετε υπεγράφει συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας όπου αναφέρεται ότι θα εφαρμοστεί αυτό το πλαίσιο νέων, νέας παροχής. Και η Ρωσία και η Ουκρανία καταδεικνύουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις, ε, στις υποσχέσεις τους. Αυτό οδηγεί όμως σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις προς τους Ευρωπαίους καταναλωτές. Θα ήθελα να πω προς τη Μόσχα και το Κίεβο ότι αν δεν αρθούν στο ύψος των περιστάσεων θα ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αχθούν ενώπιον ε, του δικαστηρίου, του ΔΕΚ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε εναλλακτικές πηγές Εναλλακτικέ πηγές παροχής ενέργειας. Θα δούμε λοιπόν εντάχει κατά πόσο υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πολιτικές προθέσεις και βούληση για να ανταποκριθούν στη συμφωνία. Εάν δεν τηρήσουν τη συμφωνία τους, η Ρωσία και η Ουκρανία δεν είναι αξιόπιστοι εταίροι για την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την παροχή ενέργειας. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρώπη μετά από την αναθεώρηση του παρελθόντος Νοεμβρίου. Ως προς τα 5 δις ευρώ για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει να προωθηθούν και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Τσεχική Προεδρία διότι ε, δέχτηκε αυτές, αυτά τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μην αντιμετωπίσουμε τέτοιες ε, καταστάσεις στο μέλλον. Ως προς την οικονομία βλέπουμε ότι αυξάνεται η ανεργία και η παραγωγή ακολουθεί φθήνουσα πορεία. Δεν αποκρύπτουμε τη σοβαρότητα της κατάστασης, αλλά δεν θα πρέπει να είμαστε και ητοπαθείς. Έχουμε αναπτύξει τις σωστές στρατηγικές και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις πλέον ευάλωτες κατηγορίες. Μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις που θα μας οδηγήσουν στα κατάλληλα μέτρα αντιμετώπισης αυτής της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και το σχέδιο ανάκαμψης της Επιτροπής και του Συμβουλίου είναι η σωστή απάντηση που θα έχει αντίκτυπο σε κάθε κράτος μέλος. Γιατί το 1,5% του ΑΕΠ αποτελεί ένα ε, μεγάλο ποσό εάν δαπανηθεί βεβαίως σωστά και ανταποκρίνεται σε δύο στόχους, την μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και τις μεσοπρόθεσμες οικονομικές οθήσεις. Αυτή η κρίση αφορά τους Ευρωπαίους, την ευημερία τους, το βιωτικό τους επίπεδο και νομίζω ότι θα πρέπει να ανταποκριθούμε σωστά στην κρίση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, σωστή ευρωπαϊκή διάσταση του ζητήματος έτσι ώστε να υπάρχει θετικός αντίκτυπος σε όλα τα κράτη-μέλη μέσα στα πλαίσια αυτής της διάδρασης. Χρειάζεται βεβαίως η δέσμευση της Προεδρίας των κρατών μελών και του Κοινοβουλίου. Επίσης, θα πρέπει να προωθήσουμε τις ε, νομικές αποφάσεις μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αντιμετώπισης της Παγκοσμιοποίησης. Μιλάμε για 5 δις ευρώ μη ε, δαπανηθισών πιστώσεων υποχρεώσεων και οι ουκρανικές τιμές καταδεικνύουν ότι θα πρέπει να πληρώσουμε αυτά τα χάσματα τα οποία υπάρχουν. Η πραγματική εφαρμογή του σχεδίου αφορά 200 δις ευρώ που θα πρέπει να εισρεύσουν στις οικονομίες μας και θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μέσα στα πλαίσια αυτής της δράσης δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις μακρόπνοες πολιτικές. Θα πρέπει να στηριχθούμε στις ε, επιτυχίες μας, όπως την εσωτερική αγορά. Η Ευρώπη χωρίς σύνορα και χωρίς προσκόμματα είναι ένα πολύ καλό λογότυπο, το λογότυπο της ε, Τσεχικής Προεδρίας. Μια Ευρώπη χωρίς προσκόμματα χρειάζεται κανόνες έτσι ώστε να υπάρχει ίση πρόσβαση στην αγορά μεταξύ των οικονομικών φορέων. Κανόνες λοιπόν έτσι ώστε να είναι ε, σαφείς οι κανόνες για τους πολίτες. Οι κανόνες για να διασφαλίσουν μακροπρόθεσμα και ένα νέο τρόπο ζωής. Εμείς θα συνεργαστούμε στενά με την Προεδρία και με το Κοινοβούλιο προς αυτή την κατεύθυνση. Διότι η Ευρώπη την οποία επιθυμούμε είναι μια Ευρώπη που συνδυάζει την ελευθερία, την αλληλεγγύη και την ασφάλεια προς όφελος όλων των Ευρωπαίων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Και τώρα λοιπόν οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων, ο κύριος ε, Ιούζεφ Ντάουλ για πέντε λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά της, η Τσεχική Προεδρία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες και έχει το βαρύ καθήκον να διαχειριστεί τρεις σημαντικές κρίσεις συνεχίζεται η οικονομική και η κοινωνική κρίση. Η σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για το φυσικό αέριο που δημιουργεί προβλήματα στην Ευρώπη και στη γειτονική ε, περιοχή και η έκρηξη νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ενάντια αυτών των προκλήσεων η μόνη στάση για τις χώρες μας είναι να ενωθούν, να αποδείξουν ότι μπορούν να δείξουν αλληλεγγύη και να δράσουν συντονισμένα και αποφασιστικά. Και διαπιστώνω με θικανοποίησεως ότι η Τσεχική Δημοκρατία σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έδρασε ταχαία και ενωμένα στην ενεργειακή κρίση που θέτει σε αντιπαράθεση Μόσχα και Κίεβο. Παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί η λύση, δεν μπορούμε να δεχτούμε να είμαστε όμοιροι, θα πρέπει να δράσουμε με ενεργητικότητα. Και έχετε δίκιο κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ανάμεσα στις σημαντικές προτεραιότητες, προβλέποντας τον τομέα της ενέργειας, Τονίζοντας το αυτό, έδειξε με το δάχτυλο το σημαντική πρόκληση τα επόμενα χρόνια για την Ευρώπη. Η ενεργειακή μας ε, ανεξαρτησία απαιτεί και να έχουμε ποικιλόμορφη προμήθεια μορφών ενεργείας. Και το ΕΛΚ, όπως και οι Ευρωπαίοι πολίτες, ανησυχούμε πάρα πολύ από αυτή την αντιπαράθεση και από την απειλή που δημιουργεί για τις ευρωπαϊκές χώρες. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε τα κράτη-μέλη της Ενώσεως να είναι όμοιροι σε αυτή την αντιπαράθεση. Και για μία ακόμη φορά αυτό δείχνει την ανάγκη να συμφωνήσουμε κατεπηγόντως επί ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενέργεια. Θα πρέπει λοιπόν σοβαρά να προβληματιστούμε πώς θα μειώσουμε την εξάρτησή μας και να δράσουμε για τη δημιουργία του σωστού ενεργειακού μείγματος. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή μας δείχνει την ανάγκη που υπάρχει να επομιστούμε τις ευθύνες μας στο παγκόσμιο προσκήνιο. Ναι, η Ευρώπη είναι η πρώτη δωρήτρια ανθρωπιστικής βοήθειας στον κόσμο. Και μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό και θα πρέπει να συνεχίσουμε. Αλλά δεν είναι η ανθρωπιστική βοήθεια από μόνη της που θα επιλύσει τη σύγκρουση που θέτει σε αντιπαράθεση τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους. Αυτό που χρειάζεται είναι ισχυρή πολιτική βούληση στην Ευρώπη διαθρωμένη με τους απαραίτητους ανθρώπινους, στατιωτικούς και οικονομικούς πόρους, ούτως ώστε να είμαστε ένας φορές αξιόπιστος στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει τα μάτια καρφωμένα στον Μπαράκ Ομπάμα, διότι η Ευρώπη δεν ακόμα ικανή να προβάλλει τα οράματά της, τα ιδεώδη της και την τεχνογνωσία της. Η Ευρώπη επέκρινε και σωστά τη μονομερή προσέγγιση που ακολούθησε η παρούσα Αμερικανική κυβέρνηση. Και αν όπως το ελπίζω τα πράγματα αλλάξουν, με τον νέο ε, πρόεδρο της, τον ΙΠΑ, ε, θα μας επιτρέψει, θα πρέπει και εμείς να συμμετάσχουμε στην πολυμερή προσέγγιση, να χρησιμοποιήσουμε τη θετική ισχύ όχι για να κάνουμε πόλεμο, για να εξασφαλίσουμε την ειρήνη. Ας δώσουμε και οικονομικούς πόρους, ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε την πολιτική μας. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, σωστά τι εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κάνετε προτεραιότητα. Η επικαιρότητα μας δίνει πολλά παραδείγματα για το πόσο χρειάζεται αυτά τα θέματα να αντιμετωπίσουμε. Όπως η σχέση με τη Ρωσία, με τις σχέσεις με τη ΣΥΠΑ, τη Μέση Ανατολή. Και να μην αναφερθούμε στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο, την Αφρική και τι αναπτυσσόμενε χώρε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε περιμένουν από την Ευρώπη να παίξει το ρόλο τη στο διεθνέ προσκήνιο. Όλε οι δημοσκοπήσει το δείχνουν επί σειρά ετών. Γιατί να περιμένουμε Τέλος, η Προεδρία θα πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική και κοινωνική κρίση, φροντίζοντας να δημιουργηθούν και να εφαρμοστούν εθνικά σχέδια ανάκαμψης και στις G20 να κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση το μήνα Απρίλιο. Καλούμε την Τσεχική Δημοκρατία να συνεργαστεί στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τους ώστε να καθοριστούν και να εφαρμοστούν με τους διεθνείς εταίρους μας οι κανόνες που χρειάζονται να εφαρμοστούν για τους οικονομικούς φορείς. Θα πρέπει να προσπιστούμε το κοινωνικό μας μοντέλο, την κοινωνική οικονομία της αγοράς και να προωθήσουμε στην παγκόσμια χρηματοδοτική αγορά ένα σύστημα εποπτείας των αγορών ε, που είναι παρόμοιες με τις δικές μας, στη διαχείριση της οικονομικής κρίσεως και τη χρηματοστατική κρίση θα πρέπει να είναι ενωμένη η Ευρώπη και αποφασιστική. Βασιζόμαστε σε εσά, κύριε Τοπολάνεκ, στην Προεδρία σας για να δείξετε ε, πόσο πρόθυμοι είστε να λύσετε αυτά τα προβλήματα και να μας κατευθύνετε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρου ε, των Σοσιαλδημοκρατών, ο κύριος Μάρτιν Σούλτς επίσης για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τοπολάνεκ, κύριε Πρωθυπουργέ, εσείς ε, θα έχετε την τελευταία Προεδρία του Συμβουλίου ε, κατά αυτήν την θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό παλαιότερα ήταν ε, η Ολλανδική. Είχαμε τότε τον κύριο Μπαλκενέντε. Κανείς δεν θυμάται τι είχε πει εδώ τότε και τι του είχαμε απαντήσει. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται το εξής κρίσιμο ερώτημα. Αυτά τα οποία θα συζητήσουμε και θα επιτύχουμε τους επόμενους 5-6 μήνες αυτά θα είναι και η προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πολιτών στις ευρωεκλογέ. Αν δηλαδή οι πολίτες δουν ότι μεσούσεις της κρίσης το Κοινοβούλιο ή η Κομισιόν το Συμβούλιο κατόρθωσαν να ανταπεξέλθουν στην κρίση αυτή, τότε είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξει μια ε, θετική ατμόσφαιρα λίγο πριν από τις ευρωεκλογέ. Γι' αυτό λοιπόν εμείς ως σοσιαλδημοκράτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφερόμεθα ιδιαίτερα να επιτύχει η δική σας η Προεδρία στην αρχή της Προεδρίας, ε, τις πρώτες ημέρες, είχα κάποιες αμφιβολίες. Ο κύριος Σβάτσενμπερκ είπε ότι το Ισραήλ ε, καταφεύγει στο δικαίωμά του αυτοάμυνας ε, και με τον τρόπο αυτό ο κύριος Σβάτσενμπερκ τοποθετήθηκε μονομερός. Διορθώθηκε βέβαια, καλώς αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι αντικειμενική. Είπατε επίσης ότι στην διένεξη περί αερίου δεν θα παίξουμε το ρόλο του διαπραγματευτή. Το διορθώσατε και αυτό καλό και αυτό. Στην αρχή υπήρξαν δυσκολίες, αλλά τώρα φαίνεται να είσαστε ψύχρεμοι. Καλό και αυτό. Αυτά δηλαδή που ήταν οι αρχικές ε, δυσκολίες, αν αυτά, και εδώ έχει δίκιο ο κύριος ε, Μπαρόζο, οδήγησαν στο να είναι θετικές οι ενεργειές σας, τότε ε, και εσείς μπορείτε να υπολογίζετε στην υποστήριξη της πολιτικής μας ομάδας. Αυτά ισχύουν και για την ομιλία που κάνατε σήμερα το πρωί εδώ. Ε, μια ομιλία στην οποία εμείς είχαμε την ιδιαίτερα ευήκονους. Ε, λάβαμε ιδιαίτερα υπόψη μας ε, την ε, ομιλία σας. Θα αναφερθώ σε κάτι που είπατε. Παραθέσατε κάτι που είχε αναφέρει ο κύριος Ιούζεφ Ντάουλ ότι ε, όσον αφορά τη χρηματοπιστωτική κρίση δεν πρόκειται για ήττα του καπιταλισμού. Ναι, πράγματι δεν πρόκειται για ήττα του καπιταλισμού. Ο καπιταλισμός δυστυχώς εξακολουθεί να εφίσταται. Είναι όμως ήττα των καπιταλιστών, οι οποίοι χρόνια ολόκληρα μας έλεγαν ότι δεν χρειαζόμαστε κανόνες, η αγορά θα αυτορυθμιστεί μόνη της. Αυτοί λοιπόν υπέστησαν την ήττα και εάν εσείς ε, ο οποίος ε, μέχρι τώρα χαράσετε μια ε, πολιτική με βάση το ότι δεν χρειάζεται η αγορά κανόνες. Αν εσείς λοιπόν εδώ σήμερα το πρωί ε, λέτε ότι χρειαζόμαστε μια Ευρώπη των κανόνων, εγώ θα σας πω ναι, χρειαζόμαστε πράγματι κανόνες για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και με τα λόγια αυτά σας καλωσορίζουμε κύριε Τοπολάνεκ στο δικό μας το κλαμπ, στη δική μας την λέσχη εκείνων που επιθυμούν να υπάρχουν κανόνες. Από ό,τι φαίνεται το μάθατε το μάθημά σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη φάση της διεθνούς πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εάν θέλει να παίξει το ρόλο του παγκόσμιου παίκτη, κάτι το οποίο παρουσίασε ο πρόεδρος της Επιτροπής, κυρίως όσον αφορά θέματα ενέργειας. Αν θέλουμε να έχουμε πρωταρχικό ρόλο στην σύραξη της Γάζας, τότε η Ευρώπη δεν πρέπει να δεχθεί να κατατμηθεί σε μεμονωμένα τμήματα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τα 27 κράτη ως ένα ισχυρό πολιτικό και οικονομικό σύμπλεγμα. Γιατί μόνο αν αρνηθούμε αυτή τη διαίρεση, μόνο τότε θα είμαστε ισχυροί. Η δύναμη των άλλων έγκυται στο ότι θεωρούν οι Ευρωπαίοι ποτέ δεν θα είναι ενωμένοι. Ο Σβάτσεμπεκ λέει ε, το Ισραήλ αμήνεται, ο Λουί Μισελ λέει το Ισραήλ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και οι υπόλοιποι λένε «Ε, τι να την κάνουμε τώρα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν οι Ρούσοι και οι Ικρανοί πιστεύουν ότι μένουν από εδώ και οι άλλοι από εκεί, αυτό μας αποδυναμώνει. Ισχυροί είμαστε μόνο εφόσον έχουμε μια ισχυρή ε, συνταγματική βάση. Και τέτοια ισχυρή βάση είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη δική σας την κυβέρνηση, με τη δική σας την ε, Προεδρία και η δική σας κυβέρνηση παρεπιπτώσει, επιτρέψτε μου να πω, ήδη αρκετά τιμωρείτε με τον Πρόεδρο που σας έτυχε. Εάν λοιπόν εσείς ε, ε κατορθώσετε να κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας, αυτό θα είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για μια πολύ ισχυρή Ευρώπη. Τον κύριο Κλάους θα τον ακούσουμε το Φεβρουάριο. Θα έρθει στις Βρυξέλλες. Ε, στον πύργο της ε, Πράγας, ε, το είπατε κύριε πολάνεκ εκεί ήταν και ο Κάρολος ο Τέταρτος, ο οποίος κατασκεύασε το χρυσό δρόμο από την Πράγα στη Νιρεμβέργη. Την εποχή εκείνη ήταν ένα εκπληκτικό κατόρθωμα, ένα κατόρθωμα με στόχο να συνδέσει λαούς. Και ο Κάρλος ο Τέταρτος πριν γίνει Γερμανός αυτοκράτορας είχε έδρα στην Πράγα και ήταν δούκας του Λουξεμβούργου. Γι' αυτό λοιπόν οι εποχές αυτές ε, με τον πύργο της ε, Πράγας ήταν καθαρά ευρωπαϊκές και θέλουμε να ελπίζουμε ότι στον πύργο της Πράγας βρίσκεται σήμερα κάποιος ο οποίος είναι εξίσου Ευρωπαίος όπως ο Κάρολος ο Τέταρτος. Ε, για να δούμε τώρα οι φιλελεύθεροι. Περιμένουμε να δούμε με πολύ ενδιαφέρον τι είδους φιλικά αισθήματα αισθάνεται ο κ. Γότσον και για ποιον. Σας καλωσορίζω και εγώ εξ ονόματος της ομάδας μου, ένας μεγάλος ε, Τσέχος. Είχε πει πλέον ότι αναμένονται στόχοι από μένα και πρέπει να τους φτάσω. Αυτό ίσχυε για τον Μιλάν Μπάρος αλλά και για εσάς. Ως προς την οικονομία, είπατε ότι τα προσκόμματα στην αγορά πρέπει να αρθούν, εσωτερική και εξωτερική. Θα πρέπει να απαντήσουμε, να δώσουμε μία απάντηση στην ύφεση. Αυτό δεν σημαίνει μόνο δαπάνες, αλλά και καλύτερο ανταγωνισμό. Ε, απελευθέρωση της αγοράς και ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Βρισκόμαστε και διανύουμε πολύ δύσκολους ε, καιρούς. Πολλοί θα αμφισβητήσουν τη συνταγή σας, όχι όμως οι φιλελεύθεροι. Έχετε μεγάλη πείρα ως τσεχική δημοκρατία και βλέπουμε ότι η δύναμη της αγοράς είναι πολύ μεγάλη. Ως προς την ενέργεια έχετε απόλυτο δίκιο, ως προς την αναθεώρηση της στρατηγικής, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να αποτελέσει την οροφή των ε, φιλοδοξιών μας, αλλά εφαλτήριο για μεγαλύτερα βήματα. Έτσι ώστε από την ε, εξορυκτική βιομηχανία και ενέργεια να περάσουμε σε άλλες μορφές ενέργειας και να μην εξαρτώμεθα έτσι. Ε, ξέρουμε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν μπλοκάρει την κατάσταση. Οι Ρώσοι λένε ότι δεν μπορούν να δεχτούν αυτή τη συμφωνία διότι οι Ουκρανοί παραβιάζουν τους όρους της. Οι Ουκρανοί λένε ότι δεν έχουν φυσικό αέριο για να διαμετακομίσουν. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τους πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι αμφισβητούνται. Αλλά έτσι θα ξαναλειτουργήσουν γιατί καταλαβαίνετε ότι ζούμε ε, μέσα σε μια κατάσταση όπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ψύχος, τις ψυχρές νύχτες και γι' αυτό θα πρέπει να προσπαθήσετε να οδηγηθείτε στις κατάλληλες επενδύσεις. Ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο δεχόμαστε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και να προωθήσει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν θέλετε όμως να διευρύνετε τη δυνατότητα δράσης, γιατί καθυστερήσατε την ε, κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας. Αν θέλετε να σταματήσετε την, ε, την χρήση όπλων και την ε, διάδοση όπλων, γιατί δεχόσαστε την ασπίδα την ε, ασπίδα αυτή όπλων και βαλιστικών πυράβλων. Πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολο να μην δεχτούμε αυτό το πλαίσιο και χρειάζεται μία ε, κοινή δράση. Βεβαίως σφάλουν και οι δύο πλευρές. Χρειάζεται λοιπόν και άμεση κατάπαυση του πυρός και στο, στην ε, λωρίδα της Γάζας. Βεβαίως η Χαμάς φέρει μεγάλη ευθύνη, αλλά θα πρέπει να δούμε τις ευθύνες και των δύο πλευρών. Εσείς μιλάτε, μιλάτε για Ευρώπη χωρίς σύνορα και προσκόμματα. Θα πρέπει να προστατευτούμε όχι ε, με φράκτες, αλλά να προστατευτούμε με πολλούς φίλους. Πιστεύω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σαν την Σοβιετική, την πρώην Σοβιετική Ένωση. Όποιος θέλει να μείνει στο περιθώριο μπορεί να το κάνει, αλλά αυτή είναι μια ένωση φίλων. Φίλων, ίσων φίλων και ίσων εταίρων. Έχετε φιλόδοξους στόχους και τους υποστηρίζουμε. Εάν αρκεστείτε σε αυτούς, τότε εμείς θα σας υποστηρίξουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μπραν Κρόλι, εκ μέρου ε, τη ε, πολιτική ομάδα ε, Ευρώπη τη ΟΕΝ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, οι πολιτικές σχέσεις για να δημιουργηθούν μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ΕΠΑ πρέπει να γίνουν προσπάθειες να βελτιωθούν και ελπίζω ότι η τσεχική δημοκρατία θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό το εξάμεινο που ακολουθεί. Θα έχουμε νέο πρόεδρο τον ΗΠΑ την επόμενη εβδομάδα. Αντιμετωπίζουμε όλοι σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τα προβλήματα που ανακύπτουν και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ταχύτερο δυνατόν. Λοιπόν, σήμερα καλωσορίζουμε την Προεδρία της Δημοκρατία Δημοκρατίας που αναλαμβάνει την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε πολύ κρίσιμες στιγμές και εκ μέρους της ομάδας μας της Ευρώπης των Εθνών υποστηρίζουμε και την υποστήριξή μας προς το πρόγραμμά σας. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ισχυρότερη φωνή που θα εκφράσει την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τα κράτη-μέλη αυτής. Πολλοί συνάδελφοι ήδη αναφέρθηκαν στην σειρά κρίσεων που αντιμετωπίζουμε και θα πρέπει να αποτίσω φόρο τιμής και στην Προεδρία σας και στον Πρόεδρο Μπαρόσο για την αποφασιστική δράση που αναλήφθη όταν το θέμα της διακοπής παροχής φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ετέθη. Και όχι μόνο διότι θέλουμε να βρούμε ποιο ε, φταίει, αλλά γιατί παρενέβημε σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό επίπεδο. Ούτω ώστε να ξεκινήσουν συνομιλίε οι δύο πλευρέ, γιατί πριν δεν συνομιλούσαν. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να επεκταθεί αυτή η ιδέα της ανατολικής ε, εταιρική σχέση. Να κοιτάξουμε στην Ανατολή και προ τα Βαλκάνια, διότι εκεί βρίσκονται τα ρήγματα στην Ευρώπη. Όχι μόνο λόγω πολιτική ασταθία, αλλά και λόγω αλληλεξάρτηση που έχουμε όσον αφορά οικονομική δραστηριότητα και ενέργεια. Και τέλο, διότι έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, Θέλω να πω ότι αναφερθήκατε στην πέμπτη ελευθερία, την ελευθερία τη μετακινήσεω τη γνώσεω. Και αυτή η γνώση μπορεί να μα δώσει τα εργαλεία που τώρα μα χρειάζονται για προχωρήσουμε προς καινοτομία και έρευνα και τη δημιουργία δεξιοτήτων από την ιστορία σας κύριε Προεδρεύοντα σαν χώρα. Από ολοκληρωτισμό προς ελευθερία. Προς βελτίωση της παιδείας και της καινοτομίας. Προσβλέπουμε προς εσάς να μας οδηγήσετε στο επόμενο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνω. Παράθεση. Τζον F. Kennedy, όταν λέβεται καθήκοντά του, είπε «Σήμερα είμαστε μπροστά στα νέα σύνορα τα νέα σύνορα που αναφέρω δεν είναι υποσχέσεις αλλά προκλήσεις. Ξέρω ότι έχετε δυνατότητα να αντιμετωπίσετε αυτές τις προκλήσεις. Σας ευχαριστώ. Κυρία Φρασόν, εκ μέρους των Πρασίνων για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή που γίνεται συζήτηση πέφτουν βόμβες στη Γάζα και νομίζω ότι η μέγιστη προτεραιότητά μας και του Συμβουλίου και της Επιτροπής θα ήταν να σταματήσει σταματήσουμε τη ρήψη βομβών στους ανθρώπους της Γάζας. Αυτή, αυτό είναι το καθήκον μας πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας και την απόδοση ευθυνών. Εμείς οι πράσινοι έχουμε σαφή ιδέα επ' αυτό όπως θα πούμε το απόγευμα. Εσείς αρχίσατε μιλώντας ε, για τον Μεσαίωνα, για τον σκοταδισμό Υπήρχε βεβαίως μία ακτίδα φωτός, αλλά επικρατούσε σκοταδισμός και στο πρόγραμμά σας, πέρα από τις προσπάθειες που καταβάλλετε, βλέπουμε ότι υπάρχει μία θεώρηση του παρελθόντος. Δηλαδή είσαστε συμβατικοί για την αγορά και για τα οικονομικά συμφέροντα. Αυτά είναι εκτός σύρμου, κύριε Προεδρεύοντα. Μιλάτε για κανόνες, για ρύθμιση, για εταιρικές σχέσεις που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Μιλάμε για το περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές που φέρουν ένα κόστος. Μιλάτε για ένα πρόσκομα και όχι για ευκαιρία καινοτομία και ανάπτυξης. Και θα ήθελα να πω ότι είναι κάπως παροχημένη η θεώρησή σας όταν μιλάτε για το, τους στόχους της Βαρκελόνης. Γιατί μιλάτε γιατί, για το γεγονός ότι θα πρέπει να αποστείλουμε τις γυναίκες πάλι πίσω σπίτι σπίτι για να ασχοληθούν τα, με τα παιδιά. Αυτό είναι και κάπως εξιστικό. Επίσης, μιλάτε για πολυμερείς σχέσεις χωρίς να τονίζετε αυτό που είναι σημαντικό για μας. Μία σύγκληση, σύγκληση ως προς την εξωτερική πολιτική. Επίσης, δεν γίνεται μνήα του τομέα κατά των διακρίσεων και θα ήθελα να ξέρω ποιες είναι οι προτεραιότητές σας γιατί μιλάτε μόνο για την οδηγία κατά των διακρίσεων και την έγκριση της. Υπάρχει όμως κόσμος με μεγάλους κινδύνους και λίγες ευκαιρίες. Μιλάμε και για την διαφορά Ρωσίας-Ουκρανίας. Δεν βλέπουμε όμως να διανοίγεται μία οδός αντιμετώπισης, διότι η Σλοβακία και η Βουλγαρία θέλουν να ξανανοίξουν τους πυρηνικούς αντιδραστήρες που είναι ε, παροχημένη. Δεν υπάρχουν ασφαλή πυρηνικά πλέον κύριε Πρόεδρε, άρα ας μην συζητάμε για αυτά, γιατί πρόκειται για ένα δαπανηρό εγχείρημα που μας αποσπά από τους πραγματικούς στόχους. Επίσης μιλάμε για την αλληλεγγύη, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πραγματικά ενεργειακή αποταμίευση. Θα πρέπει να δούμε πώς ε, φτάνουμε στη μείωση της κατανάλωσης, αλλά φτάνουμε σε έναν πόλεμο, τον πόλεμο του φυσικού αερίου. Θα πρέπει να πείσετε τους συναδέλφους να θέσετε στο επίκεντρο της Ερηνής Συνόδου τον στόχο του 20% ε, ενεργειακής αποταμίευσης μέχρι το 2020 σε σχέση με το περσινό πακέτο και να ξαναδείτε τις προτεραιότητές σας έτσι ώστε να μην είναι τόσο επιφανειακές οι αποφάσεις σας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε σχέση με το μέλλον της Ευρώπης, η συνθήκη της Λισαβόνης δεν είναι τέλεια, αλλά είναι περίεργο γιατί δεν την έχετε κυρώσει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να μας εξηγήσετε γιατί και να μας πείτε πότε θα το κάνετε ίσως. Ευχαριστώ πολύ. Äh, τώρα, εξ ονόματος ε, της Ενωμένης Αριστεράς, ο κύριος Ρανστοφ για τρία λεπτά. Πρόεδρε, Ο Προεδρεύων, ο κύριος ε, Τοπολάνεφ, ε, μίλησε για τις ε, εμπειρίες μας, τις δύσκολες εμπειρίες μας από τη Ρωσία. Νομίζω η Τσεχική Προεδρία είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τη διέρεση της Ευρώπης σε Ανατολή και Δύση. Πού υπάρχει αυτή τη στιγμή ο κύριος Γιούσλαφ Χάσεφ στο βιβλίο του για τον στρατιώτη Σβέικ χρησιμοποιεί μία ρίση που αν τη μεταφράσει κανείς ελεύθερα καταδεικνύει ότι η Δύση δίνει και η Ανατολή παίρνει. Αυτή όμως η διαίρεση πρέπει να πάψει να υπάρχει και η ε, Τσεχική Προεδρία είναι μια ευκαιρία για να ξεπεράσουμε όλες αυτές τις ε, προκαταλήψεις. Παράδειγμα το άρθρο του κυρίου Κλάους όπου ε, δίνει συμβουλές για την αντιμετώπιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Δείχνει λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή αποδυναμώνονται ε, τα κοινωνικά πρότυπα γιατί από ό,τι φαίνεται Τα πρότυπα αυτά αποτελούν εμπόδιο για τις ε, ενέργειες ε, των κρατών. Θεωρώ λοιπόν ότι πλέον εσείς έχετε την ευκαιρία να αποδείξετε ότι με τα ε, σωστά πρότυπα και σωστές προδιαγραφές μπορούμε να επιτύχουμε αναθέρμανση της οικονομίας. Σε ένα θέμα, συμφωνώ με τον κύριο Τοπολάνικ, πρέπει να επενδύσουμε στις καινοτομίες. Αυτό είναι το εργαλείο που θα μας ε, οδηγήσει έξω από την κρίση. Οφείλουμε λοιπόν να αναζητήσουμε όλες τις ε, δυνατότητες έτσι ώστε οι οικονομίες μας να βγουν από το αδιέξοδο. Και εδώ θέλω να σας πω ότι το θάρρος ε, για την αλλαγή το χρειαζόμαστε όλοι. Ένας Γερμανός μεγάλος φιλόσοφος είπε ότι το μέλλον ανήκει σε εκείνους που έχουν το θάρρος να αλλάξουν. Θέλω λοιπόν να ελπίζω ότι και εμείς θα έχουμε το θάρρος να αλλάξουμε και να προσανατολιστούμε σε μια νέα ιστορία, να ξεπεράσουμε ε, το χάσμα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση, μια νέα Ευρώπη η οποία δεν θα έχει συμπλέγματα κατωτερότητας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε άλλες χώρες. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω το εξής. Ο Πρωθυπουργό ε, κύριος Τοπολάνεκ έθιξε πολλούς ε, ιερούς στόχους και κοινά συμφέροντα. Σωστό αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν φιλόδοξα προγράμματα. Εγώ όμως ε, είμαι και λιγάκι επιφυλακτικός. Ένας Πολωνός ε, συγγραφέας είπε ότι το να συμμετέχει κανείς σε ένα ταξίδι αυτό δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ε, είναι ένα ταξίδι που οδηγεί στη Ρώμη ο κ. Ζελέσνη. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή που αναλαμβάνει τη καθηκοντά της Τσεχική Προεδρία. Ποτέ δεν είχε γίνει αυτό πρώτο. Ο γαλλικός τύπος έκανε ό,τι μπορούσε για να σχεδιάσει μια ζωφερή εικόνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που θα επηρεαστεί από την Τσεχική Προεδρία διότι οι Τσέχοι δεν είναι ικανή. κυρίως ακολουθώντας μια Προεδρία που ήταν τόσο ικανή όπως η Γαλλική Προεδρία και ο Γάλλος Πρόεδρος. Και ποιο ήταν το σφάλμα των Τσέχων που δεν κύρωσαν την ε, συνθήκη της Αβώνας. Έχουν έναν πολύ ικανό πρόεδρο που είναι κατά της ε, συνθήκης της Αβώνας ε, και αναφέρεται όμως στο αυξανόμενο δημοκρατικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ένα τέτοιο έλλειμμα μας έκανε να ρίξουμε τον κομμουνισμό εδώ και 20 χρόνια. Η τσεχική ε, προεδρία θα είναι επιτυχής, έχει λογικούς στόχους και πρέπει να της ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Παρά τις κραυγές, τις ντροπιαστικές των σοσιαλιστών, ε, σοσιαλιστών που πρόδωσαν τη χώρα τους για τον ολοκληρωτισμό προσπαθούν τώρα να εμποδίσουν την προεδρία. Στο κάνουν οι σοσιαλιστές οι Τσέχοι θα πρέπει να αποδείξει η εχική δημοκρατία ότι δεν είναι ανίκανε οι μικρές χώρες και ότι μέσω της συνθήκης της Λισαβόνα θα δώσουμε ε, τα σωστά μέσα στην Ευρωπαϊκή να σε προχωρήσει. Γι' αυτό η τσεχική προεδρία είναι τόσο σημαντική. Θα δείξει ότι ακόμα και μικρότερες χώρες μπορούν να διοργανώσουν μια προεδρία χωρίς να είναι μεγαλομανείς, εγωιστές και να είναι ιστερικές όσον αφορά τις σχέση τους με το κοινό και εύχομαι στον Πρωθυπουργό και τον Πολάνεκ κάθε επιτυχία διότι θα είναι επιτυχία της χώρας μου αυτή και μιας μικρής χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της εμπειρίας μας. Οι μεγαλύτερες δημοκρατίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως ζούσαν υπό προβλεπόμενες συνθήκες. Εμείς όμως επί 50 χρόνια πρέπει να ζούμε ε, σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και αυτό θα μας είναι χρήσιμο τώρα. Συνάδελφε, είσαστε Ευρωπαίος γιατί είσαστε Τσέχος. Εκ μέρου ε, των ε, μη γεγραμμένων, η επόμενη ομιλήτρια για τέσσερα λεπτά, κύριε Μπομποσίκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, Ήταν πολύ δραστήρια η Τσεχική Προεδρία όταν αντιμετώπισε το θέμα της Γάζας και το πρόβλημα του φυσικού αερίου. Ε, ο κ. Πολάνεκ μπορεί να δείξει παρόμοια πρωτοβουλία και τώρα για τις διαπραγματεύσεις για τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο προεδρεύων του Συμβουλίου θα πρέπει να έχει τη φιλοδοξία να ηγείται των προσπαθειών. Έχετε μοναδική ευκαιρία να αποδείξετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ομάδα κρατών μελών που είναι ισότιμη εταίρη και τότε μπορείτε πράγματι να γράψετε ιστορία. Αγαπητέ Πρόεδρε, έχετε την ευκαιρία και τη δύναμη να δηλώσετε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι νεκρή μετά το Ιρλανδικό δημοψήφισμα. Ήταν αδιέξοδο τότε. Μπορείτε να προτείνετε ένα νέο οραματικό έγγραφο που θα συμπεριλαμβάνει έναν κοινό παρανομαστή των συμφερόντων των κρατών μελών και να μπορούν να ταυτιστούν οι λαοί με κάτι τέτοιο. Μπορείτε να σταματήσετε από την πρόθεση της κυρώσεως της συνθήκης της Λισαβόνας που επιβάλλει με μη δημοκρατικό τρόπο την ισχύ των γραφειοκρατών. Κύριε Πρόεδρευοντα, ε, εκπροσωπείται μια χώρα που απελευθερώθηκε από την Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία που μπόρεσε να αντιμετωπίσει τον τρόμο του ναζισμού και την ε, ε, εισβολή των στατευμάτων του Συμφώνου της Βαρσοβίας και ήσασταν σε μια χώρα που ήταν υπό την επιρροή της Σοβιετικής Ενώσεως και ζούσε σε φτώχεια ε, των χωρών της Κομεκών. Και μπόρεσε να απελευθερωθεί η χώρα σας. Δεν μπορώ να πιστέψω λοιπόν ότι εσείς με μια τέτοια ιστορική εμπειρία θέλετε η κοινωνική, η πολιτική, η ενέργεια, η φόροι, η δικαιοσύνη, όλα αυτά να αποφασίζονται αλλού και όχι στα κράτη-μέλη. Δεν πιστεύω ότι εσείς θέλετε να ισχύουν οι αποκλειστικές εξουσίες της Ενώσεως που θα υπερέχουν των εξουσιών των κρατών μελών. Δεν πιστεύω ότι θέλετε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρεμβαίνει όσον αφορά την προστασία και προώθηση της ανθρώπινης υγείας, την παιδεία, τον αθλητισμό κλπ. Ε, δεν πιστεύω ότι καλωσορίζει το γεγονό ότι η συνθήκη τη Αβώνα καταργεί το δικαίωμα τη αρνησικηρία σε πάνω από 50 τομεί και επίσης ότι μειώνει και το βάρος των μικρών χωρών συμπεριλαμβανόμενη τη δημοκρατίας. Θα πρέπει να έχετε λοιπόν το θάρρος ε, να πείτε στα 26 άλλα κράτη-μέλη, στου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων, αυτό που λέτε κατηδίαν στην τσεχική δημοκρατία. Θα πρέπει να πείτε ότι η συνθήκη τη Σαββόνα δεν είναι καλή. Δεν θα σα χειροκροτήσουν οι ευρωπαϊστέ, οι τεχνοκράτε Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όμω θα σα σεβαστούν οι πολίτε που αγνοούνται Ψυχνάκης και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι προεδρεύεται 450 ε, εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι μιας ομάδας τεχνοκρατών και πολιτικών. Στην τσεχική δημοκρατία λέτε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι αναγκαίο κακό. Αλλά γιατί είναι αναγκαία. Γιατί είναι αναγκαίο. Δεν είναι αναγκαίο κακό, απλώς είναι κακό. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσετε την επεξεργασία ενός εγγράφου που θα εμπνέεται από τη συστήκη της Ρώμης από τη διακήρυξη της Μεσίνας και θα πρέπει να προωθήσετε τα κοινά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και όχι τα συμφέροντα των ε, διαφόρων Ευρωπαίων γραφειοκρατών. Αναγκαίο κακό είναι άλοθη ε, δηλών. Δεν είστε δηλός όμως, έχετε την υποστήριξη του ιλλανδικού Δημοψηφίσματος, 55% των πολιτών μας και έχετε την ισχυρή φωνή του Προέδρου μας, του κυρίου Κλάους και εσείς θα πρέπει να ξέρετε τι πρέπει να γίνει και να μην κάνετε αυτό που δεν πρέπει να γίνει. Πρόεδρος, πολύ ωραία. Θα έχουμε λοιπόν τώρα μία πρώτη απάντηση, πρώτη αντίδραση εκ μέρους του κυρίου Τοπολάνα και μετά, και μετά του κυρίου Μπαρόζου. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας, για τις σύντομες ομιλίες σας. Και στην Τσεχία έχουμε κοινοβούλιο και είμαστε συνηθισμένοι να μην έχουν όλη την ίδια άποψη. Παρ' όλα αυτά ομολογώ ότι ξεπλάγινα από κάποιες απόψεις που άκουσα με τις οποίες διαφωνώ κάθετα. Εγώ είμαι πραγματικά ακράδαντα πεπισμένος ότι ως ε, Πρωθυπουργός ε, και ως Προεδρεύον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, οφείλω να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις, να μην τοποθετηθώ προσωπικά, όμως θα τοποθετηθώ σε κάτι που ήταν επί προσωπικού κάποια σκληρά λόγια για τον Τσέχο Πρόεδρο, τον κύριο Κλάους. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, γνωρίζουν τον κύριο Βλάτσαφ Κλάους και είμαι υπερήφανος γι' αυτό, γιατί είναι εικόνα της αλλαγής που έλαβε χώρα στην πατρίδα μας και με τη δική του την υποστήριξη μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τα δέκα πρώτα προβληματικά χρόνια. Σε αυτόν οφείλουμε το ότι το 1991 εκδιώξαμε τους ε, Ρώσους ε, στρατιώτες από τη χώρα μας, είχαμε την ανέμακτη επανάσταση, προσχωρήσαμε στο ΝΑΤΟ το 2004 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρυσι ανοίξαμε τα σύνορα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα μπορεί κανείς να ταξιδέψει χωρίς κανένα ταξιδιωτικό έγγραφο από την Ισπανία μέχρι το Βίλνις. Εγώ είμαι υπερήφανος που τα έζησα όλα αυτά και σήμερα που βρίσκομαι μπροστά σας ε, Ε, πραγματικά κλείσουμε γιατί ελέγξαν όλα αυτά εις βάρος του Πρόεδρου. Εμείς ε, έχουμε την Προεδρία, πληθυσμιακά είμαστε μικρότερη χώρα. Παρόλα αυτά όμως δεν θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χάσει την ευκαιρία να έχουμε ανοιχτή συζήτηση θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούμε να εκφράζουμε τη γνώμη μας ε, με απόλυτη ελευθερία. Γιατί αν δεν συμβαίνει αυτό ε, θα ήταν ένα τραγικό λάθος. Και γι' αυτό πρέπει να διαφωνήσουμε αυτά που ελέγχθησαν για τον πρόεδρό μας. Διότι ο πρόεδρος μας έχει μια μοναδική ικανότητα να παρουσιάζει νέες παραμέτρους ε, στις ε, συζητήσεις. Η ελεύθερη έκφραση απόψεων, ε, αυτό πρέπει να συνεχίσει να ισχύει και δεν μπορούμε να θελήσουμε να την περιορίσουμε. Όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας, θέλω να πω κάτι από αυτού. Η συνθήκη αυτή ίσως να είναι χειρότερη από αυτή της Νίκαιας και ίσως λίγο καλύτερη από αυτή που ισχύει τώρα. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ τα πράγματα. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι εγώ διαπραγματεύτηκα εκ μέρους ε, της ε, Τσεχίας για αυτή τη συνθήκη. Η συνθήκη αυτή κυρώθηκε εκ μέρους της κυβέρνησης. Εγώ προσωπικά υπέγραψα σε αυτή τη συνθήκη και το τονίζω αυτό. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη θέλουν να επιβάλλουν σε άλλα, να μην μπορούν να αποφασίζουν μόνα τους ε, κατά πόσον θέλουν να εγκρίνουν ένα έγγραφο ή όχι, αυτό μου μοιάζει παράλογο. Πάντως, οφείλουμε να αλλάξουμε τους θεσμούς. Πρέπει να ενισχύσουμε τους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, Πρέπει να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τους κανόνες. Τώρα κατά πόσο αυτό θα το επιτύχει η συνθήκη της Λισαβόνας δεν το γνωρίζω. Οι απόψεις δίστανται επ' αυτού. Κυρία Μπουσίκοβα, για μένα η συνθήκη της Λισαβόνας είναι το αποτέλεσμα συμβιβασμών. Ίσως ε, περίπλοκων συμβιβασμών, όμως εγώ θα υποστηρίξω την κύρωση της συνθήκης. Και τώρα θα μου επιτρέψετε λίγα λόγια που αφορούν στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ συχνά αναφέρεται ως big payer αλλά όχι big player που σημαίνει ότι όσον αφορά τις επενδύσεις εμείς πράγματι συμμετέχουμε σημαντικά, ε, χορηγούμε οικονομική, ανθρωπιστική βοήθεια αλλά πολλές φορές αναφέρεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρώσεις της ε, στο πλαίσιο του, των, της τετραμερούς. Έχοντας κατά νου τη νέα αμερικανική κυβέρνηση, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να επενδύουμε μόνο με, να επενδύουμε κονδύλια, αλλά να συμμετέχουμε σε μια ενεργό πολιτική. Το Ισραήλ έχει δικαίωμα ασφάλειας, έχει δικαίωμα να ζει χωρίς ε, να δέχεται πυράβλους. Εγώ ίδιος ε, πήγα στο Ασκελόν και θεωρώ ότι και ο λαός της Παλαιστίνης έχει το δικαίωμα να οικοδομήσει κράτος και αυτός ο λαός έχει το δικαίωμα ε, της σε ασφάλεια. Μέχρι τώρα κανείς δεν μπόρεσε να βρει μια ικανοποιητική λύση. Εμείς θα προτείνουμε βραχυπρόθεσμα μέτρα, κυρίως στην κατάπαυση του πυρός και κάτω από αυτό το πρίσμα θα ήθελα να σας επισημάνω ότι ο κύριος Σβάτσενμπεργκ και η αντιπροσωπεία του έπαιξαν σημαντικό ρόλο αναζητώντας τη λύση. Τα αραβικά κράτη, η Αίγυπτος, η Τουρκία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι το να υπάρξει εμπάργο όπλων ε, στη Γάζα. Αυτό μπορούμε να το επιτύχουμε από κοινού ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος μας πρέπει να είναι να επιδιώξουμε την κατάπαυση των εχθροπραξιών. Βεβαίως δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αυτό θα μπορέσουμε να το επιτύχουμε σύντομα. Όσον αφορά τώρα την ενέργεια και την ε, κλιματική αλλαγή, η Ευρωπαϊκή Ένωση διδραματίζει σημαντικό ρόλο όσον αφορά αυτό το θέμα. Ε, νομίζω όλοι μας ε, οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι στον τομέα των κλιματικών αλλαγών δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε τίποτα αν δεν συνεργαστούμε όλοι. Ευρώπη, Βραζιλία, Κίνα, γιατί μόνη της η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να επιτύχει τίποτα. Οι προσπάθειές μας ε, θα αποβούν άκαρπες εάν δεν μπορέσουμε να κάτσουμε όλοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Στόχος μας είναι να πείσουμε τις μεγάλες χώρες να μεριμνήσουν επ' αυτού. Και νομίζω εδώ τους επόμενους έξι μήνες έχουμε να διδραματίσουμε σημαντικό ρόλο γιατί το κλιματικό πακέτο έχει αποφασιστεί και τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ε, εγκρίνει το πακέτο και να το εφαρμόσετε. Όσον αφορά τώρα το ενεργειακό μείγμα, ε, το θέμα αυτό πολλές φορές αντιμετωπίζεται ε, αμυγός ε, ιδεολογικά και πολιτικά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρειαζόμαστε όμως μια ρεαλιστική προσέγγιση όπου βραχυπρόθεσμα θα ορίσουμε στόχους και τα μέσα για να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ μια χώρα η οποία είναι κατά 90% ε, εξαρτώμενη από τον άνθρακα, όπως είναι η Πολωνία, μια τέτοια χώρα να μπορεί σε 10 ή σε 20 χρόνια να αλλάξει ριζικά αυτή την κατάσταση. Βεβαίως και πρέπει να επενδύσουμε σε νέες ε, τεχνολογίες, ε, στον άνθρακα και στην πυρηνική ενέργεια. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ύπαρξη ασφαλών πυρηνικών αντιδραστήρων. Το ενεργειακό μείγμα οφείλει να βελτιώνεται διαρκώς έτσι ώστε να προστατεύεται καλύτερα το περιβάλλον. Να μην εξαρτώμεθα τόσο πολύ από ρηκτά κάψιμα. Και επιπλέον να μπορούμε οικονομικά να εξασφαλίζουμε ε, προσιτή ενέργεια για να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί σε διεθνές επίπεδο. Η κρίση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία δεν είναι μόνο κρίση εμπιστοσύνης. Ε, στην κρίση αυτή ε, σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και άλλα θέματα, πολιτικά, ε, στρατηγικά. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα και εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να είμαι αναγκασμένος να πω ποιος είναι υπεύθυνο για αυτή την κατάσταση. Νομίζω και οι δύο χώρες φέρουν ευθύνη. Η μία χώρα δεν δίνει το αέριο και η άλλη παρεμποδίζει την περαιτέρω μεταφορά του αερίου. Οφείλουμε λοιπόν να αναζητήσουμε μία λύση για να δούμε πώς μπορούμε βραχυπρόθεσμα να αντιμετωπίσουμε το θέμα και πώς μπορούμε μακροπρόθεσμα να διαφοροποιήσουμε τις ε, ενεργειακές πηγές. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα ευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας και αερίου και τι θα κάνουμε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Δεν θέλω τώρα να παίζω το ρόλο της Κασάνδρας, αλλά η κρίση δεν έχει ξεπεραστεί. Η κατάσταση στα Βαλκάνια και στη Βουλγαρία μοιάζει να είναι απελπιστική. Θέλω να σας πω ότι έχω να κάνω και κάποιες άλλες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που είπαν οι επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Νομίζω ότι η δική μας ημερήσια διάταξη δεν είναι τόσο φιλελεύθερη. Εμείς ε, ε, βασιζόμαστε στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο φύλλο πορείας που μας έδωσαν οι προηγούμενοι. Μέσα σε 14 ημέρες αποδείχθηκε λοιπόν ότι επιλέξαμε τους σωστούς στόχους. Ποτέ δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι την 1η Ιανουαρίου στις 12 και 5 ακριβώς θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε τόσο σημαντικά θέματα που να έχουν σχέση με το φυσικό αέριο, με την ενέργεια, την ενεργειακή ασφάλεια. Δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε αυτό. Και επιτρέψτε μου να κάνω και μία ε, παρατήρηση για τα κοινωνικά θέματα. Ε, είναι προφανές ότι εμείς ε, προσπαθήσαμε να επεξεργαστούμε και να ορίσουμε κάπως συμβολικά τους βασικούς στόχους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η κατάργηση διακριτικών μεταχειρήσεων είναι καθοριστική σημασίας. Και εμείς σε εθνικό επίπεδο. Έχουμε κάνει τη σχετική εμπειρία. Στην περίπτωση των, ε, του, ε, εξανα, της εξαναγκαστικής παραμονής παιδιών σε κάποια απομακρυσμένα μέρη στο βορρά. Είναι πολύ σημαντικό οι γονείς μόνοι τους αποφασίζουν τι θα κάνουν με τα παιδιά τους. Να μπορούν να εργάζονται και να διασφαλίζουν την οικονομική επιβίωση της οικογένειας. Βεβαίως, ε, η μέρημνα για τα παιδιά είναι πολύ σημαντική για να γίνουν όλα αυτά. Η, η Τσεχία ε, έχει κάνει πολλές δυσάρτητες εμπειρίες γιατί ε, κατά την περίοδο του ολοκληρωτισμού αυτή η αρχή που τώρα σας προανέφερα παραβιάστηκε επανειλημμένα. Αυτά είχα ε, να πω εν είδη εισαγωγής. δεν είναι ότι μας λείπει η αυτοπεποίθηση κάθε άλλο. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από πλευράς ε, πληθυσμιακής είμαστε κάπου στη μέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε ούτε οι σημαντικότεροι ούτε και οι μικρότεροι. Δεν έχουμε σύμπλεγμα κατωτερότητας. Όταν και η Σουηδία είχε την πρώτη της Προεδρία και εκείνη ήταν πρωτάρα, όπως είμαστε και εμείς σήμερα. Και τότε τους ε, είχαν κατηγορήσει ότι οι ε, σκεπτικιστές ε, στη Σουηδία που δεν είχαν καν εισαγάγει το ευρώ ότι αυτοί ε, δεν θα ήταν σε θέση να δρομολογήσουν συζητήσεις για την κύρωση της συνθήκης της Νίκαιας. Πολλοί τότε είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το κατά πόσον οι Σουηδοί θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ηγετικό ρόλο και εμεί τώρα βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Αλλά σας τονίζω και για άλλη μια φορά, εμείς συμπλέγματα κατωτερότητε δεν έχουμε. Ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Μπαρόζο, δεν θα παρέμβει μια δεύτερη φορά και ερχόμαστε στον κατάλογο των ομιλητών μα, Ο κ. Ζαχραλντή έχει το λόγο. Για δύο λεπτά. Προσπαθήστε να είστε συνεπεί στον χρόνο που σα έχει ε, διατεθεί για να μπορέσουμε να πάμε ομαλά στι ψηφοφορίε. Ευχαριστώ. Κύριε Προεδρεύοντα, θα σταθώ στην τσεχική θεώρηση των πραγμάτων, όπως τονίσατε στην ομιλία σας. Βλέπουμε ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές θα διενεργηθούν σχετικά σύντομα, άρα ίσως υπάρξουν πολύ μεγάλες ε, συνεισφορές μέσα στα πλαίσια της ε, προεκλογικής εκστρατείας σε σχέση με τις προτεραιότητες που μας ε, καταθέσατε εδώ. Νομίζω ότι οι πρώτες μέρες της ε, Τσεχικής Προεδρίας ήταν μια πραγματική δοκιμή και δοκιμασία για την Τσεχική κυβέρνηση και ανταποκρίθηκε σε αυτή την ε, δοκιμασία η Τσεχική κυβέρνηση και η οικονομία, ενέργεια και εξωτερικές σχέσεις, οι τρεις προτεραιότητες, δηλαδή το τρίπτυχο αυτό της Τσεχικής Προεδρίας, επελέγει πολύ σωστά, διότι αυτό που συνέβη στις αρχές του έτους ήταν το εξή. Η Γάζα και η κρίση του φυσικού αερίου εμπίπτουν στις δύο από τις τρεις αυτές προτεραιότητες. Βλέπουμε λοιπόν σαφώς ότι το θέμα της ενέργειας είναι ύψης της σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο μέλλον, πολύ πιο σημαντικό από άλλα θέματα όπως ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας, διότι η συνθήκη της ε, ε, Λισαβόνας δεν θα μας παράσχει ούτε ηλεκτρικό ούτε θέρμανση. Αυτό αποτελεί λοιπόν μεγάλη πρόκληση για την Τσεχική Προεδρία και αποτελεί τιμή για μας να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στην πρόοδο αυτού του θέματος και οι τρεις αυτές προτεραιότητες είναι αλληλένδετες διότι το φυσικό αέριο έχει επίπτωση στην οικονομία καθώς και επίπτωση στις εξωτερικές σχέσεις γιατί θα πρέπει να υπάρχουν ε, να υπάρχουν άρρηκτοι δεσμοί με τους γείτονες, όπως παραδείγματος χάρη με την Τουρκία, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρχει ασφάλεια προμηθειών η διαφοροποίηση των πηγών. Ελπίζω λοιπόν ότι η Τσεχική Προεδρία θα μπορέσει να συνεισφέρει σε, αυτή την, ε, σε αυτό το εξάμεινο επικοδομητικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαχραντή. Ο κύριος Ρούτσεκ για τρία λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα, τον κύριο Τοπολάνεκ, καθώς και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής. Ε, κυρίες και κύριοι, όλα τα μέλη ε, επιθυμούν την επιτυχία της Τσεχικής Προεδρίας. Τα παλαιότερα ή τα νεότερα κράτη-μέλη όλα επιθυμούν την ε, επιτυχία αυτού του εγχειρήματος και ευχόμαστε κάθε επιτυχία και στην Τσεχική Προεδρία μεταξύ άλλων. Ανεξάρτητα από την ε, πολιτική συνιστόσα ή το πολιτικό κόμμα στο οποίο ανήκουν. Δυστυχώς όμως και πρέπει να το τονίσω αυτό, υπάρχουν ε, ορισμένοι φόβοι για το κατά πόσον ε, η τσεχική προεδρία θα μπορέσει να επιτύχει και υπάρχει πληθώρα λόγων γι' αυτόν. Καταρχήν υπάρχει έλλειψη σταθερότητας μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής ε, συμμαχίας. Εμείς δεν κατανοούμε γιατί στην αρχή της Προεδρίας αποφασίσατε αυτό τον κυβερνητικό ανασχηματισμό. Αυτό δείχνει μία σαθρότητα του συστήματος όπου είχαμε νέους υπουργούς ε, μεταξύ αυτών και τον νέο υπουργό μεταφορών. Τα μέλη αυτά είναι νέα, άπειρα και ξέρετε ότι οι χριστιανοδημοκράτες αποφάσισαν να διοργανώσουν ε, την ε, διάσκεψή τους κατά τη διάρκεια της τσεχικής προεδρίας. Θα ήθελα μία σαφή απάντηση για αυτή την πολιτική συμμαχία και τον πολιτικό συνασπισμό και κατά πόσο συμφωνείτε με τον πρόεδρο Κλάους, ο οποίος απορρίπτει τη συνθήκη της Λισαβόνας και δεν δέχεται ότι υπάρχει θέμα κλιματικών αλλαγών και υπερθέρμανσης του πλανήτη. Και η χρηματοπιστωτική κρίση έχει πηγές κακοδαιμονίας και τα αίτια αυτά μπορούν να αναλυθούν, όπως έκανε και η καγκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος Σαρκοζή. Πιστεύετε ότι θα ακυρώσετε την ε, συνθήκη της Λισαβόνας. Πότε θα ακυρωθεί από το τσεχικό κοινοβούλιο και γιατί καθυστερεί τόσο πολύ η κύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας που θα έπρεπε να γίνει πέρσι τον Δεκέμβρη. Και τι θα γίνει με την διμερή συμφωνία ως προς την ε, πυραυλική ασπίδα. Ακούσαμε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας είναι απόλυτα αναγκαία και για τις τσεχικές ε, προτεραιότητες. Την χρειαζόμαστε λοιπόν για να επιτελεστεί πρόοδος σε θέματα ενέργειας, για να υπάρχει συμπληρωματική συνεργασία σε άλλους τομείς και, εν πάση περιπτώσει, σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Μόνο σεβαστείτε, κύριε συνάδελφοι. Η κυρία Κόσο έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ε... Η Ευρωπαϊκή Ένωση έζησε έξι μήνες ε, Σαρκοζή με δράμα, δυναμική και δηλώσεις. Και τώρα λαμβάνετε εσείς ε, με ένα χιούμορ το οποίο πρώτα απ' όλα πρέπει να το συνηθίσουμε. Εμείς ε, ελπίζουμε να είσαστε επικοδομητικός πρόεδρος γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλές προκλήσεις. Εσείς ο ίδιος μιλήσατε για τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και για την οικονομική κρίση. Ε, κρεμούν και εσωτερικά θέματα η συνθήκη της Λισαβόνας. Όμως θα αναφερθώ σε ένα σημείο της ομιλίας σας στην ενεργειακή ασφάλεια. Ε, θίξατε την ε, θεμελιώδη σημασία αυτού του θέματος. Συμφωνώ, η ενέργεια είναι ε, το βασικό αγαθό της σύγχρονης κοινωνίας. Το, ο τρόπος διαβίωσής μας, η περαιτέρω ανάπτυξή μας εξαρτάται από αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε εξαρτώμενοι από την ενέργεια. Χρειαζόμαστε ένα καλό μείγμα από διαφορετικές πηγές ενέργειας για να είμαστε ανεξάρτητοι. Γι' αυτό και εγώ επιμένω για το ότι με τον ανοιχτό σας τρόπο αντιμετώπιση των πραγμάτων μπορείτε να κινητοποιήσετε τους Ευρωπαίου σε μια νέα συζήτηση για την ενέργεια. Ε, να ε, πείσετε την γερμανική κυβέρνηση να αποσυρθεί από την πυρηνική ενέργεια. Αυτό το επιβάλλει η πυρός μας. Ακόμα υπολείπονται πάρα πολλά, υπάρχουν όμως και πολλές ευκαιρίες για να προχωρήσει η Ευρώπη. Σας ε, εμπιστεύομαι, σας ευχαριστώ και προσβλέπω σε καλή συνεργασία. Ο κύριος Σουμάσκι έχει το λόγο τώρα για ένα λεπτό. Όπως ξέρετε υπάρχει ένα κριτήριο για την επιτυχία της Τσεχικής Προεδρίας που τόνισε και η κυβέρνησή σας, δηλαδή η ενεργειακή πολιτική στο, βρισκόμαστε στο τέλος αυτού του κεφαλαίου της διαφοράς ε, μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, αλλά δεν υπάρχει πολιτικό πλαίσιο έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον. Μετά από την ενεργειακή κρίση του 2004, 2005 και 2006, θα πρέπει να αρχίσουμε αυτή την εργασία διαφοροποίησης ως προς τους ενεργειακούς πόρους και τις πρώτες ύλες. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε χρηματοδοτική υποστήριξη για τον αγωγό του Ναμπούκο. Ελπίζουμε να ληφθούν μέτρα έτσι ώστε να μην ε, υπάρχουν αυτές οι προτεραιότητες που είχαμε μέχρι τώρα και πιστεύουμε ότι διαφορετικά θα έχουμε μεγάλα προβλήματα του χρόνου το χειμώνα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα, το θέμα ενεργειακό, αφορά την αξιοπιστία της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Μπαγούζο για τα σαφέστατα λόγια σας σήμερα το πρωί. Για την Gazprom και την Αυσποζά Gas, ε, εδώ τέσσερις πέντε μέρες λένε απίστευτα πράγματα. Και πρέπει να πούμε, κύριοι, φτάνει. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να κινηθούμε μαζί, ομού. Ευχαριστώ που τα συντονίσατε καλά τα πράγματα. Υπάρχει κανείς εδώ που πάμε εξηγήσει το ταξίδι του Σλοβάκου Πρωθυπουργού και του Βουλγάρου Πρωθυπουργού στη Μόσχα. Τι είναι αυτό, τι πράγματα είναι αυτά. Ήδη δείχνουμε στην ΚΑΣΠΡΟΜΟ ότι δεν είμαστε ενωμένοι. Δώστε μου μια εξήγηση λοιπόν για τα δύο ταξίδια. Δεύτερον και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει μεγάλο ρόλο να παίξει σε αυτό. Πρέπει να καταρτήσουμε σχέδιο κατεπήγων για το φυσικό αέριο. Το πρώτο πράγμα είναι να αναδιαμορφώσουμε την οδηγία για την ασφάλεια του φυσικού αερίου. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έχει αρκετέ πολιτικέ εξουσίε για να δράσει. Χρειάζεται συντονισμό ευρωπαϊκό. Δεύτερον, Χρειάζεται κατεπήγον σχέδιο για υποδομές για το φυσικό αέριο για την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Με τα διαθέσιμα χρήματα. Τρίτον, θα πρέπει να συνδυαστεί η οικονομική ανάκαμψη ευρωπαϊκή με ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο για την ενέργεια. Πρώτη προτεραιότητα τα κτίρια στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι σκάνδαλο να βλέπει κανείς τόσα λίγα χρήματα από τα ταμεία να, να δίνονται σε αυτό που είναι χρήσιμο αντί να κατασκευάζονται στάδια για ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Εγώ προτιμώ να επενδύουμε για τους πολίτες. Κτίρια, δίκτυα θέρμανσης, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τελευταία παρατήρηση όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια εξαρτώμεθα περισσότερο από το φυσικό αέριο. Εισάγουμε 99% των καυσίμων μας των πυρηνικών. Σταματήστε να συνδέετε την πυρηνική ενέργεια από την ανεξαρτησία. είναι γελίο αυτό που υπόθηκε και αυτό που αναφέρθηκε από μια κυρία συνάδελφο. Ο κύριος Μαστάλκα για δυόμιση λεπτά. Κυρίες και κύριοι, κύριε Προεδρεύοντα, Κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση σας, στη θέση της ε, τσεχικής προεδρίας, ούτε ψήλο στον κόρφο σας. Εσείς μιλάτε για Ευρώπη χωρίς σύνορα, χωρίς εμπόδια. Αυτό, αυτό είναι το σύνθημά σας. Μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ποικιλοτρόπως. Νομίζω ότι δεν σημαίνει περισσότερες ελευθερίες για τις αγορές και τους ε, χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς αποτελεί μια πρόκληση για τη βελτίωση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, έτσι ώστε να είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στη άρση των ε, προσκομμάτων των ανετιολόγητων προσκομμάτων, ιδιαίτερα προς την απασχόληση των πολιτών, αλλά και ίση μεταχείριση όλων των πολιτών και των εργαζομένων. Και ελπίζω η Τσεχική Προεδρία να συνεισφέρει στην πρόταση ως προς την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Αν θέλουμε μια Ευρώπη χωρίς σύνορα, και εμπόδια, ας μην δημιουργούμε περισσότερα στον τομέα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η στρατηγική σας προς τις ε, γείτονες χώρες, περιλαμβάνοντας το Κωσυφοπαίδιο και τη Σερβή. Αναφέρομαι και στη Μολδαβία, η οποία έχει επιτελέσει μεγάλες ε, πρόοδους, μεγάλη πρόοδο, Ας μην δημιουργηθούν λοιπόν νέα προσκόμματα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια σαφή πολιτική έναντι της Ρωσίας και της Κίνας και μια εξισορροπημένη πολιτική για τα συμφέροντα της Ευρώπης. Ευρώπη χωρίς προσκόμματα σημαίνει ότι θα πρέπει να σεβαστούμε και τις μειονότητες και ιδιαίτερα για αυτούς που είναι απάτριδες και δεν έχουν άσυλο. Επίσης θα πρέπει να προωθήσουμε νέες ε, πολιτικές για να μην υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά που πολλές φορές εφαρμόζονται. Εσείς είπατε ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία κατά τη λήψη αποφάσεων. Άρα οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να έχουν την ε, δυνατότητα να διενεργήσουν ε, δημοψηφίσματα. Θα ονόματι της ομάδας της ε, ΙΝΤΕΜ να χαιρετήσω με κάθε σεβασμό την Τσεχική Προεδρία. Την χαιρετώ εκφράζοντας και τις απόψεις μας. Λαμβάνουμε υπόψη ότι πέρασε μεγάλη δοκιμασία ο τσεχικός λαός και είναι σε καλύτερη θέση από περισσότερους από εμά να καταλάβει το τίμημα και το νόημα της λέξης ελευθερία. Χαιρετίζω επίση την Προεδρία και που συνοδεύεται ο χαιρετισμό αυτός από τις ελπίδες μας. Κύριε Τοπολάνεκ, κύριε Βάκλαβ Κλάους, ε, εκφράζεται κάποιες ελπίδες μας. Ακούστε τη φωνή των λαών. Ας γίνουν σεβαστά τα δημοψηφίσματα της Δίκης Αβώνας όλη την Ευρώπη. Και δώστε στους λαούς την ελευθερία τους να απελευθερωθούν οι λαοί από την γραφειοκρατία των Βρυξελών που μας βυθίζει. Σήμερα όλο και περισσότεροι οι λαοί της Ευρώπης ε, είναι, θέλουν να απομακρυνθούν από την Ευρώπη, τις Βρυξέλλες. Ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ ένα μόνο πράγμα ε, θέλω να ζητήσω από την Προεδρία. Βοηθήστε μας έτσι ώστε ε, να γίνουν σεβαστοί οι θεσμοί της δημοκρατίας. Όταν έχουμε δημοκρατία αποφασίζει ο λαός. Και ο λαός αποφάσισε στην Ολλανδία, στην Ιρλανδία, στη Γαλλία. Ο λαός ε, αποφάσισε ε, να ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων τη συνθήκη της Λισαβόνας σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία στην έκφραση των απόψεων. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν τίποτα για την μη προσχώρηση άλλων ευρωπαϊκών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί οι τεχνοκράτες επιβάλλουν τη θέλησή τους. Η Τσεχία μόλις πριν από λίγο καιρό αποτείναξε τη δικτατορία. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι πραγματικά έχετε δυνατότητα να αντιμετωπίσετε τη νομενκλατούρα των Βρυξελών και η δική σας χώρα μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Πρωθυπουργέ και το Πολάνεκ, σα καλωσορίζω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι παλέ συζητήσει είναι πολύ σε καλά χέρια η Ευρώπη το επόμενο εξάμεινο. Είναι ιστορική στιγμή για την τσεχική δημοκρατία και θα επιδείξετε τις γνωστές πολιτικές σας επιδεξιότητες. Το πρόγραμμα το τσεχικό θέτει την ενέργεια, την οικονομική βελτίωση και το ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο σαν ε, πρωταρχικέ προτεραιότητε και στι πρώτε μέρε τη Προεδρία σα αντιμετωπίσατε σημαντικέ προκλήσει. Πήγατε Κίεβο, πήγατε Μόσχα και εργάζεστε σκληρά για να πετύχετε μια συμφωνία για να αποκατασταθεί η ροή φυσικού αερίου προ ευρωπαϊκέ χώρε. Επιδείξατε μεγάλε διπλωματικέ δεξιότητε μέχρι τώρα, συνεργασία με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά είναι ζωτική σημασία στη ρωσική κυβέρνηση να καταλάβει ότι να είναι όμοιροι οι χώρε δεν είναι ένα τρόπο για επιχειρήν στο σημερινό κόσμο Υγηθήκατε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι τώρα και σα συγχαίρω γι' αυτό. Επίση, προσπαθώντας να επιλύσετε την κρίση στη Μέση Ανατολή. Να επιφέρετε αξιόπιστη κατάβαση του πυρός που θα οδηγήσει σε συνομιλίες συνευτικές. Καλές προσπάθειες. Η οικονομική κρίση έχει προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας. Προτείνετε λογικά μέτρα για την μετώπιση της οικονομικής υφήσεως. Υπήρχατε σαφείς για τη σημασία που έχουν τα κράτη-μέλη και η Ευρώπη να μην επιβάλλουν ε, επαχθείς κανόνες ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και να κινητοποιηθούν οι χώρε που έχουν παρόμοια φιλελεύθερη οικονομική προσέγγιση για να αντιταχθούν στον προστατευτισμό σε αυτή τη φάση. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να εξασφαλίσουμε ότι οποιαδήποτε ρυθμιστική αλλαγή είναι ανάλογη και λογική. Τέλο, σε μία εβδομάδα θα έχουμε νέο πρόεδρο τον ΗΠΑ στο Λευκό Οίκο. Ξέρω ότι μπορούμε να συστούμε σε εσά, κύριε Πρωθυπουργέ, ώστε να έχετε καλέ σχέσει με τον κλαγέντα πρόεδρο Ομπάμα. Συμμερίζετε την άποψή μου ότι το μέλλον τη διατατική αυτή συμμαχία είναι ζωτική σημασία για την ασφάλειά μα και την ευμάρειά μα. Σα εύχομαι κάθε επιτυχία. Και όπω είπε ο Βίστον Τσέρτσελ στη μεγάλη τελευταία ομιλία του Συμβουλίου των Κοινοτήτων, ποτέ να μην ταράζεσαι, ποτέ μην κουράζεσαι και ποτέ μην απελπίσεσαι. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κύρκοφ. Ο κύριος Βίγγενεν έχει το λόγο για δύο λεπτά. Κύριε Μπαρόζο, κύριε Τοπολάνεκ, αγαπητοί συνάδελφοι, θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Τσεχική Προεδρία είχε μια πολύ δύσκολη αρχή με την χρηματοπιστωτική ε, κρίση, την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας και την παροχή φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δραστηριότητά σας θα είναι ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας και της προεκλογικής εκστρατείας για τις ευρωεκλογές θα έχουμε 532 νέα μέλη και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την συνθήκη της Λισαβόνας. Θα την κυρώσετε ή όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μία από τις προτεραιότητες ε, της ατζέντα σας είναι, είσαστε πολύ κακότυχοι που υγείστε της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια τέτοια κατάσταση, αλλά νομίζω ότι μπορείτε να καταστήσετε την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο αξιόπιστη στη Μέση Ανατολή, να προωθήσετε την ε, παροχή ενέργειας, δηλαδή φυσικού εργείου και να δημιουργήσετε νέες θέσεις εργασίας. Κύριε Τοπολάνεκ, ελπίζω να επιτύχετε. Αφέρετε μια συγκεκριμένη ευθύνη δίνει και φαίνεται έτσι δείχνεται ότι οι νεοφερμένοι μπορούν να ασκήσουν ηγετικό ρόλο. Ελπίζω να ε, μπορέσουν τα 27 κράτη-μέλη να ακολουθήσουν μια ενιαία πολιτική, αλλά αυτό ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ενότητα στην ίδια την τσεχική δημοκρατία που δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Άρα ε, σταματήστε τα εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, διότι η Σλοβενία είναι ένα παράδειγμα που μπορείτε να ακολουθήσετε. Επίσης θα πρέπει να ενώσετε τα βασικά πολιτικά κόμματα και συνασπισμού σε αυτό το κοινοβούλιο και να διευρύνετε το διάλογο. Έχετε πολλά μαθήματα να λάβετε από την γαλλική κυβέρνηση. Επίσης θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον αντισημιτισμό και την ξενοφοβία θα ήθελα να περιλάβετε αυτό το θέμα στην ατζέντα σας, ιδιαίτερα ενώπιον των, ευ... των επόμενων ευρωεκλογών. Η κυρία Βάλεν έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κρατήστε το χρόνο μιλία σας παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου που ήρθε εδώ σήμερα για να παρουσιάσει το πρόγραμμα της Εχικής Προεδρίας, όμως να επιστήσω την προσοχή επί κάποιων θεμάτων που ελπίζω ότι η Προεδρία σας θα μπορέσει να εξετάσει. Πρώτα απ' όλα το σύνθημα που επιλέξατε είναι Ευρώπη χωρίς φραγμούς. Συμφωνώ με το πνεύμα αυτού του συνθήματος και θα πρέπει να αληθεύει για τους Ευρωπαίους πολίτες κυρίως που έχουν το δικαίωμα να μετακινούνται και να κατοικούν οπουδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι εισηγήτη για την εφαρμογή τη οδηγία για την ελεύθερη μετακίνηση, διακίνηση. Δυστυχώ φαίνεται το σύνθημά σα απειλείται από τι εθνικέ αρχέ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα εξέδωσε μια έκθεση όσον αφορά την εφαρμογή της εν λόγω ε, που είναι άκουσα απογοητευτική. Ακόμα και η σωστή εφαρμογή της οδηγία από τα κράτη-μέλη ε, δεν ξέρω αν θα λύσει το πρόβλημα. Να δώσετε μεγαλύτερο βάρο στο θέμα, ελπίζω, από αυτό που παρουσιάσατε στο πρόγραμμά σα όσον αφορά τον τομέα ελευθερία και ασφάλεια. Δεύτερον, πέρα των σημαντικών θεμάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια τη Προεδρία σα, όπω είναι η συνεχιζόμενη κρηματοπιστωτική κρίση και οι ανησυχίε για τον ασφαλή εφοδιασμό σε ενέργεια, έχετε και πάρα πολύ μεγάλο νομοθετικό βάρο. Οπότε ελπίζω και πιστεύω ότι θα χρησιμοποιήσετε όλα τα αναγκαία μέσα, ώστε να ολοκληρωθούν τα διάφορα, οι διάφορε εκκρεμεί εκθέσει εγκαίρω πριν το τέλο τη κοινοβουλευτική θητεία. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν και δημιουργήθηκαν προσδοκίε για του Ευρωπαίου πολίτε όσον αφορά τη μείωση των τιμών για, την, για το roaming, για τη φωνητική τηλεφωνία και, και ελπίζω να καταλήξετε με την ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση από τα θέματα. Αυτά και καλή επιτυχία για την Προεδρία σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος για ένα λεπτό. Λοιπόν, ε, ε, Ελπίζω από τα άχρηστα λόγια των Βρυξελών να περάσει στις πράξεις η Ευρώπη μέσω της ε, τσεχικής δημοκρατίας και από το σωματεμπόριο κλπ. να λύσει τα προβλήματα και με τους παρανόμους μετανάστες. Λοιπόν, σε πρόσφατη η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιταλία και η Μάλτα, ο Υπουργό ο κύριος Μαρόνι ε, είπε ότι η Ευρώπη πρέπει να επαγρυπνεί και θα πρέπει να λάβει υπόψη που σοβαρή είναι η κατάσταση στη Μεσόγειο όσον αφορά την παράνομη με τα εμπόριο ε, ναρκωτικών από την Ασία και είναι απαραίτητο να ληφθούν ειδικά μέτρα και θα πρέπει οι Υπουργοί Εσωτερικών να συνάψουν συμφωνίες με τις χώρες προέλευση για την επανεισδοχή των παρανόμων μεταναστών. Θα πρέπει να ενισχυθεί η δράση του Frontex, που θα πρέπει να είναι συντονισμένη η δράση με τα κατάλληλα μέσα και θα πρέπει να καταλάβει η Ευρώπη ότι θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν υπάρχουν συμφωνίες επανεισδοχής των παρανόμων μεταναστών με χώρες άλλε. Και ειδικά οι χώρε πρέπει να, όπω οι δικοί μου, να λάβουν μέτρα. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Λαμπετούσα, αν δείτε πόσο σοβαρό είναι το πρόβλημα. Και, θα, και το κέντρο της καταπολέμησης το εμπορίου ναρκωτικών στη Μεσόγειο ε, θα πρέπει να κάτι να γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, είναι καλύτερο νησί της Μεσογείου η Λαμπεντούσα και έχει προβλήματα παράμονους μετανάστες. Τσεκ για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε κύριε Πρόεδρε και για την παρέμβαση αυτή από πλευράς του κυρίου Τοπολάνεκα και της Τσεχικής Προεδρίας και σε σχέση με την εκλογή στην Ευρωβουλή χαίρομαι για το ότι η Τσεχία θα έχει την Προεδρία του Συμβουλίου τους επόμενους έξι μήνες. Εδώ και πάνω από 40 χρόνια υπό την κατοχή της Τσεχίας, της Τσεχοσλοβακίας είχα πάει στη Γερμανία και είναι θαύμα το ότι στην Τσεχία και στην κεντρική Ευρώπη ζούμε σήμερα σε ελευθερία και μπορούμε να, μπορέσαμε να οικοδομήσουμε τη δημοκρατία και να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η σημερινή πολιτική, οικονομική και οικολογική ανάπτυξη για κάθε προεδρία του Συμβουλίου θα σήμαινε μια μεγάλη πρόκληση, ούτως ή άλλως. Αυτό πιστεύω θα είναι κάτι που θα μπορέσει να ξεπεράσει η Τσεχική Προεδρία ω πρόκληση. Εύχομαι στην Τσεχία αλλά και σε εμά ό,τι καλύτερο για αυτή την Προεδρία. Ευχαριστώ. Στο χρόνο. Ο κύριο Αδάμου για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε τη Επιτροπή, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, στις προτεραιότητες τη υφιστάμενη Προεδρία σα βρίσκεται και το εξή. Για να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλαμβάνει διεθνή δράση, χρειάζεται να προσδέσει την ασφάλεια τη σε μια στρατηγική συνεργασία με το νατο και να αναπτύξει δικέ τη αμυντικέ δυνατότητε συμπληρωματικέ του νατο. οι πολίτε διαρωτούνται από ποιου απειλείται η ευρωπαϊκή ένωση ώστε να χρειάζεται να προσθέσει την ασφάλεια τη στο νατο. αντίθετα μια ορατή απειλή για την ευρωπαϊκή ένωση είναι η στρατηγική που ακολουθεί το ισραήλ στρατηγική του πολέμου την οποία η ευρωπαϊκή ένωση δεν καταδικάζει ξεκάθαρα και δεν επιβάλλει κυρώσει πράγμα που κάνει για άλλε περιπτώσει. περαιτέρω δηλώνεται ότι θέλετε μια οικονομία χωρί σύνορα και ότι θα πρέπει να αποφευθεί η υπερβολική ρύθμιση να αποφευθεί η αύξηση στο επίπεδο του προστατευτισμού. αυτά είναι τα μαθήματα που παίρνουμε σαν ευρωπαϊκή ένωση από την οικονομική κρίση. η μη προστασία των αδυνάτων και η κερδοσκοπία της αγοράς δεν είναι παράξενο επομένω που οι πολίτε δυσανασχετούν με τι πολιτικέ τη ευρωπαϊκή ένωση. το δείχνει και το ευρωβαρόμετρο το οποίο ποτέ δεν λαμβάνουμε υπόψη εκείνο που είναι επίκαιρο σήμερα και το οποίο αναδεικνύουν οι μαζικέ διαδηλώσει είναι η ανάγκη για πολιτική ειρήνη και όχι συνένοχη ουδετερότητα. οι αντιδράσει και η λαϊκή διαμαρτυρία αποτελούν κραβαλαία απόδειξη τη ανάγκη για δικαιοσύνη και για πολιτική ελέγχου τη αγορά και των τιμών των αγαθών που να επιτρέπει σε έκαστο κράτο να αναλαμβάνει τον κοινωνικό ρόλο που οι πολίτε του αναθέτουν χωρί του δογματικού περιορισμού του Συμφώνου της Σταθερότητας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Δάμ, και εσείς είστε συνεπείς στο χρόνο. Η κυρία Σίνωτ για ένα λεπτό. Mr. President, um, I'd like to welcome... Κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω, εύχομαι ότι το καλύτερο για την Προεδρία σας. Ως Ιρλανδί θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση και το λαό σας. Οι δικοί μου πολίτες κατεψήφισαν τη συνθήκη Λισαβόνα σε δημοψήφισμα και μόνο οι Τσέχοι είπαν ότι θα σεβαστούν την απόφαση αυτή των Ιρλανδών. Ενώ βέβαια οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί που είχαν επίσης καταψηφίσει δεν έχουν το δικαίωμα αυτή τη φορά να εκφραστούν. Είναι απαραίτητος τέτοιος σεβασμός γιατί στην Ευρώπη έχουμε αντιμετωπίσει πολλές κρίσεις και χρειάζεται μία αντιμετώπιση που θα συμπεριλαμβάνει απαραίτητος και το σεβασμό των λαών των χωρών μελών αν θέλουμε να πετύχει. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το σεβασμό που επέδειξατε κι εσείς και ο λαός σας και φαίνεται πιθανό και οι Τσέχοι να απορρίψουν τη συνθήκη της Λισαβόνας. κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ίσως εσείς κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, κύριε Τοπολάνεκ, ίσως με τέτοια χαρμόσυνη υποδοχή δεν υπολογίζατε στην Ευρωβουλή. Όμως η Τσεχική Προεδρία του Συμβουλίου είναι ένα μεγάλο γεγονός. Γεγονός θα ήθελα να πω με μια πνοή ιστορική σημασία. Στην πολιτική μου ζωή δύο κυριότερα πολιτικά γεγονότα έζησα. Πρώτον την επανένωση της Γερμανίας, αφετέρου την Ευρωπαϊκή Επανένωση μετά από δύο αιματηρούς εμφύλιους ευρωπαϊκούς πολέμους τον προηγούμενο αιώνα και το ότι σήμερα η Τσεχία έχει την Προεδρία ε, ε, στο Συμβούλιο και την εκπροσωπή εδώ είναι απόδειξη αυτών των ιστορικών σημαντικών αλλαγών και είμαστε ευγνώμονε σε εσά. Σίγουρα θα έχετε την υποστήριξη τη ομάδα ΕΛΚΕΔ χωρί επιφύλαξη και χωρί όρου και προποθέσει και επιφυλάξει. Σωστά και δίκαια αναφέρατε το εύρο αυτό το ιστορικό με τον Κάρολο τον Τέταρτο που ξεκινάει έναν από του πρώτου ε, Ευρωπαίου αρχιτέκτονε του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών αλλά και έναν από του ιδρυτέ των αρχαιότερων Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Και έτσι εκπρόσωπο ενός παγκοσμίου πνεύματος από την Ευρώπη που εμάς τους Ευρωπαίους ε, με τον ίδιο τρόπο μας χαρακτηρίζει ε, ίσως όπως και οι ίδιες οι συνθήκες που συνάψαμε. Θα βρείτε την αποδοχή από πλευράς μας πέρα από την ε, μία ή άλλη ευρωσκεπτιστική ευρωεπιφύλαξη που εκφράζεται από τη χώρα σας. Υπάρχουν πεπισμένοι Ευρωπαίοι, αλλά για όλους αυτούς τους λόγους ακριβώς είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε λαθασμένες εξελίξεις ε, και πορείες και να συνεισφέρουμε να επανορθωθούν, να διορθωθούν. Και για την ε, διόρθωση τέτοιων ε, ολιστημάτων η συνθήκη της Λισαβόνας είναι ένα εξαιρετικό μέσο, εργαλείο που θα έχουμε στα χέρια μας. Και αναμένουμε και προσδοκούμε εσείς ως Προεδρεύων του Συμβουλίου να συνεισφέρετε, να αρχίσει να ισχύει αυτή η συνθήκη. Να μπορέσετε να συνεισφέρετε ώστε η χώρα σας να επικυρώσει αυτή τη συνθήκη το δυνατόν γοργότερα. Για 1,5 λεπτό κύριος Μπαρόν Κρέσπο Σα Ευχαριστώ Σας ευχαριστώ. Στα ελληνικά, ο κύριος Κρέσπο. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω την Τσεχική Προεδρία με την ίδια φιλία και πνεύμα φιλίας ε, όπω ω πρόεδρο ε, του Κοινοβουλίου είχα απευθυνθεί στο παρελθόν το 1991 προ του τσέχου για να του προσκαλέσω να ενωθούν ε, με του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Αυτή η μεγάλη γενεά εκείνων των Τσέχων, Τσεχοσλοβάκων εκείνης της εποχής ενσαρκώνεται σε μια μεγάλη προσωπικότητα στον κόσμο και στην Τσεχία. Αναφέρομαι στον πρόεδρο Βάσλαβ Χάβελ. Δύο σκέψεις και ερωτήσεις προς τον Προεδρεύοντα. Εσείς λάβατε μια απόφαση και χαίρομαι για το ότι γίνεται λόγος για την Ευρώπη των κανόνων και αποφασίσατε να εντάξετε την κύρωση της συνθήκης της ε, Λισαβόνας με την επικύρωση του, της αντιπυραυλικής ε, ασπίδας. Εσείς λάβατε ούτως ή άλλως μία απόφαση να εντάξετε την ίδια τη χώρα σας, ε, κάτι που πρέπει να εξεταστεί από κοινού λοιπόν δεν πρέπει να γνωρίσουμε ένα γεγονός και αυτό είναι ότι η σύραξη για το φυσικό αέριο είναι πολιτική σύραξη. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει πολιτική προς, προς την Ανατολική Συνιστόσα υπό αυτούς τους όρους και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όντας η Τσεχία ένας λαός υπερήφανος για την ανεξαρτησία του, γιατί υποτάσσετε και εντάσσετε εσείς αυτό το οποίο ε, θα πρέπει να αποφασίσουν οι Τσέχοι στην απόφαση των Ιρλανδών. Κατά δεύτερο λόγο, κύριε Προεδρεύοντα, μιλήσατε για το ευρώ. Χθε είχαμε εδώ την ε, εορταστική εκδήλωση για την δεκαετία του ευρώ και την ένταξη της Σλοβακίας στη ζώνη ευρώ. Τι θα κάνετε για την προστασία του ευρώ υπό την Τσεχική Προεδρία. Ερώτημα. Ευχαριστώ. Κλείνα, το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Τοπολάνο και κύριε Μπαρόζο, θα ήθελα Κύριε Πρόεδρε, να αναφερθώ ω εξή. Βρισκόμαστε σε δύο κρίσει. Μία κρίση κλίματο και μία χρηματοοικονομική κρίση. Και τώρα προστίθεται η ενεργειακή κρίση επιπλέον. Γι' αυτό είναι σημαντικό να επικεντρωνόμαστε στα ουσιοδέστερα. Κύριε Τοπολάνεκ τώρα, η Τσεχία θα μεριμνήσει, θα ενδιαφερθεί ώστε τα προγράμματα για την ανάκαμψη τη οικονομία θα μπορέσουν να λειτουργήσουν ώστε να επιληθούν τα προβλήματα τη κλιματική κρίση. Θέλουμε τους πολίτες μας να του οδηγήσουμε για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά από μια οικονομική κρίση πρέπει να αλλάξει και η πορεία που ακολουθείται και ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα θέματα. Να έχουμε ενεργειακά σπίτια συλλογής ε, ε, ηλιακής ενέργειας. Γι' αυτό πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις για τις κλιματικές αλλαγές, ώστε να δημιουργήσουμε τον ιστό εκείνο που χρειάζεται η Ευρώπη. Ενεργειακά φιλικές τεχνολογίες που θα εξοικονομούν ενέργεια. Μόνο έτσι μπορούμε να κάνουμε κάτι κατά των Ρώσων και της σημερινής πολιτικής. Εκείνοι που ήταν κατά του ενεργειακού πακέτου θα κατανοήσουν. Γιατί καταβάλαμε τέτοιες μεγάλες προσπάθειες για να μιλάει η Ευρώπη με μια φωνή που θα αρθρώνει ενωμένη οι πολίτες της Ευρώπης ε, θα κατανοήσουν σίγουρα και κατανοούν ποιο είναι το διακύβευμα. Δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκή ολοκλήρωση όταν ο ένας δρά κατά του άλλου και υπάρχουν ε, ε παρεκκλίνουσες ε, κατευθύνσεις και πορείες. Κατά τη διάρκεια της τσεχικής προεδρίας ελπίζω ότι θα υπάρξει καλή συνεργασία και αυτό θα είναι θετικό και για την επόμενη προεδρία του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ότι το κομμουνιστικό καθεστώς θα ήθελα να συγχαρώ την ε, την ε, τσεχική ε, προεδρία ε, γιατί αντιμετωπίζει τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει η αρχική πολιτική. Ωστόσο οι ευρωπαίοι πολιτικοί επηρεάζονται από την πραγματική πολιτική και επηρεάζονται και δεν μπορούν να τα δουν όλα αυτά. Δυστυχώς από τη στιγμή που τα εγκλήματα του ναζί κατά καταδικάζονται ως ε, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αλλά τα σοβιετικά εγκλήματα τα οποία διέπραξε το κομμουνιστικό καθεστώς δικαιολογούνται. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι διχασμένη μεταξύ Ανατολή και Δύσης, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του φυσικού αερίου και όσο αυτό συνεχίζεται οι ευρωπαϊκέ αρχέ δεν θα είναι ολοκληρωμένες και η Ευρώπη θα είναι διχασμένη. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για την πρώτη προεδρία μιας, ε, πρώην, ε, μιας χώρας του πρώην Σοβιετικού Μπλόκου και πραγματικά ευχόμαστε να επιτύχετε. Ξεκινήσατε την προεδρία σας σε πολύ θερμό πολιτικό κλίμα και με τους παγωμένους ανέμους της ενεργειακής κρίσης. Θα ήθελα να σας συγχαρώ κύριε Τοπολάνεκ για την ταχεία σας δράση και για την εξέβρεση λύσης στην κρίση του φυσικού αερίου καθώς και για τη διαμεσολάβηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Δύο βασικές προτεραιότητες, η ενέργεια και η ανατολική εταιρική σχέση. Αυτά χρειάζονται την παροχή φυσικού αερίου και αυτά ε, στο σταυροδρόμι ε, της δικής σας Προεδρίας. Θα πρέπει να βρείτε επίγουσα λύση αλληλεγγύης ε, τώρα θα πρέπει να δουλέψετε στην απεμπλοκή των, ε, της παροχής φυσικού αερίου που κάνει να υποφέρουν 18 κράτη-μέλη, πολίτες και επιχειρήσεις. Και έπειτα θα πρέπει να βρείτε μια διαρκή λύση μόνιμη ε, και σταθερή για το μέλλον. Χρειάζεται μια μακροπρόθεσμη πολιτική που θα πρέπει εσείς να τη σχεδιάσετε. Επίσης καλωσορίζω την προτεραιότητά σας για την ανατολική συνεργασία που θα μας δώσει ένα επαρκές πλαίσιο για καλύτερη συνεργασία με τους ε, ε, έρους μας ε, στα σύνορά μας. Θα το συμπληρώσουμε αυτό με τη δημιουργία της Euronest, ε, μιας διακοινοβουλευτικής συνέλευσης. Είμαι πεπισμένο ότι η Τσεχική Προεδρία που αντιμετωπίζει τόσο μεγάλες προκλήσεις και είναι αναγκασμένη να διαχειριστεί τόσες κρίσεις θα ανταποκριθεί στι προσδοκίες μας και σε λίγους μήνες θα έχουμε λιγότερους φραγμούς και μια ισχυρότερη και ε, ασφαλέστερη Ευρώπη. Και όπως λέτε και στο σλόγγαν σας, ε, η Ευρώπη θα είναι πιο γλυκιά και πιο ήρεμη. Ο κύριος Λάνεν, κύριε Προεδρεύοντα το Πολάνα και η Ευρώπη χωρίς φραγμούς ε, είναι καλό σύνθημα, διότι αφορά τον πυρήνα της ευρωπαϊκής ε, ιδέας ε, και ιδανικού να ενωθούν οι άνθρωποι. Ελπίζω όμως ότι οι φραγμοί θα εξαφανιστούν από τους εγκεφάλους και την οτροπία που με πολιτικά και με πολιτικές και ιδεολογικές επιφυλάξεις εναντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγούν σε αυτοτροχοπαίδηση για την περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως προβλέπεται και σε σχέση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πρέπει πολλή δουλειά να γίνει από τη χώρα σας. Η μεταρρυθμιστική συνθήκη πρέπει να περάσει. Πώς θα κάνουμε ενεργειακή πολιτική χωρί τα θεμέλια της συνθήκης της Λισαβόνας που προβλέπονται για κάτι τέτοιο. Δεν είναι εφικτό κάτι τέτοιο και για πολλέ άλλε πολιτικέ έτσι μπορεί να αντιμετωπίσει κανεί τα πράγματα. Είναι απόλυτα παράδεκτο η επικύρωση να εξαρτάται από άλλα εσωτερική πολιτική υφή προβλήματα. Είναι απαράδεκτο αυτό επειδή πρόκειται για μια κοινή συνθήκη και όχι για εσωτερικέ πολιτικέ αντιπαραθέσει, αντιπολίτευση κατά τη κυβέρνηση ή αντίστροφα. Η Ευρώπη είναι μια ενότητα αξιών. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου βρίσκονται στο επίκεντρο. Και στη χώρα σα υπάρχουν σχετικά ε, ελλείψεις, ελλείμματα. Και ίσως θα ήθελα να δραχτώ της ευκαιρίας να αναφέρω την περίπτωση που εδώ και 14 χρόνια αγωνίζεται για την αποζημίωση η ομάδα. Θα ήθελα να ε, μεριμνήσει η Προεδρία σας για το αίτημα αυτό που είχε κάνει στο παρελθόν ο Βάτσλαφ Χάβελ απεργία πείνα. Ο Σαρκοζή είπε ότι έξι μήνε ε, τη Προεδρία του τον άλλαξαν ω άνθρωπο. Ελπίζω ότι και σε εσά ε, θα ισχύσει το ίδιο. Μέσω αυτή τη πείρα θα μπορέσετε να αλλάξετε και εσεί ε, και η Τσεχική Δημοκρατία. Ευχαριστώ. Micro, please. Prime Minister. Κύριε Πρωθυπουργέ, τέσσερις ερωτήσεις. Εάν δείτε ότι η συνθήκη της Λισαβόνας η συνθήκη της νίκης μάλλον καλύτερα προηγουμένως. Δεν σας ικανοποιούσε γιατί την υπογράψατε. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι η τσεχική δημοκρατία δεν θα μπει στον πειρασμό να ακολουθήσει τους Ιρλανδούς και δεν θα προσπαθήσει να διαρρήξει το πακέτο της Λισαβόνας. Τρίτον, δεν βλέπετε να υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο ότι έρχεστε εδώ και επενείτε την νομιμότητα του Κοινοβουλίου ενώ αρνείστε να υποστηρίξετε τη συνθήκη που αυξάνει τις εξουσίες του. Και τέταρτον, η Τεχική Προεδρία μπορεί πραγματικά να έχει μπορεί πραγματικά να έχει κύρος μέχρι ότου η τσεχική δημοκρατία να επικυρώσει τη συνθήκη. Για ένα λεπτό Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, είναι παράδοξο ότι αυτή η κρίση που έπληξε όλο τον κόσμο αλλά και την Ευρώπη μπορεί για σας να είναι ένας σύμμαχος διότι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να δίνουν κάποια διδάγματα. Εσείς είσαστε οι υπεύθυνοι για το ότι καταλήξαμε σε αυτή την κρίση. Εσείς, ε, ε, ε, αυτοί οδήγησαν σε αυτή την κρίση. Βλέπουμε σήμερα ένα πνεύμα στον λόγο που εκφωνήσατε και ελπίζουμε και ευχόμαστε στην Τσεχική Προεδρία κάθε επιτυχία. Από την ιστορία θα ήθελα να υπενθυμίσω ένα γεγονός σε εσά που πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Το 1618 στο Μπουργ, στο κάστρο της Πράγας υπήρξε ένα μήνυμα το οποίο απεστάλλει και ήταν ιδιαίτερα λαζονικό και οι Τσέχοι αντιστάθηκαν είχαμε την εκπαραθύρωση τότε της Πράγας. Γι' αυτό σας παρακαλώ να εκπαραθυρώσετε μέσω της λογικής και του ορθού λόγου όλους τους συμβούλους που σας τροχοπεδούν και να προχωρήσετε προς τα εμπρός για να επιτευχθεί πρόοδος. Αυτό θα ε, ικανοποιήσει τους πολίτες της Ευρώπης. Να μην ακούσετε τους πλάνους που σας συμβουλεύουν. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ανέκαθεν στην Ευρώπη ζούμε πολύ σημαντικές ιστορικές στιγμές και το εξάμεινο της τσεχικής προεδρίας σίγουρα θα είναι ανάμεσα σε αυτές τις ιστορικές στιγμές. Τα προβλήματα επιτάπητος τα οποία θα πρέπει να βρει λύσεις η προεδρία είναι πολλαπλά και κέρια. Συνθήκη Λισαβόνας που χρειάζεται να εγκριθεί οριστικά. ώστε να μην ε, παραταθεί πέρα από την, ε, το τρέχον έτος ε, η διαδικασία της επικύρωσης. Η τρέχουσα οικονομική κρίση θα έχει επιπτώσεις που θα φανούν μέσα στη διάρκεια του επόμενου έτους. Και έπειτα, η Γαλλική Προεδρία έχει στρώσει το δρόμο ώστε οι επόμενες προεδρίες να πετύχουν ε, ε, αποτελέσματα θετικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα της ενεργειακής κρίσης, πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Το θέμα με περίπλοκη λύση. Ωστόσο, φαίνεται να έχει εξευρεθεί μια λύση. Θα πρέπει ωστόσο να διαβεβαιώσουμε και να διασφαλίσουμε το μέλλον ε, του ανεφοδιασμού σε φυσικό αέριο ε, για το μέλλον, για πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και, η και το δικό μου. Θα πρέπει ωστόσο να σταματήσουν, ε, για τη λωρίδα της Γάζας, άλλο πολύ σοβαρό θέμα, θα πρέπει να σταματήσουν ε, οι βολές ρουκετών και να τεθεί τέλος σε, αυτήν, σε αυτόν τον παράλογο πόλεμο. Έπειτα, θα πρέπει επίσης να προσέξουμε πολύ την κατάσταση κρατών όπως η Μάλτα ε, σε σχέση με την μετανάστευση. Το πρόβλημα της Κύπρου θα πρέπει να επίσης να αντιμετωπιστεί για να λυθεί μια και η σχέση μεταξύ Ευρω... Ελλάδας και Τουρκίας, Ευρώπης και Τουρκίας που περιμένει ε, εντωμεταξύ στην πόρτα για να προσχωρήσει στην Ένωση. Τέλος, Πρόεδρε Τοπολάνευ, ε, περιμένουμε να σας βλέπουμε πάντοτε παρόντα σε αυτή την αίθουσα και σας εύχομαι καλή δουλειά. και σας συγχαίρω για τη δική σας πρώτη εισήγηση. Δεν είμαστε πολύ συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους εισηγήσει. Για λεπτό παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ανακάλυψα στους τσέχους ιστορικούς του λόγους για τους οποίους δεν επικυρώσατε τη συνθήκη της Λισαβόνας διότι μιλούν για την, ε, το μαγικό χαρακτήρα του αριθμού 8, όπως το 2008. Αυτό έχει σημαδέψει την ιστορία σας. Ε, 1918 δημιουργείται η και κτλ. λοιπά ε, Και τρία τελευταία οδυνηρά στοιχεία. 1938 που η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία σας εγκαταλείπουν. 1948 όπου πάτε από την άλλη μεριά μέσω πραξικοπήματος και έπειτα 1968 τα σοβιετικά άρματα. 2008 το καταλαβαίνω, τα αφήσατε να περάσει. Ε, γιατί πιστεύατε ότι το να επικυρώσετε τη συνθήκη εκείνη το χρόνο μπορεί να ήταν ε, ε, ύποπτο ή κακό ε, Επιπλέον ακούσαμε σε διάφορα στόματα τη σύγκριση ανάμεσα στις περιορισμένες κυριαρχίες του Μπρέσνιεφ και της συνθήκης. Ο σύντροφος Μπαρόζο που είναι εδώ, παρά όλα τα ελαττώματά του, δεν είναι ο και παρά το παρελθόν του. Βρισκόμαστε σε μια ε, ε, δομή με μοιρασμένη κυριαρχία που ελεύθερα έχουμε φτιάξει. Και η συνθήκη της Λισαβόνας είναι μόνο μια φάση σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και σας συγκετεύω το 2008 τέλειωσε. Επικυρώστε μέσα το 2009. Το πολύ. Τώρα το λόγο έχει η κυρία Σταρκεβιτσιούτε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ η τσεχική δημοκρατία αναλαμβάνει τη σκητάλη της Προεδρίας μέσα σε συζητήσεις για μεταρρυθμίσεις και την επιλογή του προτύπου που θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Περισσότερο κοινωνικό ή περισσότερο φιλελεύθερο πρότυπο. Καμιά φορά παρουσιάζονται αυτά ως μια συζήτηση μεταξύ της παλαιάς γυραιάς Ευρώπης και της νέας Ευρώπης. Πιστεύω ότι η τσεχική δημοκρατία θα βρει συνενετική πορεία. Αυτές οι δύο έννοιες δεν είναι τόσο αντιφατικές και αντίθετες μεταξύ τους. Οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση και στην πολυπολιτισμική οικονομική κατάσταση η κατάσταση. Ο ορισμός της οικονομίας της αγοράς διαφορετική ερμηνεία την χάνει από διαφορετικούς ανθρώπους. Είναι και εδώ το θέμα των διαφορετικών συμπεριφορών. Έχουμε και το θέμα του πρώην μπλοκ, του Σοβιτικού μπλοκ. Ε, η θέσπιση νόμων αποκλειστικά δεν ε, διασφαλίζει την λειτουργία των αγορών με ικανοποιητικό τρόπο. Θα πρέπει να, κάνουμε, να καταστήσουμε κατανοητές ε, τις ανάγκες των πολιτών και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους. Καμιά φορά για πολιτικούς λόγους αυτά τα πολιτικά πρότυπα πρέπει να υπογραμμίζονται. Όμως σε μακροπρόθεσμη πολιτική προοπτική οι μεταρρυθμίσεις της οικονομίας της αγοράς λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές ε, του οικονομικού περίγυρου δημιουργούν μια δυνατότητα για ριζοσπαστική και λαϊκίστικη δράση ομάδων που προσπαθούν να αποκτήσουν την εξουσία. Και παραπάνω ακόμα, δημιουργούν πολιτική αστάθεια, πολλές φορές και οδηγούν σε τροχοπέδηση. Προχωρούμε στον επόμενο μιλητή, ο κύριος Μπρόκ, για δύο λεπτά. Herr Κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα, συνάδελφοι, και εγώ θα ήθελα στην Τσεχική Προεδρία να εκφράσω συγχαρητήρια με την έναρξη αυτού του αξιώματος της Προεδρίας. Είναι η πρώτη Προεδρία ενός κράτους πρώην μέλους του Συμφώνου της Βαρσοβίας και επιπλέον πρόσθετα σε αυτά που σωστά ανέφερε ο κ. Νασάουε νομίζω έχει συμβολική σημασία αυτό το γεγονός. Και εγώ πιστεύω προσωπικά ότι στο θέμα των διαπραγματεύσεων για το φυσικό αέριο και στο θέμα της δραστηριότητας ε, της, ε, του Προεδρεύοντος του Συμβουλίου Σβάρτσενμπεργκ στη Μέση Ανατολή και με πολλά άλλα παραδείγματα βλέπουμε ότι η Τσεχική Προεδρία έχει καλά προετοιμαστεί για τη δουλειά που την αναμένει. Και γι' αυτό θα ήθελα ακριβώς να τονίσω, να υπογραμμίσω κάτι, ότι αυτή η στρατηγική προσέγγιση από κοινού με τα ενεργειακά θέματα για τον ανεφοδιασμό μας έχει μεγάλη σημασία και να καταστήσουμε σαφές ότι με αυτό το παράδειγμα ακριβώς ότι υπάρχουν πολλοί τομείς, πολλές πτυχές όπου δεν είναι δυνατόν τα κράτη-μέλη μόνα τους αποκλειστικά να μεριμνήσουν για τα συμφέροντα των πολιτών τους, αλλά είναι ένα κοινό συμφέρον της Ευρώπης που πρέπει να εκφράζεται. Κύριε Προεδρεύοντα, ο ανεφοδιασμός ε, της, ε, ε, προϊόντα ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτά τα οποία κάνουμε τώρα είναι θέματα συντονισμού και μη υποχρεωτικά, μη δεσμευτικά. Πολλά από εκείνα που πρέπει να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω της δραστηριοποίησης που μας επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας καθίστανται εφικτά. Με τη δυνατότητα δυνατότητα μια ενισχυμένη ενό ενισχυμένου εκδημοκρατισμού με ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη ενδυνάμωση των δικαιωμάτων και αρμοδιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων αντίστοιχα. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορεί κανεί να πει ότι η μετάφραση σε σχέση με τα γερμανικά μπορεί να μην ήταν σωστή όταν ακούστηκε ότι η συνθήκη τη Νίκαια μπορεί λέει να ήταν καλύτερη από τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Νομίζω την γερμανική μετάφραση θα έπρεπε να την διορθώσουμε. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα. Να καταστήσουμε σαφέ ότι έχουμε κοινέ προκλήσει που πρέπει από κοινού να αντιμετωπιστούν. Με όλα αυτά τα σημεία μόνο με τι συνθήκε Λισαβόνα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Στρέλα για δύο λεπτά. Για ενάμιση λεπτό, κυρία Στρέλα. Μιλήσατε για μια Ευρώπη κανόνων. Μιλήσατε μάλιστα πολύ για τους κανόνες γενικά. Μια, ένας από τους κανόνες της δημοκρατίας είναι η πραγματοποίηση των υποσχέσεων. Εσείς είχατε υποσχεθεί ότι θα υπογράψετε τη συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά μέχρι το 2008 δεν το κάνατε. Κακώς. Άρα λοιπόν πότε η Δημοκρατία της Τσεχίας θα επικυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Εσείς επίσης μιλήσατε για εμπιστοσύνη στον εαυτό σας και για να μην πω για υπεροψία. Ε, η τσεχική κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά δεν μπορεί να ξεχνά ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι αυτή τη στιγμή μιλά στο όνομα γύρω των 450 εκατομμυρίων πολιτών και των 27 κρατών μελών. 25 ε, ε, κράτη-μέλη ήδη επικύρωσαν ε, τη συνθήκη της Λισαβόνας και η Ιρλανδία ήδη προβλέπει δεύτερο δημοψήφισμα. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν την πλειοψηφία στο ναι. Οι Ιρλανδοί κατάλαβαν ότι σε αυτή την διεθνή συγκυρία, η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολη, το να ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζώνη του ευρώ τους προστατεύει από χειρότερες ακόμη καταστάσεις. Ε, τώρα λείπει να μας πει η τσεχική δημοκρατία πότε θα επικυρώσει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Όπως είπε και ο ηγέτης μας ο Μάρτιν Σούλτζ, σε μια στιγμή όπου η Ευρώπη έχει να αντιμετωπίσει άνευ προηγουμένου προκλήσεις, είναι πολύ απαραίτητο να μιλάμε μια φωνή. Και αυτό θα είναι μόνο δυνατόν εφόσον υπογραφεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε ε, Πρόεδρε το μιλήσατε για την ε, ανατολική εταιρική σχέση ανατολική partnership. Ε, τώρα το partnership, αυτή η εταιρική σχέση, είναι μια σχετικά πρόσφατη εφεύρεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπήρχε στην Ευρώπη που ήθελαν οι ιδρυτικοί πατέρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρώπη των πρώτων ετών μετά από τον Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτή η Ευρώπη όμως έδινε στα σύνορά της την προοπτική της προσχώρησης. Ακόμα και στην Ανατολική Ευρώπη. Η Ευρώπη αποτέλεσε έναν παράγοντα ειρήνης όχι γιατί προσέφερε προοπτικέ εταιρικής σχέσης με τους ε, όμορε χώρες αλλά γιατί προσέφερε την προοπτική της συμμετοχή, του μέλους, του membership. Η προηγούμενη προεδρία η Γαλλική που προηγήθηκε τη δική σα ήταν πολύ ξεκάθαρη όσον αφορά τους φραγμούς ε, στο να ορίσει τα σύνορα της Ευρώπη, ε, κλείνοντα τι πόρτες στα μούτρα της Τουρκίας και καθιστώντα σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να κλείσει τα σύνορά της. Το αποτέλεσμα αυτού είναι ότι τα σύνορα της Ευρώπης ε, τις περασμένες δεκαετίες υπήρχε μια ελπίδα για τις χώρες όπως η δική σας. Τώρα σήμερα έχουμε πολέμους και ένταση. Μέση Ανατολή, Βαλκάνια, Κάυκασος, Μαγκρέμπ. Εμείς ως ε, μη βίαιο ριζοσπαστικό κόμμα σα καλώ να λάβετε υπόψη την επίγουσα ανάγκη για οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Ευρώπης που θα είναι ανοιχτά στα μέλη και όχι στις γηχημένες σχέσεις στι partners τη εταιρική σχέση, η οποία αρνείται την ολοκλήρωση αυτό που είναι το πιο σημαντικό δηλαδή των αστικών, των πολιτικών και ε, δικαιωμάτων των πολιτών τη Ευρώπη, αλλά και των πολιτών των όμορων χωρών. Mr. Prime Minister, Κύριε Πρωθυπουργέ, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας συγχαρώ για την ικανότητα που κατέδειξε ήδη η Προεδρία σας σε ένα συγκεκριμένο αριθμό θεμάτων. Και να σας αποκαλύψω επιπλέον ότι για μας τους Σουηδούς εξακολουθούμε να έχουμε την εντύπωση ότι η Πράγα είναι ανατολικά της Στοκχόλμης και λόγω της κληρονομίας της πολιτικής γεωγραφίας του προηγούμενου αιώνα. Λάθος όμως αυτό. Η Προεδρία σας θα επανατοποθετήσει την τσεχική δημοκρατία στην σωστή θέση των χαρτών στην οτροπία μας και στους εγκεφάλους μας, στην καρδιά της Ευρώπης και στην ίδια την ιστορία και ως προς το μέλλον. Επίσης ελπίζω ότι θα προλιαθεί το έδαφος για τη Σουηδική Προεδρία που θα ακολουθήσει όσον αφορά θέματα κλιματικά, και τα θέματα που θα είναι τόσο σημαντικά ώστε να μπορέσει να καταδειχθεί ότι τα οικονομικά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ανοιχτό πνεύμα, χωρί προστατευτικό χαρακτήρα και προστατευτισμό και με τη δυναμική μια ανοιχτή οικονομία αγορά. Και φυσικά λαμβάνοντα υπόψη τα ενεργειακά θέματα επίση το ίδιο. Θα διαδραματίσετε εσεί κέριο ρόλο κέρια σημασία. Είναι προφανέ ότι βρίσκεστε στη σωστή θέση και οι καιροί που αντιμετωπίζουμε υπογραμμίζουν την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Και είναι νομίζω σωστό να πει κανείς ότι η αλληλεγγύη η αλληλεγγύη, η ασφάλεια όσον αφορά τα θέματα ανεφοδιασμού με ενεργειακά προϊόντα σημαίνουν ότι πρέπει να μεταρρυθμίσουμε και να εμβαθύνουμε την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας. Χωρίς αυτό το στοιχείο θα είμαστε πάντα εκτεθειμένοι σε διαφορετικά διαφορετικές προσπάθειες να κατακαιρματιστούμε και να χωριστούμε. Ένα στόχο είναι να διασφαλίσουμε τα πράγματα. Κανεί όμω δεν θα μπορέσει να ελέγξει την παροχή και την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια και φυσικού αερίου, όπω ταυτόχρονα και την διανομή του. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μία ενιαία κοινή αγορά. Και αν αυτό μπορεί να επιτευχθεί κατά την Προεδρία σα, αυτό θα είναι ένα στρατηγική σημασία βήμα προ τα εμπρό. Και νομίζω ότι όλοι θα μπορούμε να σα συγχαρούμε για αυτού του έξι μήνε που θα στεφθούν με αυτή την επιτυχία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε <clears throat> κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Αποκινούμε διάφορους συναδέλφους που βρίσκονται στην αίθουσα σήμερα και εγώ πριν από το 2004 ανήκα σε εκείνους τους ευρωβουλευτές, εκείνους βουλευτές που με ιδιαίτερο τρόπο ήταν υπέρ της ένταξης της ε, Τσεχίας ε, στην μεικτή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία. Και γι' αυτό σήμερα και για τους μη Τσέχους ε, βουλευτές είναι μια ιδιαίτερη ημέρα με ιδιαίτερη σημασία. Μπορούμε να χαιρετήσουμε εμεί από κοινού την Τσεχική Προεδρία και ω Αυστριακή Ευρωβουλευτή να μπορώ να πω ότι δεν ήταν πάντα δημοφιλέ στην Αυστρία να εκφράζεται κανεί υπέρ τη ένταξη και προσχώρηση τη Αυστρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανήκουμε σίγουρα λοιπόν εμεί εκείνου που όσον αφορά την Τσεχική Προεδρία θέλουμε να προσφέρουμε ειδική υποστήριξη και συνεισφορά. Και τι πρώτε αρχικέ δυσκολίε δεν πρέπει να τι υπερτιμήσουμε και να μην υπερβάλλουμε. Και αναφέρθηκε κιόλας και για την μονομερή τοποθέτηση που υπήρξε για την σύραξη στη Γάζα και σε σχέση με τον πρόεδρο που ουσιαστικά σε υψηλέ ε, προδιαγραφές όσον αφορά τα διάφορα θέματα θα πρέπει να οδηγήσει σε μια κατανόηση όσον αφορά την, τον ρόλο της Σλοβακία που αποφασίζει να επαναλειτουργήσει τον πυρηνικό σταθμό του Μποχουνίτσε και που σίγουρα αυτό θέτει κάποια προβλήματα. Εδώ όσον αφορά τον ε, φιλόσοφο Ιέσικ Ρούζα υπάρχει εδώ ιδιαίτερη συνιστόσα για την Τσεχία. Μπορώ εδώ για τους συναδέλφους να συστήσω αυτό το ε, χωριστικό κείμενο να το διαβάσετε, να το απολαύσετε. Δεν υπάρχει οδηγία, δεν υπάρχουν οδηγίες χρήσης για την Ευρώπη. Αν υπάρξουν ποτέ κάποτε, τότε κάθε νέα Προεδρία καλό θα ήταν προσφορά συνεργασίας που γίνεται στην Ευρωβουλή ή από κυβερνήσει των γειτονικών κρατών να μην την αποκρούν και να μην την απορρίπτουν. Ευχαριστώ. Και Κάρας για δύο λεπτά. Σεβαστείτε το χρόνο παρακαλώ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Πλησιάζουν στις ψηφοφορίες θα αναγκαστώ να κλείνω το μικρόφωνο όταν τον ξεπερνάτε. Κύριε Κάρα, κυρία Πρόεδρε, κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, έχετε ιδιαίτερη ευθύνη, κύριε Προεδρεύοντα. Η Τσεχική Προεδρία που ξεκίνησε με ανώμαλο τρόπο οδήγησε σε προκλήσει, οδήγησε σε οργή. Όμω η προσπάθεια να βρείτε το σωστό βηματισμό ώστε να εκφράζεται η ευθύνη για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι το οποίο νιώθει κανείς σήμερα μόλι για πρώτη φορά. Η προετοιμασία φαίνεται να είναι καλή. Στο πρόγραμμά σα θέτετε τα σωστά κέντρα βάρου εμείς όμως θα σας κρίνουμε και θα σας αξιολογήσουμε με, ποια, με ποιο σθένος, ποια αποφασιστικότητα, ποια προσπάθεια εκφράζεται αυτή την ενιαία άποψη της Ευρώπης και ποια βήματα γίνονται για να εκφραστεί αυτή. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεώρησε ότι ε, ΕΕ σε αυτό το εξάμεινο θα δοκιμαστεί. Θα δοκιμαστεί είπε. Η Τσεχική Προεδρία και η Τσεχική Κυβέρνηση στα ευρωπαϊκά πολιτικά θέματα βρίσκονται στο δοκιμαστήριο. Θα δοκιμαστούν. Θα ξεπεράσετε αυτή τη δοκιμασία μόνο αν δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Και γι' αυτό παρακαλώ να σταματήσετε την εσωτερική πολιτική στα δικά σας θέματα να την θέτετε κατά των ευρωπαϊκών θεμάτων και να επιβαρύνετε η ευρωπαϊκή πορεία λόγω εσωτερικών αντιπαραθέσεων. Πείτε στους πολίτες σαφώς με κάθε κάθετο τρόπο ότι τώρα νιώθουμε το τι συμβάνει, συμβαίνει και με τη λωρίδα της Γάζας και με τα ενεργειακά θέματα και με τον Πόχου Νίτσε της Σλοβακίας ότι θέλετε πιο ενδυναμωμένα από την πράγμα να δράσετε για να υπάρξει εξισορρόπηση από κοινού με τα άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση αξιών και κράτους δικαίου. Μάλιστα έχουμε κανόνες του παιχνιδιού. Όποιος δεν τηρεί αυτούς τους κανόνες του παιχνιδιού <clears throat> όποιος τις υποσχέσεις δεν τις στηρεί, τότε δεν εκφράζει σωστά την αλληλεγγύη προς την Ευρώπη. Η ενότητα αξιών, η ένωση αυτή υπέ της επίτευξης κοινών στόχων μας ενώνουν, μας συνενώνουν όλους παρά τις διαφορές μας. Γι' αυτό παρακαλώ να μην χρησιμοποιείτε πρόσχημα τις διαφορές της εσωτερικής πολιτικής στη χώρα σας. Να επικυρώσετε τις συνθήκες Λισαβόνας ε, κατά τη διάρκεια του 2009, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας. Θα σας μετρήσουμε με το αποτέλεσμα των πράξεων πράξεών σα και όχι με τι διακηρύξει που κάνατε ω Προεδρεύον. Κύριε Κάρα, ο κύριο Τίτλε για 1,5 λεπτό. Ναι. Δεν φαίνεται στην Νέα Σφαγιός τίτλη. Ο κύριος Ζιελένιτς για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν σας άκουσα. Ε, ο Τσέχος Προεδρεύων είπε ότι η αντιπολίτευση θέλει να τορπιλήσει την τσεχική κυβέρνηση γιατί ε, νομίζω ότι από μόνη της η τσεχική προεδρία κάνει ό,τι μπορεί για να αυτοτορπιλιστεί. Επίσης διαπίστωσε ότι κάνει ό,τι μπορεί να διευρύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και προς την Κροατία. Αφού κάνουν ό,τι μπορούν, γιατί δεν μπορούν να επικυρώνουν τη Λισαβόνα. Αφού η τσεχική προεδρία το έχει συμφωνήσει και ούτως ή άλλως θα πρέπει να τηρήσει την υποχρέωση αυτή. Πρέπει να το ομολογήσουμε ότι δεν είναι και πολύ σπουδαία η αρχή. Η Τσεχική Προεδρία μιλά για ανόητη πολυτέλεια όταν μιλάμε για τη δέσμη των περιβαλλοντικών μέτρων. Μιλά για κομμουνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα αριστούργημα ε, για όλους και ιδιαίτερα για τους Βουλγαρούς και, ε, για τους Βουλγαρούς και, πρέπει αργότερα να αποσύρει την ίδια της τη δήλωση λίγες ώρες μόλις μετά. Ε, τώρα, από τη στιγμή που θα ε, Έχουμε λέει full time προεδρία του Συμβουλίου, ε, τόσο το καλύτερο, γιατί μόνο αυτή η συνεπής δράση θα δώσει καλύτερη Ευρώπη ε, και οικονομική ανάκαμψη. Ας έχουμε λοιπόν κάποια ηγετική δυνατότητα και να συγχαρώ και τον Πρόεδρο Μπαρόζο για τις δικές του ενέργειες. Ο ε, Κυρία Πρόεδρε, η Τσεχική Προεδρία κατέβαλε προσπάθειες να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει η Ευρώπη όσον αφορά το φυσικό αέριο και την κρίση στην Ουκρανία. Έχουμε όμω ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να επιληθεί. Είναι σαφέ αυτό. Αυτό αναφέρεται στι Ευρω... στις ρωσικέ φιλοδοξίε και την επέκταση αυτών των φιλοδοξιών όσον αφορά την εξουσία και επιρροή στην κεντρική Ευρώπη. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε την προσοχή μα στην Ουκρανία μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Διότι δεν είναι δυνατόν η Ουκρανία να εξακολουθεί να έχει αυτέ τι αδιάφανε τιμέ και θα πρέπει να δούμε ότι θα υπάρχει το θέμα εξάρτηση τη Ουκρανίας από τη Ρωσία. Στις προτεραιότητες της ε, Τσεχικής Προεδρία ανήκει ο ασφαλή ανεφοδιασμός ε, με ηλεκτρικό ρεύμα ή με ε, φυσικό αέριο. Η πιο σημαντική πτυχή είναι να βοηθήσουμε την Ουκρανία να εισαγάγει τιμές τη αγορά και σε μακροπρόθεσμε συνθήκε που θα διαπραγματευτούμε να μπορέσει να λυθεί το πρόβλημα. Πρέπει να ασκηθεί πίεση στο Κίεβο η αδιαφανή δομή των της οικονομίας ε, να αποσαφινιστεί, διότι δεν βοηθά αυτό την δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Μόνο έντονη πίεση εκ των έξω προς την Ουκρανία και μια ενεργοποιημένη συνεργασία μπορεί να οδηγήσει να εγκαταλειφθούν ε, τα κοντοπρόθεσμα, τα μειοπικά ε, συμφέροντα και να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Αν η Ουκρανία δεν δημιουργήσει, δεν θέσει εντάξει τα του οίκου της, τότε εμείς ως ΕΕ δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα κατά των Ρώσων που είναι όλο και πιο φιλόδοξοι και όλο και πιο στεναροί και σε συνεργασία με την ΕΕ η Ουκρανία. Αυτή είναι ακριβώ τη χρονική συγκυρία. Πρέπει η συνεργασία αυτή με την Ουκρανία να ενδυναμωθεί. Τώρα που φτάσαμε σε αυτή την κρίση και πρέπει μέσα στο πλαίσιο τη ΕΕ να ασκήσουμε την πίεσή μα ώστε να διαμορφωθούν τα πράγματα όπω πρέπει. Αλλιώ θα χάσουμε το παιχνίδι. Να ότι θα κόβεται πια το μικρόφωνο. Ο κύριο Ντερόσα για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ όπως και όλοι στο Κοινοβούλιο. Εύχομαι ε, καλή επιτυχία στην Τσεχική Προεδρία. Ωστόσο, με ε, εξόργησε το, η, φρικτή σας δήλωση σήμερα το πρωί ότι η Λισαβόνα είναι χειρότερη από την Νίκαια. Αυτό όχι μόνο δεν είναι αληθινό, α, είναι ψευδές, αλλά είναι και... Ε, αποτελεί μια ρήξη. Θα πρέπει ίσω να αποσύρετε το σημερινό σα σχόλιο. Χρειαζόμαστε πιο ενωμένη Ευρώπη, όπω μα την προσφέρει η Λισαβόνα, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία μπορεί να αποτύξουν ολόκληρο τον κόσμο στη σύγκρουση. Η ενεργειακή κρίση, η οικονομική και η χρηματοπιστωτική κρίση και πόλεμη σε πολλέ περιοχέ. Ω Προεδρία πρέπει να μεσολαβήσετε υπέρ και, για την Ευρώπη με βάση κοινέ αρχέ αλληλεγγύη ε, εσωτερικά και εξωτερικά, κοινωνική οικονομία τη αγορά, πολυμέρεια και ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και αυτό σημαίνει τα δικαιώματα ανδρών και γυναικών να μοιράζονται ε, μεταξύ τους τα διάφορα καθήκοντα. Κύριε Πρόεδρε, είστε συντηρητικός και φιλελεύθερος, αλλά ε, θα πρέπει αυτό να το ξεχάσετε τους επόμενους έξι μήνες, γιατί διαφορετικά θα έχετε συνέχεια συγκρούσει με αυτό το κοινοβούλιο. Η Ιρλανδία θα ε, κάνει πιθανότατα δημοψήφισμα για το φθινόπωρο για μια εν μέρη αναθεωρημένη συνθήκη της Λισαβόνας. Εγώ θα δουλέψω υπέρ του ναι. Ε, όμως αν αποτύχει το δημοψήφισμα δεν θα σας ευχαριστήσω ψηφίσουν η πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Διακόπτω το μικρό. Δύο λεπτά τώρα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ τον κύριο Τοπολάνεκ για την ανάληψη της Προεδρίας της Ένωσης και επίσης για την επιτυχία των πρώτων δύο εβδομάδων της Προεδρίας. Κατανοώ αυτά που είπατε για την εθνική ταυτότητα, διότι οι εθνικές ταυτότητες οικοδομήθηκαν με διαφορετικό τρόπο στην Ανατολική από ό,τι στη Δυτική Ευρώπη. Θα ήθελα να αναφέρω τα κύρια θέματα που πρέπει να θυγούν τους επόμενους έξι μήνες. Το είναι η ενεργειακή δέσμη καταρχήν, όπου θέλουμε να δημιουργηθεί μια κοινή αγορά ενεργείας και ένα, μια υπηρεσία για τους συντονισμού των ρυθμιστών και κοινέ επενδύσεις. Αυτό βέβαια σημαίνει ένα πράγμα, αλληλεγγύη. Αλληλεγγύη ως προς τις ενεργειακές προμήθειες. Η ενεργειακή δέσμη σημαίνει επίσης απελευθέρωση. Δίκαιο, ανταγωνισμό και πρόσβαση στα δίκτυα με εγγύηση μιας ανταγωνιστικής αγοράς και αυτό σημαίνει λιγότερη βλάβη για το περιβάλλον και φτηνότερη ενέργεια για τους καταναλωτές άρα και για το σύνολο της οικονομίας για να ξεπεράσουμε την τρέχουσα οικονομική κρίση. Τέλος, η ενεργειακή αυτή δέσμη επίσης σημαίνει συνεργασία με χώρες εκτός της Ένωσης εκείνες που μας προμηθεύουν την ενέργεια, δηλαδή και εκείνες που την μεταφέρουν. Η ανατολική διάσταση επίσης υπάρχει στην ενεργειακή δέσμη άρα. Η διασφάλιση των αναγκών της οικονομίας μας λοιπόν και η ανατολική διάσταση είναι τα δύο βάθρα της πολιτικής αυτής. Σας καλώ λοιπόν να τα σεβαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαιρετίζω την τσεχική προεδρία του Συμβουλίου. Κατά τη διάρκεια αυτής της ε, προεδρίας ε, θα έχουμε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Η ανεργία θα αυξηθεί. Θα έχουμε επίσης και μια οικονομικά πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία. Την προηγούμενη εβδομάδα διάβασα τους Financial Times. Ο πρόεδρος Κλάους της Τσεχίας πρότεινε λέει κάποιες λύσεις με τις οποίες ε, θα μπορούσα να συμφωνήσω. Είπε ότι πρέπει φιλόδοξοι να είμαστε για την κλιματική πολιτική αλλά να προσαρμόσουμε τις ε, ανάγκες μας και τις φιλοδοκίες μας ε, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα. Θα ήταν λάθος όμως να ακολουθήσουμε μια πορεία που να είμαστε λιγότερο φιλόδοξοι. Πρέπει να παίξουμε το χαρτί της σύγχρονης τεχνολογίας των σύγχρονων υποδομών, ώστε να έχουμε μακροπρόθεσμα μια βιώσιμη αηφόρο κοινωνία και μια δραστήρια πολιτική για τα θέματα του κλίματος. Αυτό ισχύει επίσης και για την κοινωνική πολιτική. Κοινωνική πολιτική με δίκαιες ε, συνθήκες ε, και όρους ε, του παιχνιδιού. Ένα ισοδίκαιο πλαίσιο για το παιχνίδι που θα διεξάγεται. Αυτό δεν σημαίνει λιγότερη ανάπτυξη, σημαίνει αηφόρο ανάπτυξη σε πιο μακροπρόθεσμη κλίμακα. Και για την πολιτική για τις οικογένειες. Αν δούμε το πρόγραμμά σας ε, για τις οικογένειες είναι ένα παλαιομοδίτικο πρόγραμμα για την, τις οικογένειες. Μια σύγχρονη πολιτική για τις οικογένειες σημαίνει οι άνδρες και οι γυναίκες ε, να είναι εξίσου αρμόδιοι για την ε, ανατροφή των παιδιών και να έχουν το ίδιο βάρος σε αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ ερχόμενη από τη Βουλγαρία καλωσορίζω την ε, τσεχική προεδρία και τη συγχαίρω που έχει βάλει στις προτεραιότητες της την ενέργεια. Τις τελευταίες μέρες πολλά ευρωπαϊκά κράτη-μέλη έπεσαν όμοιροι της ε, διαμάχης μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Μόνο στη Βουλγαρία πάνω από 160.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς θέρμανση. Δυστυχώς η βουλγαρική κυβέρνηση δεν μπόρεσε να βοηθήσει τους πολίτες της κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης. Ήταν η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν, είχε, που δεν έχει εναλλακτικέ ε, παροχές ε, φυσικού αερίου ε, νομίζω θα πρέπει από αυτό να βγάλουμε ένα συμπέρασμα. Νομίζω πως μιλάμε, μιλάω εξ ονόματος του Κοινοβουλίου ολόκληρο όταν μιλώ ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε οι πολίτες της Ευρώπης να πληρώνουν ε, τα σπασμένα των πολιτικών παιχνιδιών. Χρειάζεται μια κοινή ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη και σημαντικό στοιχείο αυτής της πολιτικής είναι η βελτίωση των υποδομών ενέργειας. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την ενέργεια σημαίνει κοινά ενεργειακά προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφυγή τη σημερινή πρακτική διμερών συμφωνιών. Επίση θα ήθελα να πιστεύω ότι σύντομα θα είναι δυνατόν να οικοδομηθούν νέοι, να κατασκευαστούν νέοι πυρηνικοί σταθμοί, κοινή ευρωπαϊκή πυρηνική σταθμή ω κοινά ε, προγράμματα των κρατών μελών. Και σε αυτό το πλαίσιο καλωσορίζω την Τσεχική Προεδρία που εντόπισε ως προτεραιότητα την ευρύτερη συνεργασία με τις ε, χώρες της, ε, του Καυκάσου και των Ανατολικών Βαλκανίων. Να μπορούμε να εγγυηθούμε την υπέρβαση κρίσεων όπως αυτή του φυσικού αερίου. Θα πρέπει να φτιάξουμε μια κοινή ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική και εύχομαι κάθε επιτυχία στην Τσεχική Προεδρία. Ευχαριστώ. Λεπτό παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρώπη χωρίς σύνορα, χωρίς φραγμούς είπατε είναι το σύνθημά σας. Ένα σημείο κέντρου βάρους είναι η ενεργειακή πολιτική για σας και η οικονομική σταθερότητα. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω επιπλέον ότι υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Για παράδειγμα, οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα έλεγα περισσότερα να γίνουν, μεγαλύτερη προσοχή να στρέψουμε στα καθημερινά προβλήματα των πολιτών μας, γυναικών και ανδρών θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές και την εφαρμογή του. Σημαντικό είναι το θέμα της ισότητας των ευκαιριών, η αλληλεγγύη. Πρέπει να διασφαλίζουμε και την προστασία των μειονοτήτων επιπλέον. Και συμφωνώ όσον αφορά με τη συνθήκη της πρέπει να επικυρωθεί αυτή η συνθήκη. Νομίζω τα κοινωνικά προγράμματα, τα κοινωνικά πακέτα, οι δέσμες μέτρων και η έλλειψη αυτών των προγραμμάτων ή των δεσμών μέτρων οδηγούν στο να μην έχουν εμπιστοσύνη πλέον οι πολίτες μας απέναντί μας. Και όσον αφορά την παιδεία και εκπαίδευση πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. předsedo η αρχή της τσεχικής ε, προεδρίας ε, σηματοδοτήθηκε από την κρίση στη Γάζα και την ενεργειακή κρίση. Και ακούστηκαν ε, διάφορες αντικρώμενες απόψεις. Η τσεχική κυβέρνηση θα προεδρεύσει της Ένωσης και τώρα η Ένωση παρακολουθεί με πολύ προσοχή αυτέ τι απροσδόκητε κρίσεις. Αναρωτιέμαι Όμω αν ήταν πραγματικά απροσδόκητε ή αν έπρεπε ήδη να τι είχαμε προβλέψει. Η γαλλική προεδρία δεν μπόρεσε να τι προβλέψει ε, στην αρχή. Θα ήταν καλό να αρχίσετε να διαπραγματεύεστε και με την Κίνα που συνεχίζει να ε, υποστηρίζει τον αθέμητο ανταγωνισμό βλάπτοντας και την υγεία των Ευρωπαίων καταναλωτών με ελαττωματικά προϊόντα. Α πούμε τώρα οι Ευρωπαίοι γονεί έχουν δυσκολία να αγοράσουν ε, παπούτσια για τα παιδιά τους που να μην είναι βλαβερά. Γι' αυτό και θα πρέπει να μιλήσουμε για την Ευρώπη στον κόσμο. Η Ευρώπη είναι πολύ ανοιχτή όσον αφορά τις διεθνείς συναλλαγές, ωστόσο Καμία Προεδρία του Συμβουλίου δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής να εγγυηθεί την αμοιβαιότητα με πλήρες άνοιγμα της ε, κινέζικης αγορά και για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Είμαι πεπισμένη ότι θα είσαι ε, επιτυχία. Συγχαρητήρια για την ε, παρουσίαση ενός πραγματικά συγκεκριμένου προγράμματος για την Ευρώπη και για τη δική σας προσωπική εξέλιξη που προέρχεται από ένα πολιτικό κόμμα το οποίο οι υπουργοί το 2003 καταψήφισαν την είσοδο στην Ένωση. Παρ' όλα αυτά, εσείς έχετε εξαιρετικό, εξαιρετική εικόνα στην Ευρώπη. Ελπίζουμε λοιπόν πως θα εξελιχθούν έτσι και οι δικοί σας συνάδελφοι ε, σε σχέση με την συνθήκη της Λισαβόνας. Οι Ιρλανδοί αρχίζουν να καταλαβαίνουν πως πρόκειται για μια, ένα μέσο το οποίο σωστά έχει συγγραφεί και θα βοηθήσει σε στιγμές κρίσης. Ελπίζω πως και εσείς θα υιοθετήσετε αυτή τη θέση, αν και ίσως ο Πρόεδρος Κλάους θα σβήσει το δικό σας αριθμό από το κινητό του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, πέρα των ζητημάτων της εξωτερικής πολιτικής, της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης και της επικύρωσης της συνθήκης της Λισαβόνας, μία από τις βασικότερες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι η νεολαία. Διάβασα την προτεραιότητα στο πρόγραμμά σας. Πιστεύω ότι το πρόγραμμά σας θα πρέπει να είναι πιο ολοκληρωμένο και πιο διαδραστικό στα ζητήματα της νεολαίας οι νέοι δεν πείθονται πλέον με διακηρύξεις και υποσχέσεις δεν αισθάνονται ασφάλεια έναντι ενός κράτους που καταραίει ανήμπορο να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση δεν αποδέχονται τα εκπαιδευτικά συστήματα που τους βάζουν στην αγορά της ανεργίας και της κοινωνικής απαξίωσης δεν αποδέχονται τον ευρωσκεπτικισμό τη φοβία απέναντι στην ευρώπη δεν ε, έχουν πρόβλημα με την επικύρωση της συνθήκης της λισαβόνας συγκρούονται σε καθημερινή βάση. η νέα γενιά είναι αυτή που μπορεί να κατανοήσει τι σημαίνει και να Λυπάμαι κυρία Μπαζελή, σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπόουις για δύο λεπτά. Χωρίς μικρόφωνο. Κύριε Πρωθυπουργέ, για μένα η Τσεχία είναι ο Γιάν Πάλατ και ο Φράντ Κάφκα και οι δύο συμβολίζουν τον αγώνα για τη δημοκρατία και την ελευθερία και επίσης δείχνουν πόσο έχει υποφέρει η χώρα για τους αγώνες αυτούς. Γι' αυτό νομίζω ότι και εσείς πρέπει να καταλάβετε τι πόνο υποφέρουν οι άνθρωποι στη Γάζα και ελπίζω και εσείς να κάνετε ό,τι μπορείτε για να σταματήσει η σφαγή εκεί. Επίσης, μπορείτε να δηλώσετε στον Αμερικανό Πρόεδρο ορισμένα πράγματα για τις κλιματολογικές αλλαγές. Στην Τσεχία μπορείτε να τελειώσετε τις ε, νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν αρχίσει να αναλαμβάνονται εκεί. Ξέρω ότι το έχετε στο πρόγραμμά σας αναφέρατε την ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ιατρική γνώση και ιδίως για την ψυχιατρική. Είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στη δημιουργία της ιστοσελίδας για τις μεταρρυθμίσεις στην Τσεχία για τα ψυχιατρία και ελπίζω τέτοιες μεταρρυθμίσεις να εφαρμοστούν πράγματι όχι μόνο στην Τσεχία αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τον 2 Ιούνιο όταν θα περάσει η δέσμη για τα ψυχιατρία στην Ευρώπη. Ελπίζω να φροντίσετε και τότε να το έχετε στο πρόγραμμα της διάσκεψης γιατί πρόκειται για ιδιαίτερα ευπαθή και ευαίσθητα άτομα στην κοινωνία μας και ελπίζω να κάνετε ό,τι μπορείτε και γι' αυτό. Νιώργια, ένα λεπτό παρακαλώ. Θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ένα γεγονός πριν από 21 χρόνια στην συνάντηση των αντιπολιτευομένων ε, δυνάμεων στο Κάκενόσε μεταξύ Πολωνίας και Τσεχοσλοβακίας τότε. Η Τσεχική Δημοκρατία είναι η πρώτη από τις ανατολικές χώρες που αναλαμβάνει προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα και αυτό οδηγεί και σε υποχρεώσεις από πλευράς της. Η Τσεχική Δημοκρατία έχουσα την Προεδρία αναλαμβάνει το κληροδότημα όλων των αγώνων στην Ανατολική Ευρώπη να υπάρξει ένα πρότυπο δημοκρατικής κοινωνίας στην καταπολέμηση του σίδηρου παραπετάσματος. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία η Τσεχική Προεδρία. Υπάρχουν αρκετές προτεραιότητες που αντιμετωπίζεται. Πρώτη, η, η κύρωση της συνθήκης Λισαβόνας και η ενδυνάμωση τη εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει τεράστια σημασία να προετοιμάστε στρατηγικέ για τι διατλαντικέ σχέσει λαμβάνοντας υπόψη τη νέα εκλογή του νέου Προέδρου στη ΣΥΠΑ. Θέλω να ευχηθώ στον Πρόεδρο Βάσλαβ Χάβελ ταχύ ανάρρωση. Θέλω να αναφερθώ στην ετοιμότητα για την παρέμβαση όταν το θέμα των διαπραγματεύσεων με την Κροατία οδηγήθηκαν σε πάγωμα. Να υπενθυμίσω ότι κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να υποβάλει αυθεντικά έγγραφα και θα πρέπει πάντα να υπενθυμίζεται αυτή η ευθύνη που έχουν. Η Κροατία ουσιαστικά συμπεριέλαβε στοιχεία στους φακέλους. Δεν είπε όμως ότι τα σύνορα ετίθενται υπό αμφισβήτηση και κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν αυτό να θεωρηθεί αυθεντικό αξιόπιστο έγγραφο από πλευρά της ε, Κροατία. Είναι διμερή ε, αμφισβήτηση συνόρων μεταξύ μιας και άλλη χώρα. Ε, Κροατίας και άλλης. Πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα πρώτα και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να υπογραμμίσω. Δεν είναι το κέφι ή οποιαδήποτε ε, προτίμηση της ε, Σλοβενίας. Εδώ πρέπει να υπενθυμηθεί η ανάγκη αυθεντικών εγγράφων που πρέπει να υποβάλλονται που θα ευθυγραμμίζονται με τις απαιτήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια είναι μια πιθανή λύση. Πολλές προτάσεις υπάρχουν και πιστεύω και ευελπιστώ ότι η Τσεχική Προεδρία θα εξετάσει με τον δέοντα τρόπο την επαρκή απάντηση που πρέπει να δοθεί. Ίσως η μία απάντηση είναι να υποβάλει η Κροατία εν ολοκληρώσει τα ε, τις θέσεις της ε, αναφερόμενη σε σχέση με τα σύνορα αυτά αν είναι προσωρινά ή όχι λαμβάνοντας υπόψη μια τέτοια τοποθέτηση θα μπορούσαμε βήμα προς βήμα νομίζω να σημειώσουμε κάποια πρόοδο και να δώσουμε τη δυνατότητα στην Κροατία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δυνατόν γοργότερα και αυτό θα ήταν προς ε, όφελος και της Σλοβενίας Σας εύχομαι κάθε επιτυχία λοιπόν ε, στο έργο αυτών των διαπραγματεύσεων Λεπτό το λόγο snesla se na hlavu předsedy rady kritika já se umyslím. Ακούσαμε επικρίσεις για την Προεδρία και εγώ συμφωνώ. Όμως, στις ε, ε, τσεχικές τέργες υπάρχει πάντοτε ένα σοφός που δεν ε, φαίνεται και που ενεργεί σιωπηρά. Στο κάστρο της Πράγας είμαι βέβαιος ότι υπάρχει κάποιος τέτοιος άνθρωπος και είμαι βέβαιος και ότι η τσεχική προεδρία θα μπορέσει να εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις και θα επιτρέψει την οικονομική ανάπτυξη και σας εύχομαι κάθε επιτυχία ώστε να ισχύσουν τα όσα λένε οι Ισπανοί και οι Εγγλέζοι, αλλά και εγώ, ότι δηλαδή η σοφία φέρνει καλά αποτελέσματα. Κύριε, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το ότι η τσεχική δημοκρατία από την αρχή ήδη της Προεδρίας της διέλυσε τις αμφιβολίες για την ικανότητα που υπήρχαν ως προς την ικανότητα μιας νέας χώρας μέλους να αναλάβει προεδρία. Οι δύο κύριες κρίσεις, δηλαδή η Γάζα και η διακοπή της παροχής του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, είναι οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει. Η Τσεχία με τη Βουλγαρία είναι οι χώρες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ως προς το φυσικό αέριο και ο κύριος πολλάνε και ελπίζουμε να κάνει τις διαπραγματεύσεις που απαιτούνται με τη Ρωσία. Η Σλοβακία δεν έχει δικό της αέριο, γι' αυτό χρειάζεται τη βοήθειά σας. Η Ευρώπη χρειάζεται κοινή ενεργειακή πολιτική για να ενισχύσει τη διαπραγματευτική της θέση στα ενεργειακά. Άλλο πρόβλημα είχε αρχίσει με τη διαμάχη μεταξύ Γεωργίας και Ρωσίας και τώρα υπάρχει διαμάχη Ρωσίας-Ουκρανίας. Καιρό είναι πια να πάρουμε μαθήματα από τα γεγονότα αυτά. Πρέπει να δούμε σε ποιους τομείς εξαρτάται η Ένωση από τη Ρωσία και σε ποιους η Ρωσία εξαρτάται από την Ένωση. Οι σχέσεις με τη Ρωσία είναι σημαντικές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να καταχράτε τη δεσπόζουσα της θέση η Ρωσία για το φυσικό αέριο. Πρέπει να διαφοροποιήσουμε τις πηγές μας. Παραδείγματο χάρη την, ε, τον αεριαγωγό Ναμπουχοδονόσορο. Η Σλοβακία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και ελπίζουμε η στρατηγική απόφαση που θα ληφθεί και για τους πυρηνικούς σταθμούς εκεί να ληφθεί σοβαρά υπόψη από εσά. Υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες ακόμη, σοβαρές φραγμοί ακόμη για την εφαρμογή της ελεύθερης διακίνησης των προσώπων και πρέπει οι φραγμοί αυτοί να αφαιρεθούν. Θα ήθελα η Τσεχική Προεδρία να κάνει πράγματι αυτά που δήλωσε ότι θα κάνει. Το λόγο για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, σας εύχομαι ως συμπατριώτη σας, κύριε Τοπολάνεκ, καλή τύχη για την ε, Τσεχική Προεδρία. Πιστεύω ότι εκτός από τα οικονομικά δεν θα ξεχάσετε και τα κοινωνικά θέματα. Στην ε, τελετή της ένταξης της Σλοβακίας είχε ζητηθεί στενότερη συνεργασία από όλες τις χώρες. Θα ήθελα όμως να κάνετε μια ιδιαίτερη προσπάθεια για την ε, έγκριση την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας γιατί αν θέλουμε η Ένωση να παίξει σοβαρό ρόλο διεθνή πρέπει να εγκριθεί η συνθήκη αυτή. Άλλη σημαντική στιγμή της Προεδρίας σας θα είναι η συμμετοχή τα επόμενα πέντε χρόνια στην επίλυση των ενεργειακών. Έχουν ζητήσει αρκετοί συνάδελφοι το λόγο. Δεν θα μπορέσουν να τον πάρουν όλοι γιατί έχει περάσει ο χρόνος. Πέντε συνάδελφοι, όχι περισσότερο από ένα λεπτό ο καθένας σας παρακαλώ. Ο κύριος Κέλαμ πρώτος έχει το λόγο. Κύριε Κέλαμ, you have the floor. Prime Minister, I'd like to extend the... Πρόεδρε, θέλω να Κύριε Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ε, απευθύνω όλοι μου τις θερμότερες ευχές και την υποστήριξη. Ε, για την επιτυχή Προεδρία. Η αντιμετώπιση της ε, κρίσης, ε, της ενεργειακής κρίσης σημαίνει την πρόθεση των τεσσάρων ελευθεριών. Υποστηρίζω την δική σας διευθέτηση. Είναι πολύ σημαντικό χώρες όπως η Ουκρανία και η Ρωσία να υποκούσουν στον στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατική εμείς θεωρούμε πως εσείς θα ηγηθείτε για να πείσετε όλες τις 27 κυβερνήσεις να αρχίσουν ε, από τον επόμενο Αύγουστο την ε, σηματοδότηση ε, της ημέρας για επίσης να αναγνωριστούν τα εγκλήματα που έγιναν υπό τον κομμουνιστικό πολιταρχισμό. Έχει το λόγο μόνο για ένα λεπτό doamnă președintă domnule comisar domnule Πριν ministru economie energie și uniunea europeană în lume este motoul președinției. κυρία πρόεδρε κύριε πρωθυπουργέ οι ευρωπαίοι πολίτες αναμένουν από την ένωση και από τους θεσμούς της να τους προστατέψει κατά των επιπτώσεων της κρίσης και να βελτιώσει το βιωτικό τους επίπεδο. Το σχέδιο αναθέρμανσης με μεγαλύτερη ενεργειακή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των προμηθειών είναι ουσιώδη και ζωτικά για τους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από την τεχική Προεδρία στις επόμενες ευρωεκλογές να φανεί ότι υπάρχει όραμα να μπορούμε και εμείς να πούμε στους πολίτες μας ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό όραμα για τη μεγαλύτερη παραδείγματο χάρη ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Επίση θα ήθελα και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να σας υποστηρίξουν για, ως προς τις προτεραιότητές σας. Για να υπάρξει προτεραιότητα ιδίως για αυτή την οδηγία για την ενέργεια. Ευχαριστούμε κυρία Τικάου. Το λόγο για ένα λεπτό. Πρωθυπουργέ, μετά από την δραματική εμπειρία του ρωσικού κομμουνισμού στο παρελθόν, η χώρα σα τώρα έχει περάσει στο άλλο άκρο και έχει προσκοληθεί σταθερά και με ε, δουλικότητα στη ΣΥΠΑ. Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο από τι τάσει για την υπόθεση τη Γάζας και τη συνθήκη τη Λισαβόνα, αλλά και επειδή θέλετε την εγκατάσταση των Αμερικανικών πυράβλων στο τσεχικό έδαφο διακινδυνεύεται την ειρήνη στην Ευρώπη με αυτή σα τη στάση και αυτό είναι απαράδεκτο και ύποπτο. Η χώρα σα είναι μέλο τη Ένωση, κύριε Πρωθυπουργέ, όχι τον ΙΠΑ. και θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η κυβέρνησή σα θα ενεργεί αντιστοίχω. Τα, αμερικανικά δορυφο... κράτη, τα κράτη δορυφόρη τη Αμερική δεν έχουν θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αποφασίσετε. Ευρωπαϊκή Ένωση ή ΗΠΑ. Δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δύο. Ευχαριστώ. Ησυχία παρακαλώ. Τώρα το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Πιοτρόφσκι, παρακαλώ. Ο κύριος... Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Η Τσεχική Προεδρία είναι η πρώτη μετά από ολόκληρη σειρά ετών που δεν συμπεριλαμβάνει το Σύνταγμα που τώρα αποκαλείται Συνθήκη Λισαβόνα ω μία από τι προτεραιότητε. Είμαι ευελπιστό για την Προεδρία σα, γιατί αυτό σημαίνει θα σέβεστε τη δημοκρατία και την αρχή τη ομοφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τσεχική Προεδρία επικεντρώθηκε στα σημαντικά ουσιοθέστερα θέματα, όπω την ασφάλεια του ανεφοδιασμού με ενεργειακά προϊόντα τη Ευρώπη. Όμω, από την άλλη πλευρά, ίσω έχει ήδη κάνει και καλή δουλειά όσον αφορά την αντιπαράθεση μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών για το φυσικό αέριο. Φυσικά σε έξι μήνε δεν θα επιτύχετε όλους τους στόχου σας. Όμως οι πρώτες δύο εβδομάδες ήδη κατέδειξαν ότι μπορεί να είσαστε αποτελεσματικοί. παρόλε τι ε, ακραία αρνητικές ε, προτάσεις ε, κάποιων μελών στο σώμα. Βάνοφ, ένα λεπτό παρακαλώ κύριε Στοβάνοφ. Ησυχία κύριε και κύριοι συνάδελφοι. Κύριε Στοβάνοφ. Стоянов. Παρακαλώ, ο κύριος Στογιανόφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα ότι υπό την Τσεχική Προεδρία υπάρχει η εικόνα της Βουλγαρίας ως τουρκικού αποχωρητηρίου. οι ευρωπαϊκές αξίες απαιτούν αμέσως να, να χορηγηθεί αίτηση συγγνώμης. Να το αποσύρουν αυτό. Και εγώ και οι συνάδελφοί μου θα διαμαρτυρηθούμε έντονα. Ο, ε, ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Στοπάλαν, ε, ε, εξ του Συμβουλίου, έχει το λόγο. Ja Κυρία Πρόεδρε, στον καταληκτικό μου αυτόν λόγο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα είπατε σήμερα εδώ. Για μένα ήταν πολύ ενθαρρυντικά, περισσότερο από όσο ανέμενα. Η Προεδρία μας και εγώ προσωπικά το Συμβούλιο θα τηρούμε στενή επαφή και συνεργασία και με την Επιτροπή και με το Κοινοβούλιο. Οι πρώτες ήδη εβδομάδες έδειξαν ότι η καθημερινή συνεργασία και με τον κύριο Μπαρόσο και με το σύνολο των Επιτρόπων είναι κάτι που μπορεί να διασφαλίσει με την κοινή προσπάθεια μια κοινή διαδικασία με την οποία να προχωρήσουμε όλοι στον ίδιο δρόμο και με πολύ απτή πρόοδο. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τη συνεργασία. Πριν να έρθω είχα υποσχεθεί ότι δεν θα αστιευτώ Προσπάθησα παρόλα αυτά να σας πω και κάτι αστείο φαίνεται δεν έγινε αντιληπτό. είχα πει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας πρέπει να θεωρηθεί σαν μέσον και όχι σαν σκοπός. Είναι μέσον με το οποίο να υπάρξει καλύτερη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό σκοπός. Αλλά κάθε χώρα μέλος βέβαια έχει τα δικά της εργαλεία για την επικύρωσή της. Εγώ δεν είπα, δεν είπα ότι μπορώ να επηρεάσω τα πράγματα και στην Άνω και στην Κάτω Βουλή της Τσεχίας είναι ανεξάρτητα όργανα. Ούτε μπορώ να επηρεάσω την απόφαση του Ιρλανδικού λαού γιατί η συνθήκη δεν πρέπει να εφαρμοστεί με το ζόρι. Πιστεύω όμως ότι χρειάζεται κάποια αναμονή να περιμένουμε την απόφαση του Ιρλανδικού λαού και αναμένω η έγκριση της συνθήκη να διευκολύνει τη λειτουργία της Ένωσης. Δεν χρειάζεται νομίζω να πω τίποτε παραπάνω. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω όμως μια άλλη παραπομπή στον Τσόρτσιλ ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι όπως είχε πει εκείνος ότι δεν θα υπάρξει άλλη κρίση γιατί είναι το πρόγραμμά μου ήδη γεμάτο από τέτοιες. Οι πρώτες δύο εβδομάδες της Τσεχικής Προεδρίας δείχνουν ότι αν θέσουμε σωστά τις προτεραιότητές μας μπορούμε όμως να τις αντιμετωπίσουμε ακόμη και αν υπάρξουν και άλλες κρίσεις. Ήδη από τα τέλη της Γαλλικής Προεδρίας είχαμε αρχίσει την προετοιμασία μας Ζητώ συγγνώμη αν δεν απαντήσω σε όλους προσωπικά, αλλά γενικά θα έλεγα ότι το πρόβλημα της δουλεμπορίας ιδίως παιδιών δεν είναι κάτι που το αγνοώ. Το κοινοβούλιο σας το συζητάει εδώ και αρκετό καιρό καθώς και το γενικότερο πρόβλημα εξισορρόπησης της ελευθερίας με την ασφάλεια. Παρόμοια συζήτηση γίνεται και στη χώρα μου και με αυτό εννοώ ότι το νομοθετικό πρόγραμμα προβλέπει μια απόφαση του Συμβουλίου για τη δουλεμπορία, για την εμπορία ανθρωπίνων όντων και άρα δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αγνοήσουμε. Επίσης έγινε συζήτηση για τον αεριαγωγό Ναμπούκο ο οποίος μπορεί να συμπληρώσει τους υπάρχοντες με χρήσιμο τρόπο. Τώρα για την κρίση στην Ουκρανία. Ένας τσέχος συνάδελφος είπε ε, ασαφώς τι συνέβαινε. Είναι γεωπολιτικό πρόβλημα και αν δεν δώσουμε την ευκαιρία στην Ουκρανία να λύσει το εσωτερικό της πρόβλημα αν δεν επηρεάσουμε τη συμπεριφορά όλων των παραγόντων στην αγορά του αερίου, τότε μπορούμε να χάσουμε την Ουκρανία. Α, είναι σοβαρό γεωπολιτικό πρόβλημα, δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα γίνει, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε τι μπορεί να δημιουργήσει η κρίση αυτή ως προς τις τιμές ή τι πίεση θα ασκηθεί για την δημιουργία του North Stream ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να εμποδίσει την Ουκρανία στην πρόοδό της. Το πρόβλημα πάντως πρέπει να το δούμε μέσα στο γενικότερο μακροπρόθεσμο πλαίσιο και να μην επιζητήσουμε μία βραχυπρόθεσμη μόνο λύση. Τώρα το κατά πόσον πρέπει η Ευρώπη να έχει περισσότερο φιλελεύθερο ή περισσότερο σοσιαλιστικό χαρακτήρα, ας κάνω ένα αστιάκι επιτρέψτε μου έναν συμβιβασμό δηλαδή, να είναι μια φιλελευθεροσυντηρητική Ευρώπη. Αυτό θέλω εγώ. Άλλο αστείο δεν θα σας πω, σας το υπόσχομαι. Οι ευρωπαϊκές οικονομίες όταν θα είναι όλες στην Ευρωζώνη, γιατί από την 1η Νοεμβρίου φέτος η Τσεχική Δημοκρατία θα ανακοινώσει πότε μπορεί να μπει στο ευρώ και θα μπουν στο ευρώ και άλλες χώρες και η ίδια εφόσον έχει πληρώσει τα περισσότερα κριτήρια του Μάστριχτ θα ακολουθήσει η Σλοβακία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα ως προς το σύμφωνο σταθερότητας και την πλήρωση των υπολείπων κριτηρίων. Φοβάμαι ότι αν αποδυναμώσουμε τους κανόνες αν βάλουμε νερό στο κρασί μας θα, καταστρέψουμε όλα. Πρέπει να εφαρμόζουμε τους κανόνες που έχουμε εγκρίνει. Και μόνο έτσι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα μας. Γι' αυτό επιμένουμε και για την εφαρμογή των οδηγιών ως προς τις δημόσιες επιχορηγήσεις και τον ανταγωνισμό. Βέβαια οι κανόνες πρέπει να γίνονται σεβαστοί και τους καλούς και τους κακούς καιρούς και πρέπει να τους σεβόμαστε απόλυτα. Όσο για την Ευρώπη χωρίς σύνορα ή χωρίς φραγμούς, εδώ υπάρχουν τρεις έννοιες που μπορεί να έχει οικονομικά, Αυτό θα σήμαινε την κατάργηση των φραγμών στην εσωτερική αγορά. Υπάρχει όμως και μία πιο διανοητική, πιο πνευματική έννοια, δηλαδή στα μυαλά να καταργηθούν οι φραγμοί στα μυαλά των πολιτών, των Ευρωπαίων. Και έπειτα υπάρχει και η έννοια της απελευθέρωσης γενικότερα της ευρωπαϊκής οικονομίας μέσω της οποίας μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης και να σεβαστούμε τα συμπεράσματα της Ουάσιγκτον και κάτι άλλο ακόμη που προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ. Δυστυχώς ο Βάτσλαβ Χάβελ λέει ο μιλητής είναι στο νοσοκομείο πολύ σοβαρά άρρωστος έχει γίνει, έχει γίνει το σύμβολο της αλλαγής και και τις ε, πτώσεις του σιδηρού παραπετάσματος στη χώρα μας. Είναι ο πρώτος που μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εξ ονόματος όλων μας του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση. Και τώρα δύο λόγια για να απαντήσω συγκεκριμένα σε όσα είπαν ορισμένοι ευρωβουλευτέ. Την ανησυχία του κυρίου Τσέκ την βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσα και, και συγκινητική. Τα τελευταία 15 χρόνια τουλάχιστον 6 ε. τουλάχιστον έξι προηγούμενα υπάρχουν για επιτυχής προεδρίες με ανάλογα προβλήματα. Παραδείγματος χάρη. Ο ανασχηματισμός στο Βέλγιο, η επικύρωση της συνθήκης του Αμστελοδάμου, η γερμανική προεδρία τότε υπό τον Σρέντερ αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα και όταν εγκρίθηκε και το ευρώ επίσης, κατά την Ισπανική Προεδρία Υπό τον Αθνάρη υπήρχαν πολλά προβλήματα, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίστηκαν. Μην ανησυχείτε λοιπόν για τα εσωτερικά προβλήματα της Τσεχίας δεν θα επηρεάσουν την τσεχική προεδρία της Ευρωένωσης. Για την πυρηνική ενέργεια τώρα δεν μπορούμε να την αναλύσουμε μόνο από την άποψη των πρασίνων ή των συντηρητικών. Εμείς θέλουμε το πυρηνικό βήμα, το πυρηνικό σεμινάριο που θα οργανώσουμε στην Πρατισλάβα να αρχίσει μια καινούργια συζήτηση γενικότερα για τις δυνατότητες και τους κινδύνους που εμπεριέχει η πυρηνική ενέργεια. Θέλουμε να πάψει να υπάρχει το ταμπού εναντίον της που υπάρχει. στην Ουκρανία χάρη στην ε, στην Ουκρανία ως προς το πρόβλημα που έχει η Ουκρανία μάλλον έχει επιπτώσει στην Βουλγαρία και την Σλοβακία ιδιαίτερα η ροή του αερίου από τη Ρωσία μέσω της Ουκρανίας εκεί. Είναι πολύ δύσκολη η κατάστασή τους και εγώ έχω καθημερινές επαφές με τον πρόεδρο της Ουκρανίας. Ελπίζω να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα αυτό γιατί είναι διπλή η προσπάθεια που πρέπει να γίνει και με τον Κασπρόμ και με την Ουκρανία. Οι προσπάθειες αυτές πρέπει να είναι πολύ εντατικότερες βέβαια και η Τσεχική Προεδρία θα κάνει ό,τι μπορεί. Πρέπει όμως παράλληλα να βρεθούν νέες πηγές ίσως και νέες τεχνολογίες γιατί το αέριο το χρησιμοποιούμε καμιά φορά σαν δικαιολογία για να μην ερευνήσουμε νέες και εναλλακτικές ενεργειακές πηγές. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα, Σλοβενι... τα προβλήματα μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας στην προενταξιακή διαδικασία της τελευταίας είναι επίσης σημαντικά και είναι κάτι που έχει ήδη επιπτώσεις στις προενταξιακές συνομιλίες. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω διαπραγματεύσεις και με τους Προέδρους Κροατίας και Σλοβενίας για να κάνω έτσι την προσωπική μου συμβολή στην επίλυση των μεθοριακών προβλημάτων μεταξύ Σλοβενίας και Κροατίας. Θα ήθελα να πω περισσότερα, αλλά ας μην σας κουράσω. Για να μπορέσετε και να συνεχίσετε τη δουλειά σας απρόσκοπτα. Τέλος, εκτιμούμε δεόντως τη δυνατότητα που είχαμε να γίνουμε μέλος μιας διεθνούς κοινότητας όπως της Ευρωπαϊκής που στηρίζεται στις ίδιες αξίες με τις δικές μας. από τον Νοέμβριο του 89 εννοώ και μετά. Και είμαστε, είναι για μας ιδιαίτερη τιμή που προεδρεύουμε της Ένωσης αυτής. Το 89 δεν μπορούσαμε ούτε καν να το ονειρευτούμε. Είναι λοιπόν όντως μια μεγάλη τιμή και τιμούμε ιδιαίτερο τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ελεύθερες συζητήσεις γιατί τα προβλήματα μεν υπάρχουν αλλά η δυνατότητα μιας, ενός ελεύθερου διαλόγου μπορεί να τα ταυτίσει και να δοθεί η δυνατότητα της επίλυσης τους. Η δημοκρατία σημαίνει συζήτηση ακριβώς και αυτό ακριβώς θα εφαρμόσω και εγώ. Είμαι ανοιχτός για συζήτηση πάντοτε. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω να σας ξαναμιλήσω άλλη φορά. Ησυχία σας παρακαλώ για να ολοκληρώσουμε. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Μπαρόζο, έχετε λόγο. Thank you very much, Madam President. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, αξιότιμα μέλη ευρωβουλευτές. Ενθαρρύνομαι από τη συζήτηση και κοινή προσέγγιση ανάλυσης των προκλήσεων και γενικά με την υποστήριξη που έχει εκφραστεί υπέρ τη Τσεχική Προεδρίας. Και πάλι για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω την επιθυμία μου να συνεργαστούμε με το πιο επικοδομητικό πνεύμα με τους Τσέχους φίλους μας. Η δική του επιτυχία είναι επίσης η επιτυχία της Ευρώπης. Όπως κάποιοι από εσάς υπογράμμισαν, αυτή είναι η τελευταία προεδρία πριν από τις ευρωεκλογές του 2009. Νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των μενών θα πρέπει όλοι να δείξουμε ότι όλα τα θεσμικά μας όργανα καταβάλουν προσπάθειες για την ευημερία, την αλληλεγγύη των πολιτών μας συνολικά. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε σωστά, να περάσει αυτό το μήνυμα και να επικοινωνούμε. Και αυτό δεν μπορεί να γίνεται μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή από τα ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει από κοινού να συνεργαζόμαστε υπό αυθεντικό πνεύμα αλληλεγγύης. Πολλά από αυτά που θα γίνουν αυτούς τους έξι μήνες θα είναι πολύ σημαντικά λοιπόν για το μέλλον της Ευρώπης. Και επίσης για τον σεβασμό των θεσμικών οργάνων μας πανευρωπαϊκά. Θα ήθελα να δραχθώ τη ευκαιρία να απαντήσω κάποιε συγκεκριμένες ερωτήσεις που μου διατυπώθηκαν, ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα της ενέργειας. Μάλιστα, ναι, χρειαζόμαστε ταχύτατα αναθεώρηση της οδηγίας για ανεφοδιασμό με φυσικό αέριο. Ήδη το είπε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παρουσιάσαμε την ευρωπαϊκή πολιτική μας στρατηγικής αναθεώρησης για αυτό το θέμα και εργαζόμαστε για να υπάρξει η ε, νομοθετική πρόταση ενώπιον της Ευρωβουλής και του Συμβουλίου των δυνατών ταχύτερα. Ναι, μάλιστα, χρειαζόμαστε περισσότερη, μεγαλύτερη αλληλεγγύη, μεγαλύτερη πρόοδο που θα επιτευχθεί όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Αυτό ήταν το περιεχόμενο της στρατηγικής μας αναθεώρησης όσον αφορά αυτά τα θέματα και της υποβολής ε, αντίστοιχης πρότασης από πλευρά μας. Και θέλω να δραχτώ αυτή τη ευκαιρία για άλλη μια φορά να ζητήσω από όλα τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεργαστούν με πιο ενεργό τρόπο στους μηχανισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Αλληλεγγύης. Ναι, μάλιστα, πρέπει επίσης να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις υποδομές για την ενέργεια, στη διασύνδεση και στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Γι' αυτό για όλους αυτούς τους λόγους είναι τόσο σημαντικό τα 5 δις ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό να διατεθούν για αυτούς τους στόχους. Απευθύνω έκκληση σε εσάς, στην Ευρωπαϊκή, την Ευρωβουλή και την Τσεχική Προεδρία να μεταφραστούν σε πράξεις όλοι αυτοί οι στόχοι το δυνατόν γοργότερα. Ναι, μάλιστα η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συνοδεύεται με την ευφυή πράσινη αναπτυξιακή πολιτική αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στι προκλήσει. Οι προτάσει μα ευρίσκονται επί τραπέζης. Να επιταχυνθεί η χρήση των ε, διαθωτικών ταμείων υπέρ αυτών των στόχων Κονδύλια χρειάζονται λοιπόν για την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ενεργειακή αλληλοδιασύνδεση και μέσω συντονισμού των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινήτρων θα προσανατολίσουμε τις εθνικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση ευθυγραμμιζόμενη με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου πάντα. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω και κάτι άλλο. Να πω δηλαδή ότι να η αντιμετώπιση αυτής της οικονομικής κρίσης και η επαναφορά της Ευρώπης σε αηφόρο ανάπτυξη θα απαιτήσει επίσης και τον σεβασμό των ευρωπαϊκών κανόνων του παιχνιδιού για τις ίσες ευκαιρίες. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει διευκολύνοντας την συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην οικονομική δραστηριότητα και βοηθώντας να συνδυαστεί η οικονομική ζωή με την επαγγελματική ζωή αυτών των ατόμων. Δύο λόγια για συνθήκη της Λισαβόνας επίσης που πολλοί από ε, προανέφεραν τη χρειαζόμαστε αυτή τη συνθήκη περισσότερο από ποτέ που θα έχει επικυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Ναι, μάλιστα, πρέπει να σεβόμαστε όλε τι διαδικασίε από πλευρά των κρατών μελών για την επικύρωση. Όταν όμω μια κυβέρνηση εξ ονόματο μια χώρα υπογραμμίζει, μια, υπογράφει μια τέτοια συνθήκη, αναλαμβάνει επίσημα την υποχρέωση υλοποίηση αυτής της συνθήκης Πολλοί από εσά έκαναν λόγο για την Σεχική Προεδρία και πόσο σημαντική είναι. Θα έλεγα, όπω και αρκετοί από εσά είπαν, ο κ. Νασάουερ, ο κ. Μπροκ και άλλοι, ότι το γεγονό ότι έχουμε την Σεχική Προεδρία είναι αφεαυτού ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονό. Είναι η πρώτη φορά ιστορικά, όπου μια πρώην χώρα κράτος μέλος του Συμφώνου της Βασοβίας αναλαμβάνει την υποχρέωση του να είναι προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Και είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό, το ότι τώρα, 20 χρόνια μετά την κατάρρευση του σιδηρού παραπετάσματος, έχουμε την τσεχική δημοκρατία επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο Πρωθυπουργός Τοπολάνεκο ίδιος, ο, όλοι οι συνεργάτες του να έχουν επομιστεί πλέον αυτές τις ευθύνες. Ευελπιστούμε και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο σας. Και επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε ένα βίωμα που είχα πέρυσι κατά την Πορτογαλική ε, Προεδρία με τον Πρωθυπουργό ε, Σόκρατες ήμουνα στα σύνορα μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας, Πολωνίας και Γερμανίας και είδα η δύσόμαση τη συγκίνηση του Πρωθυπουργού Τοπολάνεκα πώς ε, βίωνε εκείνη τη στιγμή σε εκείνα τα σύνορα που μας χώριζαν στην Ευρώπη μεταξύ των δύο πλευρών της ελεύθερης Ευρώπης και του σιδηρού παραπετάσματος. Τώρα είναι ένα, ένα ελεύθερο κομβικό σημείο για την ελεύθερη διακίνηση, κυκλοφορία των πολιτών ε, από αυτό. Πρέπει να είμαστε περήφανοι και να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προασπίζουμε τις αξίες μας για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η Προεδρία. Κάποιοι από εσά είπαν πιο πριν ότι είναι σημαντικό να στεφτεί με επιτυχία η Τσεχική Προεδρία, γιατί είναι λέει μικρή χώρα. Λυπάμαι όμως, δεν είναι μικρή χώρα η Τσεχική Δημοκρατία, πρέπει να διαφωνήσω. Και εδώ πράγματι, καμιά φορά βλέπουμε να υπάρχει ένα σύμπλεγμα κατωτερότητας, να θεωρούνται κάποια κράτη-μέλη, λέει, μικρές χώρες, μικρά κράτη. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ως ένας από τους ιδρυτές ε, είπε ο Πορανρή Σπάκ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπάρχουν πλέον εφ' μικρές και μεγάλες χώρες. Όλες τους θα είναι όχι μεγάλες, θα είναι ίσες μεταξύ τους. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχουν συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός κάποιες από αυτές τις χώρες. Πράγματι, βλέποντας τον υπόλοιπο κόσμο, όταν στρέφουμε το βλέμμα και βλέπουμε την αμερικανική δύναμη όσον υπερ, υπερδύναμη όσον αφορά τα θέματα άμυνα και τεχνολογία. Όταν δει κανεί αυτή τη διάσταση, όταν δει κανεί την τεράστια γεωγραφική έκταση ο συνιστόσα τη Ρωσία, όταν δει κανεί την πυκνότατη δημογραφία, δημογραφική ε, συνιστόσα τη Κίνα, να μιλάει κανεί για μεγάλε χώρε στην Ευρώπη, δεν υπάρχουν πια μεγάλε χώρε στην Ευρώπη. Όλε είναι μεγάλε όσον αφορά την αξιοπρέπεια, τον αυτοσεβασμό. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα κράτη-μέλη έχουν την ίδια αξιοπρέπεια και την χάνουν του ίδιου σεβασμού. Αν θέλουμε να είμαστε μεγάλοι στον κόσμο, πρέπει να δράσουμε ώστε να ενωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μιλάμε μια γλώσσα, να μιλάμε όλοι ενωμένοι ως Ευρωπαίοι. Και έτσι θα δημιουργήσουμε μια διαφορά στον κόσμο υπέρ ημών. Γι' αυτό χρειαζόμαστε τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Για ένα κοινό στόχο. Χρειαζόμαστε ισχυρά θεσμικά όργανα. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Τσεχική Προεδρία. Thank you, Mr. President. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κάτι περισσότερο από τον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά ήταν πολύ σημαντική και ενδιαφέρουσα.